Συνεχίζουμε λοιπόν την συνεδρία που διακόψαμε χθε το απόγευμα, σημείο 9 τη ημερήσια διάταξη. Έχουμε μια ανταλλαγή απόψε με τον κύριο Χώμα, τον Γενικό Διευθυντή τη ΒΑΝΤΑ, του Παγκοσμίου Οργανισμού για την Καταπλήρωση τη Φαρμακοδιέργεση. Η δική του πρωτοβουλία ήταν να έχουμε τη συνάντηση αυτή και ενδιαφερόμαστε πάρα πολύ να ακούσουμε τι έχετε να μα πείτε. Μια που ξέρουμε ότι εμεί ω Κοινοβούλιο δεν έχουμε και πολύ μεγάλη δυνατότητα, για να μην πω καμία δυνατότητα επίδραση στη ΒΑΝΤΑ. Αλλά οι εργασίε τη ΒΑΤΑ βέβαια μα ενδιαφέρουν. Γιατί όλοι θέλουμε να υπάρχει καθαρότης στον αθλητισμό. Λοιπόν, ενδιαφερόμαστε, λέω, για τον τρόπο εργασία αυτής της οργάνωσης. Θέλουμε να ξέρουμε από πού υπάρχουν επιτράσεις, θέλουμε να ξέρουμε ποιες είναι οι δυσκολίες που υπαρχουν επιτράσει, θελουμε να ξερουμε ποιε ειναι οι δυσκολιες που διαβλεπονται Και θα ήθελα να σα υπενθυμίσω ότι η ΒΑΝΤΑ καλύπτει και τα συμφέροντα της Ευρώπης που εκπροσωπείται από το Συμβούλιο της Ευρώπη. και μέσω της εκπροσώπησης του Συμβουλίου της ε, ε, Ευρώπης θέλω να τονίσω ότι αισθανόμαστε ότι εκπροσωπούμεθα πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, κύριε Χαόμαν, χαιρόμαστε που σας εδώ. Σας δίνουμε 20 λεπτά και ελπίζουμε να καταφέρετε να ολοκληρώσετε την ομιλία στα 27 λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί βουλευτές. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να έρθω εδώ και να σας μιλήσω. Είναι πραγματικά μεγάλη τιμή για μένα που μπορώ να κάνω αυτή την παρουσίαση ενώπιον ημών. Θα ήθελα καταρχήν να απαντήσω στην ερώτηση γιατί χρειάζεται να αγωνιστούμε για καθαρό αθλητισμό. όλα όσα κάνουμε στη Βάντα τονίζουμε τα δικαιώματα του καθαρού αθλητού. Και δεν θέλουμε να υπάρχουν αθλητές που καταποτούν τους κανόνες. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το μεγάλο ποσοστό των αθλητών στον κόσμο είναι καθαροί και είναι δικαίωμά τους να μπορούν να αθλούνται και να αγωνίζονται σωστά με κάθε σεβασμό προς το άθλημά τους. Και αυτό ακριβώς προσπαθούμε να κάνουμε. Υπάρχουν βέβαια προκλήσεις σε αυτό που κάνουμε. Και στρεφόμαστε τώρα στον ίδιο τον αθλητή, την ίδια την αθλήτρια. Και κοιτάζουμε τις ανθρώπινες επιδράσεις τις οποίες υφίσταται. Δάσκαλοι, προπονητές, γονείς, δικηγόροι, γιατροί, θεραπευτές, συναθλητές, Όλοι αυτοί έχουν κάποιο επίπεδο επίδρασης πάνω στον αθλητή. Και πολλές φορές αυτοί είναι εκείνοι οι οποίοι πείθουν τους απλοϊκούς αθώους αθλητές να απατήσουν για να αυξήσουν ευκαιρίες τους. Those και πολλές φορές είναι δύσκολο να βρούμε ποιος έχει συμμετάσχει στην ε, επίδραση αυτή στον αθλητή ακριβώς. Πολλές φορές υπάρχουν άτομα που δεν είναι τμήματα, που δεν είναι μέρη των αθλητικών οργανώσεων ή των ομίλων. Προσπαθούν, να εκμεταλλευτούν τι δυνατότητες που έχουν μέσα στα πλαίσια του ιατρικού επαγγελματό ή του δικηγορικού επαγγελματό για να έχουν κάποια επίδραση. Μετά προσθέτουμε τις κοινωνικέ επιδράσει στον αθλητή και βλέπουμε ότι δεν είναι μόνο θέμα αθλητικό. Είναι θέμα εγκλήματος. Είναι θέμα δημόσιας υγείας. Πολλοί μας λένε πόσο εύκολο είναι κάτι τέτοιο τώρα με το διαδίκτυο θα μπορούσαμε να πάω στο διαδίκτυο και να αγοράσω από κάπου υλικά με τα οποία μπορώ να παρασκευάσω στερεοειδή. Όταν ξεκινήσω έτσι μια, ένα εργαστήριο, ίσως με μικρό μικρό τίμημα μπορώ να κερδίσω 20.000 ευρώ. Και αυτό μπορεί να γίνει σε πολλές χώρες του κόσμου που δεν υπάρχουν κανόνες. Είναι λοιπόν μια νόμιμη δραστηριότητα εκεί και πολλοί επιχειρηματίες την εκμετάλλονται. Είναι αθλητές. Πολλές φορές είναι αθλητές. Πολλές φορές όμως αυτοί είναι μαθητές του σχολείου και αγοράζουν τα υλικά αυτά από εκείνους που τα κατασκευάζουν. Και τα αγοράζουν απλώς για να βελτιωθούν οι ίδιοι. Αυτό λοιπόν είναι ένα πρόβλημα που υπάρχει στην κοινωνία τη σημερινή. Υπάρχει ένα θέμα δημόσιας υγείας, όπως σας είπα, που εξετάζουμε. Θα ήθελα να θυμίσω, κύριε Πρόεδρε, τι είναι η ΒΑΝΤΑ. Εμείς δεν είμαστε μια υπηρεσία ελέγχου. Εμείς είμαστε διακανιστικό σώμα υπεύθυνο για την επιτήρηση του κώδικα που έχει γραφτεί και υιοθετηθεί από κάθε άθλημα, σε κάθε κράτος του κόσμου. We have an equal partnership between sport and governments είναι ένα σώμα που προσπαθεί να είναι σε εταιρική σχέση και με το άθλημα και με την κυβέρνηση. 50% στην εταιρική σχέση μεταξύ των, του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα. Και στα πλαίσια αυτής της εταιρική σχέσης προσπαθούμε να συνεργαστούμε και με τα δύο μέρη και με τις δύο πλευρές. Ξέρουμε ότι πολλά μπορούν να κάνουν οι κυβερνήσεις, από κοιμού Έχουμε λοιπόν ένα μέτωπο για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε αυτή τη μάστιγα του αθλήματος. Το μοντέλο διακυβέρνησης είναι μοναδικό, γιατί υπάρχει ευρεία συμμετοχή, 50% από το αθλητικό κίνημα, 50% από τις κυβερνήσεις του κόσμου. Τα κυβερνώντα σώματα ΣΒΑΤΑ είναι το Ιδρυτικό Συμβούλιο, 18 από κάθε πλευρά, 18 μέλη από κάθε πλευρά. Οι κυβερνήσει όλου του κόσμου έχουν ορίσει πώ θα καταμερίσουν μεταξύ του τις 18 αυτέ έδρε που δικαιούνται. Εκείνοι το κάνουν, Εμεί δεν κάνουμε. Αποφασίσανε πέντε έδρε για την Ευρώπη, τέσσερι για την Ασία, τέσσερα για την Αμερικανική Ήπειρο, τρει για την Αφρική και δύο για την Οκεανία. Ε, και υπάρχει και μια εκτελεστική επιτροπή που έχει πέντε μέλη κυβερνήσεων, ένα δηλαδή από κάθε ήπειρο του κόσμου. Μια σύντομη ιστορία της Βάντα. Βλέπετε ότι γεννηθήκαμε μετά την καταστροφή στο γύρο της Γαλλίας του 1998. Η διάσκεψη που συγκάλεσε ε, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή συνεδρίασε το 1999 και καθόρισε να συμβάλλει σημαντικά και μέσω των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων να υπάρχει μία ανεξάρτητη υπηρεσία διεθνής, η οποία είναι αυτή η ΒΑΝΤΑ. Πρώτη φορά στο Σίδνεϊ υπήρχε μία ανεξάρτητη ομάδα παρατηρητών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2000. Διευρύναμε μετά τις δυνατότητές μας και ιδρύσαμε μια εκπαιδευτική ομάδα, αν θέλετε, για να εκπαιδεύει τους αθλητές που συμμετάσχουν σε αυτούς τους ε, αγώνες. Καταρχήν στη Βιλανδία, στο Ευρωπαϊκό Φεστιβάλ ε, Ολυμπιακών Αγώνων Νεολαίας. Και υπάρχει δυνατότητα κάθε χώρα να προσαρμόσει τους ε, κώδικες και κανόνες στη ΒΑΔΑ στη δική της νοοτροπία στη δική της γλώσσα χωρίς χρήματα. Το 2002 από τη Λοζάνη μετακομίσαμε στο Μενρεάλ. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα μιας επιλογής. Εφτά πόλεις ε, θέλησαν να συμμετάσχουν, να, συγγνώμη, να υποδεχθούν το επιτελείο της ΒΑΝΤΑ και επελέχθη τελικά το Μονρεάλ. Και είμαστε σήμερα στο Μονρεάλ. υπό την ηγεσία της ε, καναδικής κυβέρνησης με ισχυρή οικονομική ενίσχυση και θα μείνουμε εκεί μέχρι το 2020 όταν ολοκληρωθεί η μελέτη τους. Μια δεύτερη διεθνή διάσκεψη το 2003 στην ε, Κοπενχάγη δέχτη τον διεθνή κανόνα αντι-doping ε, και τελικά ολοκληρώθηκε το 2004 στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Το 2005, υπό την ηγίδα του UNESCO, υπήρχε μια συνθήκη που εγγράφει και με την οποία οι κυβερνήσεις μπορούν να γνωρίσουν αυτόν τον κώδικα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι η συνθήκη αυτή γράφτηκε μέσα σε 12 μήνες. Παγκόσμιο ρεκόρ δηλαδή. Και επικυρώθηκε σε 12 μήνες. Πάλι ένα ρεκόρ παγκόσμιο για σύμβαση της UNESCO. Αποφασίσαμε το 2006 ο κώδικας που υιοθετήθηκε θα έπρεπε να αναθεωρηθεί. Θα έπρεπε να αναθεωρηθεί γιατί θα πρέπει να είναι άκαμπτοι οι κανόνες, θα, θα πρέπει να αλλάζουν ανάλογα με τις πρακτικές, με τις μεθόδους που έχουμε μάθει. Και ξεκινήσαμε έτσι σε μία μακρά περίοδο διαβούλευσης τρία προσέδια του κειμένου. Πάνω από 140 διαβουλεύσεις με ενδιαφερόμενα σώματα. Και τέλος το 2007 έχουμε την τρίτη παγκόσμια διάσκεψη στη Μαδρίτη, όπου ενεκρίθη ο αναθεωρημένος κώδικας. Το 2008 υπογράψαμε ένα σημαντικό έγγραφο με την Interpol, ένα ε, σύμφωνο συνεννόησης μαζί με τη φαρμακευτική βιομηχανία και το 2008 συγγνώμη με την ένταπορ και με τη φαρμακευτική βιομηχανία μια άλλη συμφωνία. Γιατί όταν ε, προετοιμάζουν κάποια φάρμακα για καλούς σκοπούς, για ιατρικούς σκοπούς, να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν για απάτη ή να μπορούν τουλάχιστον να ανοιχνευτούν στην περίπτωση αυτή. Και τέλος, ο λαθρεμένος κώδικας στον οποίο αναφέρθηκα ετέθησε ισχύ την 1η Ιανουαρίου του 2009. Το πλαίσιο της ΒΑΝΤΑ, έγινε δεχτό από 630 ε, οργανώσεις, αθλητικές οργανώσεις. Πάρα πολλές ε, κυβερνήσεις εγκρίθηκαν μέσω της σύμβασης του UNESCO και υπάρχουν 131 κυβερνήσεις τώρα που έχουν εγκρίνει τη σύμβαση αυτή. Περισσότερες δηλαδή από εκείνες που έχουν εγκρίνει τη σύμβαση για τα δικαιώματα των παιδιών. Όσον αφορά την Ευρώπη, 26 μέλη, χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν επικυρώσει τώρα την σύμβαση αυτή, η οποία ξεκίνησε με μια Ευρωπαϊκή Σύμβαση που ξεκίνησε, αν θέλετε, την διαδικασία αυτή και ενεκρίθη και λειτουργούσε πολύ παλιά πριν σκεφτεί κανένα στην Ουάντα. Δέχτη λοιπόν ότι η Ευρώπη είχε πάντα κατά νου το θέμα αυτό και αυτό οδήγησε, κύριε Πρόεδρε, σε μια πάρα πολύ έντονη πείρα και πολύ μεγάλη πείρα που αναπτύχθηκε μέσω της στενής συνεργασίας που είχαμε με το Συμβούλιο της Ευρώπης, τα κράτη-μέλη και που μας βοηθούν να αναπτύξουμε τον κώδικα αυτό με τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αναπτυχθεί. Όπως είπα και στην εισαγωγή, αναφερόμαστε στο άρθρο 165 της Συνθήκης της Λισαβόνας που αναφέρεται στον αθλητισμό και αναγνωρίζουμε ότι πραγματικά περιμένουμε με ανυπομονησία να συνεργαστούμε με κάθε δυνατό τρόπο μαζί σας. Ο ρόλος μας δεν είναι ρόλος ελεγκτή. Θα πρέπει να έχουμε τη βεβαιότητα ότι όλοι όσοι έχουν προσυπογράψει τη συμφωνία τη σέβονται και συμμορφώνονται. Υιοθετούν πρακτικά τον κώδικα. Συνεπώ, ε, ασκούμε εποπτεία. Έχουμε ένα πρόγραμμα συμμόρφωση και αναφερόμαστε σε αυτό δύο φορέ το χρόνο κατά την διάρκεια των συνεδριάσεων και λέμε πώ ακριβώ εφαρμόζονται οι κανόνε αυτοί. Και θα υπάρξει μια πλήρης έκθεση συμμόρφωση τον Νοέμβριο του 2012. Ο αναθεωρημένος ε, κώδικας, ο οποίος ε, άρχισε να εφαρμόζεται στις αρχές ε, της χρονιάς, είναι ένα έγγραφο στο οποίο έχουν γίνει αλλαγές. Έτσι ώστε να μπορούν να επιβληθούν κυρώσεις για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα. Αυτοί που δεν κάνουν κάτι επί τούτης, απλά και μόνο δέχονται μία προειδοποίηση. Κάτι που δεν υπήρχε, δεν προβλεπόταν στον αρχικό κώδικα. Δεν είναι καινούριο κώδικας, είναι ένας αθεωρημένος κώδικας. Δηλαδή, ο ίδιος ο κώδικας ισχύει ακόμα με ένα περισσότερο ε, αποτελεσματικό τρόπο. Μερικές από τις βασικές αλλαγές που έγιναν στον κώδικα αφορούν την αυξημένη ελαστικότητα των κυρώσεων που επιβάλλονται. Το θέμα της συνεργασίας. Πιστεύω ότι αυτό παρουσιάζει κάποιο ενδιαφέρον. Σε ό,τι αφορά μερικά από τα σπορ που ε, ασκούνται εδώ και αλλού. Υπάρχει ε, μεγαλύτερη εναρμόνιση οι περιπτώσεις αντιμετωπίζονται με πολύ πιο γρήγορους ρυθμούς, υπάρχουν, απαιτούνται υποχρεωτικά προγράμματα, εφαρμογή υποχρεωτικών προγραμμάτων από την κάθε μία από τις χώρες που έχουν υπογράψει και σε περίπτωση που δεν κυρωθεί αυτή η σύμβαση της UNESCO θα προκύψουν συγκεκριμένες επιπτώσεις. Πιστεύουμε ότι αυτό είναι πολύ πιο σοφό από ό,τι γινόταν στο παρελθόν σε περιπτώσεις μη κύρωσες. Τώρα, στον κώδικα του 2003 υπήρχε το whereabouts clause, δηλαδή οι αθλητές θα έπρεπε να κοινοποιούν το σημείο στο οποίο βρίσκονται ανα πάσα στιγμή. Αυτό αφορούσε ιδιαίτερα τους ποδηλάτες που το έκαναν χρόνια. Όταν το αναθεωρήσαμε το 2006, θεωρήθηκε ότι ήταν πάρα πολύ υπερβολικό αυτό και ότι αφορούσε πάρα πολλούς ε, αθλητές. Η όλη δομή λοιπόν εδώ προβλέπει από κάθε χώρα και κάθε ομοσπονδία να ορίζει τους αθλητές οι οποίοι θα πρέπει να υποβάλλονται σε αυτό το τεστ. Αυτό θα πρέπει να γίνεται με βάση τους κινδύνους. Δεν θα πρέπει να φορά όλους τους αθλητές ή λες τους, τους αθλητές Ομοσπονδία επίπεδου. Είναι ένα θέμα που πρέπει να εξεταστεί προσεκτικά. Αυτοί οι αθλητές κοινοποιούν το σημείο που βρίσκονται κάθε φορά έτσι ώστε η Διεθνής Αθλητική Ομοσπονδία μπορεί να ελέγξει που βρίσκονται μία ώρα την ημέρα. Και προσφέρονται για το τεστ αυτό. 13.000 αθλητές έδωσαν τα στοιχεία τους για το πού ακριβώς βρίσκονται πάνω σε αυτή τη βάση. Θα πρέπει να πω ότι οι αθλητές που δεν ανήκουν σε αυτή την ομάδα θα μπορούσαν να υποβληθούν σε εξετάσεις. Δεν χρειάζεται να ανήκει καλή σε αυτή την ομάδα για να είναι επιλέξιμος για ε, ελέγχους αλλά θα πρέπει να ανήκει σε αυτήν την ομάδα για να ε, για να γνωρίζει ε, ο υπεύθυνο ανα πάσα στιγμή που βρίσκεται. Όταν μιλάμε για ομάδα, η ομάδα κοινοποιεί το που βρίσκεται ανα πάσα στιγμή μέσω ενό ατόμου. Μετά από ένα χρόνο εφαρμογής, ε, ε, επανεξετάζομαι και συγκεντρώνουμε στοιχεία για να δούμε κατά πόσον η ελαστικότητα, η διακριτική ευχέρεια που δώσαμε στην περίπτωση αυτή έχει εφαρμοστεί με τρόπο ισότιμο. Γιατί αν όχι θα πρέπει να επιφέρουμε ορισμένες αλλαγές. Αυτή τη στιγμή, κυρία Πρόεδρε, το επανεξετάζουμε το θέμα αυτό το Μάιο θα το συζητήσουμε το θέμα στο Συμβούλιο για να δούμε τι θα μπορούσε να γίνει για να βελτιωθεί ο τρόπος εφαρμογής του. Τώρα, να περάσω σε ένα από τα βασικά προγράμματα που μας απασχόλησαν τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Ξέρουμε ότι Κάθε χώρα έχει ένα πρόγραμμα αντιντόπινγκ και το έχει τα τελευταία 20 χρόνια. Αν κοιτάξετε όμως τον παγκόσμιο χάρτη, θα διαπιστώσετε ότι 130 χώρες δεν έχουν τίποτα, συνεπώς δεν είναι παγκόσμια η οργάνωση. Έχουμε αναπτύξει λοιπόν ένα πρόγραμμα όπου σε ορισμένες περιοχές, περιφέρειες, ιδιαίτερα σε ε, αναπτυσσόμενες ε, χώρες, οι κυβερνήσεις θα μπορούσαν να, συνεργαστούν για να δημιουργήσουν μια περιφερειακή οργάνωση αντιντόπινγκ και να εφαρμόσουν προγράμματα. Και μέσα σε αυτό το, πεντατή, το 54 διάστημα, ε, εντάχθηκαν 120 χώρες σε αυτό το πρόγραμμα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, κυρία Πρόεδρε. Το κόστος ε, για την Γουάντα ε, ήταν πάνω από 2 εκατομμύρια δολάρια. Αυτό δείχνει τη συνεργασία που είχαμε από χώρες, από πολιτικές επιτροπές, από όλο τον κόσμο σε μια προσπάθεια συνεργασίας. Και θα πρέπει να πω ότι είχαμε ιδιαίτερη υποστήριξη από τις ευρωπαϊκές χώρες. Καταφέραμε να πάμε σε αυτές τις περιφέρειες και να εφαρμόσουμε αυτά τα προγράμματα. Και θα πρέπει να πω ότι είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες γι' αυτό. Είπα προηγουμένως ότι ένα από τα βασικά μας καθήκοντα είναι να ασκούμε έλεγχο. Θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι ελέγχουμε τα πραγματικά προγράμματα. Εγώ μπορώ να ελέγξω σήμερα 100 αθλητές και να πω ότι έκανε 100 τεστ και ότι δεν προέκυψε καμία θετική περίπτωση. Κατά συνέπεια ε, είναι καθαρή. Αυτό δεν είναι όμως ε, αποτελεσματικό. Τώρα προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε προγράμματα ποιοτικά και όχι ποσοτικά προγράμματα αποτελεσματικά, προγράμματα σε άμεση συνάρτηση με τα προβλήματα. Και κάνοντας αυτό εξετάζουμε ορισμένες χώρες στον κόσμο που δεν διαθέτουν εθνικά προγράμματα και πραγματικά ελπίζουμε να μπορέσει να γίνει κάτι. Για παράδειγμα, η Βραζιλία δεν έχει πρόγραμμα, η Τζαμάικα, η Ινδία. Η Τζαμάικα μόλις ξεκίνησε, η Νιγερία δεν έχει πρόβλημα, η Ρωσία, σημαντικές πρόοδοι ε, έχουν επιτευχθεί και έχουν τη δική μας στήριξη. Νότιος Κορέα. Ε, ε, και εκεί έχουμε κάνει κάτι στην Τουρκία μόλις ξεκινήσαμε. Υπάρχει και μία, ένα άλλο σημαντικό βήμα που κάναμε σε ό,τι αφορά την εφαρμογή αυτών των κανόνων. Η ε, επιστήμη δεν είναι η πανάκια. Δεν μας βοηθάει να βρούμε τις περιπτώσεις απάτης. Ε, πρέπει να πω ότι υπάρχουν περιπτώσεις που έχουν δοθεί πάρα πολλά δείγματα και μία περίπτωση προέκυψε ε, θετική. Ε, υπάρχουν περιπτώσεις που εντοπίστηκαν από τις διοκτικές αρχές και οι οποίες απεκάλυψαν ότι υπήρχαν περιπτώσεις απάτης. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Σε κάθε περίπτωση έχουμε συνεργαστεί με πάρα πολλές διοκτικές αρχές για να μπορέσουμε να να επιτελέσουμε το έργο μας. Θα πρέπει να κινούμεθα σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές. Η επιστήμη προχωράει. Δαπανίσαμε 50 εκατομμύρια δολάρια στον τομέα της έρευνας. Προσπαθούμε να συνεργαστούμε και με άλλους έτσι ώστε τα προγράμματά μας να μπορούν να εφαρμόζονται. Και έχουμε και ένα ε, βιολογικό διαβατήριο το οποίο θα αρχίσει να χρησιμοποιείται στο Βανκούβερ. Έχουμε ένα σύστημα online που επιτρέπει ε, να κοινοποιούνται όλες οι πληροφορίες σε όλους και πραγματικά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μας βοηθήσατε να βελτιώσουμε τη βάση δεδομένων και που αποτελεί σημαντικό παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής. Αυτό έγινε χάρη σε εσά ε, στην Ευρώπη που μας βοηθήσατε να περάσουμε σε ένα πολύ πιο ε, υψηλού επίπεδου έγγραφο. Το ε, τομέα της ε, εκπαίδευσης έχει καταγραφεί πρόοδος ε, και εκεί προσεγγίζουμε τους νέους με σύγχρονους τρόπους. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τους νέους με τον τρόπο που προσεγγίζουμε ανθρώπους της ε, ηλικίας μας. Τα νέα παιδιά δεν διαβάζουν βιβλία και γι' αυτό το πρόγραμμά μας έχει αναπτυχθεί με βάση την κοινωνική αλληλεπίδραση. Και θα βρείτε ότι στη Σιγκαπούρη θα εφαρμοστεί ένα καινούριο πρόγραμμα. Υπάρχουν προγράμματα που μας βοηθάνε να προωθήσουμε να βοηθήσουμε τους αθλητές, τους νέους αθλητές να μάθουν από τους άλλους αθλητές και να μην νιώσουν ποτέ τον πειρασμό να ε, κάνουν κάποια απάτη. Υπάρχει μια πολύ στενή συνεργασία μεταξύ των κυβερνήσεων και του αθλητικού κλάδου. Αυτό μπορεί να προωθηθεί μέσα από μια συνεργασία ανάμεσα σε εμά και ε, τους υπόλοιπους. Εμείς θέλουμε να συνεργαστούμε με τους εταίρους μας για να το επιτύχουμε. Βασιζόμαστε στους εταίρους μας, βασιζόμαστε και στην ε, τον έλεγχο από το κοινό. Ξέρουμε ότι βρισκόμαστε αντιμέτωποι με προκλήσεις, τις αναγνωρίζουμε αυτές τις προκλήσεις, τις αντιμετωπίζουμε και οι εταίροι μας θα μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις. Αυτό εκ των προτέρων θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Θα συνεχίσουμε να είμαστε καινοτόμοι, θα εξαρτηθούμε από τη συνεργασία με όλους τους εμπλεκόχρονια. χρόνια. Κυρία Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να επαναλάβω ότι βρισκόμαστε εδώ για να, ε, για να προασπίσουμε τα δικαιώματα των καθαρών αθλητών. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Γραμματέα, κύριε Ούμαν. Ακούγοντά σα και είχα ασχοληθεί και λιγάκι με το θέμα, θα έλεγα ο μεγάλος αδελφός σε παρατηρεί. Έτσι κάπου αισθάνομαι. Όρουελα, να μην πω τίποτα χειρότερο. Από την άλλη μεριά βέβαια δεν μπορεί να κάνουμε τίποτα άλλο. Γιατί τόσες ε, απογοητεύσει που ζήσαμε ως θεατές, ως αθλόφιλοι, μπορούν ίσως μόνο έτσι να καταπολεμηθούν. Θα ήθελα όμως να μου πείτε μετά. Αυτό το θέμα με το να ξέρετε που βρίσκονται οι αθλητές έχει προβλήματα και η ανταλλαγή των στοιχείων μπορεί επίσης να οδηγήσει σε καταχρήσεις. Και όπως το ξέρω και από τους συναδέλφους εδώ, το θέμα του Ποια στοιχεία δίνονται πού είναι ένα θέμα που μας απασχολούν πολύ και σίγουρα θα επανέλθουν πολλοί από τους συναδέλφους σε αυτό το σημείο. Πρώτο ερώτημα ο κύριος Σμιτ, αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τέλος αντιπρόεδρος του, ε, του, της ε, Επιτροπής από την Ουγγαρία. Ε, Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Ακούσαμε ότι 26 ευρωπαϊκές χώρες έχουν υπογράψει τη σύμβαση. Μπορούμε να μάθουμε ποια είναι η χώρα που λείπει και ποιες είναι οι ενδεχόμενες κυρώσεις που το απειλούν και κάτι άλλο. Για την έρευνα δαπανούνται τεράστια κονδύλια. Από όσο βλέπω, εκεί που υπάρχει τόπινγκ σήμερα, θα μπορούμε σε 10 χρόνια να το θεωρήσουμε ότι ήταν μέθοδοι τελείως παπελωμένοι, της παλαιοθυλικής εποχής θα έλεγα. Και θα μπορεί να γελάει κανένας μετά από 10 χρόνια. Σήμερα μπορεί να έχουμε ε, ντόπι γονιδίων κλπ. κλπ. Θα ξέρετε πιο καλά από μένα σίγουρα. Το μέλλον λοιπόν δεν είναι και πάρα πολύ ευχάριστο. Εσείς μας είπατε ότι μπορείτε να, δείξετε, να αναγνωρίσετε μέσω διαδικτύου που βρίσκονται εκάστοτε οι αθλητές. Τι γίνεται όμως στις χώρες που δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Εκεί το 70% περίπου των αθλητών δεν μπορούν να έρθουν σε επαφή μαζί σας μέσω διαδικτύου. Τι κάνετε στην περίπτωση αυτή. Νότια Αφρική, ε, Αφρική γενικά, Νότια Αμερική, τίμα της Ασίας. Τι γίνεται στις περιπτώσεις αυτές. Γιατί σήμερα θέλετε να γνωρίσετε κάθε ώρα που βρίσκεται ο αθλητής. Έχω μεγάλες αμφιβολίες ότι εκτός από Ιαπωνία, Κορέα, Αμερική και ε, Ευρώπη μπορεί αυτό να πραγματοποιηθεί σε άλλες χώρες. Και κάτι άλλο που μας απασχολεί είναι η λευκή βίβλος που προτίμασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υπάρχει ένα πρόγραμμα δράσης πια κουμπαρτά που αναφέρει το θέμα της από κοινού καταπολέμησης των καταχρήσεων αυτών του ντόπινγκ. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό. Ευχαριστώ. Ο Sorry, ik was nog even naar de vertaling aan het luisteren van uh, wat mijn collega net zei. Eh, Παρακολουθώ ακόμα την eh, Dat de strijd tegen doping enorm belangrijk is. Die... Θα ήθελα να πω ότι η καταπολέμηση του ντόμπινγκ είναι κάτι το πολύ σημαντικό. Συμφωνώ απόλυτα. Οι αθλητές όμως έχουν και κάποια θεμελιώδη δικαιώματα μεταξύ των οποίων σεβασμός της ιδιωτικής του ζωής. Οι κυρώσεις λοιπόν θα πρέπει να είναι ανάλογες και δεν θα πρέπει να ξεφεύγουν από κάποια νόμιμα πλαίσια. Από όσον ξέρω, στην ε, ΟΑΝΤΑ έχουν ε, ε, γίνει κάποιες προσφυγές. Όσον αφορά αυτό το θέμα του εντοπισμού των whereabouts του κάθε αθλητή, ξέρω ότι υπάρχουν ερωτηματικά. Τι κάνει η ΟΑΤΑ για να προστατεύει τα θεμελιώδη δικαιώματα των αθλητών στην Ευρώπη. κύριε αυτό. Δεύτερον, θα ήθελα να ζητήσω μια άλλη διευκρίνηση. Μου είπατε, μας είπατε ότι έχετε κάποια συμφωνία με τη FIFA για την ε, αναπροσαρμογή κάποιων κανόνων που αφορούν το ποδόσφαιρο. Και βεβαίως ξέρουμε ότι σε κάποια αθλήματα υπάρχει μεγαλύτερη τάση να καταναλώνει κανείς τέτοιες φαρμακοδιαιρετικέ ουσίες από ό,τι άλλο. Στο σκάκι φερρυπίν δεν χρειάζεται κάποιο να το παριστεί, ενώ σε άλλα αθλήματα ναι. Οι πληροφορίες που συλλέγεται επίσης είναι πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσδιοριστεί το περίγραμμα του κάθε ε, αθλητή. Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα. Διότι ο όταν ξέρει κανείς πάρα πολλά όπω για τους ε, τρομοκράτες, μήπως υπάρξει λάθος και αρχίζει και μαζεύει η Ουάντα στοιχεία και για τους αθλητές κατά... Ευχαριστώ. Ασχολούμαι με ένα πρόβλημα που αφορά την Πλάγια κλήρινση, μια σπάνια ασθένεια που πλήττει συνήθω ποδοσφαιριστές. Μεταξύ των αιτίων που το προκαλούν είναι παραλαμβανόμενα τραύματα στα κάτω άκρα, κατάχρηση αντιβιωτικών και χρήση προϊόντων ντόπινγκ σε συνδυασμό με τα ε, ζυζανιοκτώνα που χρησιμοποιούνται ε, ε, στα γήπεδα. Θεωρείτε ότι θα μπορούσε να δημιουργηθεί μια τράπεζα δεδομένων των αθλητών, την οποία θα ε, διοικούν διάφορε ομοσπονδίε όπου θα καταγράφονται τα διάφορα ατυχήματα καθώ και τα φάρμακα που έχει πάρει ένα αθλητή κατά τη διάρκεια τη σταδιοδρομία του. Η Βάντα θα ήθελε να κάνει μια μελέτη σχετικά με την σκλήρινση αυτή και σε ό,τι αφορά την χρήση απαγορευμένων ουσιών. Er Πρέπει να ξέρει πάρα πολλά ο κ. Βαντά για να απαντήσει όλες τις ερωτήσεις αυτές. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι πολύ που ήρθε ο διευθυντής της ΟΑΝΤΑ εδώ για να μιλήσει αυτό το θέμα. Εγώ στη χώρα μου ήμουν γενικός γραμματέας αθλητισμού το 98, αυτό το Άνω Και είμαι πίτιμο μέλος της ε, Ισπανικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Θα ήθελα να κάνω κάποιες συγκεκριμένε ερωτήσεις. Το κόστος των εργαστηρίων αντιντόπιν. Στην Ισπανία, Βερυπίν, συνήψαμε κάποιες συμβάσεις με την Πορτογαλία και πολλές λατινοαμερικανικές χώρες, αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι δεδομένου ότι ε, είναι πολύπλοκο το θέμα, όλο και περισσότερο επενδύσεις χρειάζονται, γιατί πάντα βρίσκονται βήμα μπρο αυτοί που κάνουν τις καταχρήσεις από τις επιστήμες. Υπάρχει κάποιο πρόγραμμα για να βοηθηθούν ε, τα εργαστήρια. Δεύτερον, υπάρχει το θέμα της δικαιοδοσίας. Όταν επιβάλλεται μία κύρωση για τόπιν, πρώτα απ' όλα η Εθνική Ομοσπονδία, η Διεθνή Ομοσπονδία είναι αυτή που επιβάλλει κυρώσει στον αθλητή. Αυτό είναι κάτι που γίνεται αμέσω. Εκ των υστέρω όμω, δεδομένου ότι βρισκόμαστε κράτη δικαίου, μπορεί να κάνει ε, προσφυγή ε, σε διοικητικό ή ποινικό δικαστήριο από τον αθλητή. Όταν ολοκληρώσει την, την αθλητική του κύρωση, αν θέλετε, ο αθλητής, έρχεται και η απόφαση του δικαστηρίου, που μπορεί πολλές φορές να βρίσκεται στην αντίθεση. Τι μπορείτε να προβλέψετε εσείς ότι θα πρέπει να γίνει για να μπορέσουν να συγκεραστούν αυτές οι κυρώσεις. Και επίσης, ε, τι προβλέπετε για κάποιους οι οποίοι είναι εντελώς εκτός ε, της ε, δικής σας δικαιοδοσίας, όπως η NBA. Για να απαντήσετε στις πρώτες ερωτήσεις, κύριε Χάουν, παρακαλώ. Yeah. Αυτό, κύριε Πρόεδρε. Ε, λαμβάνω υπόψη γεγονό ότι ο Big Brother με κοιτάει. Αυτό με προσοχή να απαντήσει στις ερωτήσεις. Προσέξω. Η χώρα που ακόμη δεν έχει κυρώσει τη σύμβαση της UNESCO είναι η Μάλτα. Όσον αφορά την έρευνα, θα πρέπει να πω ότι γνωρίζουμε πολύ καλά δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα, αυτοί που ε, παίρνουν ντόπιν, που το πάρονται, χρησιμοποιούν επιστήμονες που τους βοηθούν. Αυτό είναι το πρώτο λοιπόν. Έχουμε λοιπόν επιστήμονες οι οποίοι τους βοηθούν, να κάνουν την παλιά δουλειά. Δεύτερον, ξέρουμε κάποια πράγματα και ξέρουμε ποιε είναι, είναι αυτοί οι, οποίοι παραβαίνουν τους κανόνες. Υπάρχουν στοιχεία τα οποία ξέρουμε πολλές φορές δεν μπορούμε να τα ε, δημοσιοποιήσουμε. Και πολλέ φορές ξέρουμε ότι χρησιμοποιούνται θα πρέπει λοιπόν ε, να μπορούμε να κάνουμε κάτι ώστε εντό μηνών να αντιδράσουν τέτοιου είδου καταστάσει. Η παραδοσιακή μέθοδο να περιμένουν επιστημονικά αποτελέσματα 4-5 χρόνια είναι όπω είπατε κι εσεί ε, κάτι που ανήκει στο παρελθόν. Προχωρούμε όμως ταχύτητα για να αντεπεξέλθουμε. Τώρα, ύπο, που είναι ο αιματοποιητή που βοηθάει το αίμα. Ξέρουμε ότι υπάρχουν 30-40 διαφορετικά είδη τα οποία κυκλοφορούν. Και ξέρουμε ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πάρα πολλές, σε πάρα πολλές ουσίες. Προσπαθούμε λοιπόν να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να τα ανοιχνεύουμε έγκαιρα. Τώρα έχουμε και ένα συμπληρωματικό ε, πλεονέκτημα ε, το ότι οι φαρμακοβιομηχανίες χρησιμοποιούν νέα ε, είδη και προσπαθούμε με τη δική του συνεργασία να προχωρήσουμε γρήγορα, όπως έγινε στο Πεκίνο. Τώρα, σκολίες. Πού βρίσκουν οι αθλητές αυτές τις ουσίες, με, χρησιμοποιώντας το ίντερνετ, το SMS, το fax και με πολλές άλλες μεθόδους. Άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι το μόνο που χρησιμοποιείται είναι το ίντερνετ. Όλες οι δραστηριότητες ε, τις οποίες αναλαμβάνουμε πρέπει να δούμε κατά πόσων είναι δραστηριότητες οι οποίες αναλαμβάνονται παγκοσμίως. Ίσως κάποιος κάπου μπορεί να βρει την γη της επαγγελίας κατά κάποιο τρόπο για να προμηθεύεται ε, ναρκωτικά και τέτοιου είδους ουσίες. Πιστεύουμε λοιπόν ότι με οποιοδήποτε τρόπο πρέπει να προσπαθούμε να προκαταβάλουμε τα γεγονότα και ελπίζουμε ότι και συνεργασίες μας και τα πλαίσια της Νέας Λευκής Βίβλου θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε ακόμη καλύτερα. Τώρα, κάτι είπε μια άλλη συναδελφό σα για το θέμα τη προστασία τη ιδιωτική ζωή. Αυτό είναι κάτι με το οποίο συμφωνούμε εμείς 100%. Ε, εμείς ε, προσπαθούμε ό,τι κάνουμε να το κάνουμε στα πλαίσια της αναλογικότητας. Αν δείτε την αναλογικότητα, αν δείτε ποιες είναι υπόψεις που εγγράφονται στη δική μας ιστοσελίδα, θα δείτε ότι πάρα πολλά από τα στοιχεία καταγράφονται και ξέρουμε ότι πάντα ζητούμε τους αθλητές να μας ε, δώσουν ε, φερρυπίν δείγμα ούρων όντας γυμνή μπροστά σε κάποιον άλλο. Για να είμαστε πάρα πολύ ε, σίγουροι ότι όλα γίνονται στο φως. Και πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο Ζητείτε μόνο σε ελάχιστους αθλητές παγκοσμίες πολύ ψηλού επίπεδου. Καταλαβαίνουμε το θέμα που θέσατε, καταλαβαίνουμε το θέμα του Βελγίου που αναφέρετε και νομίζω ότι εγώ δεν θα πρέπει να κάνω κανένα σχόλιο επί αυτού. Πρέπει να σας πω ότι δεν θα ήταν σωστό να αναφερθώ σε θέματα τα οποία εκκρεμούν στη δικαιοσύνη. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πάντα εμείς ακολουθούμε τις αποφάσεις που λαμβάνουν οι δικαστικές αρχές. Και αν έρθει κάποια μέρα που αποφασίσουμε ότι πρέπει να αλλάξουμε το σύστημα, το αλλάζουμε. Όπως είδατε, το σύστημα του 2003, οι κανόνες του 2003 άλλαξαν το 2009. Αλλάζουν τα πράγματα και αλλάζουν όταν οι κανόνες που ακολουθούμε και βεβαίω είμαστε ανοιχτοί και σε οποιοδήποτε επικρίσεις και επικοδομητικές παρατηρήσεις όσον αφορά την FIFA. Ποτέ, ποτέ δεν είχαμε καμία ειδική συμφωνία με τη FIFA εμείς. Πρέπει να σας το πω τώρα και το έχω πει εκατομμύρια φορές. Ο κύριος Μπλάτερ, ο πρόεδρος της FIFA, είναι μέλος του Συμβουλίου της Βάντα και πολύ ενεργό μέλος. και οι κανόνες της FIFA συνάδουν με τους δικούς μας κανόνες. Δεν μπορώ να προσθέσω λοιπόν τίποτε παραπάνω. Δεν έχουμε καμία ειδική συμφωνία. Υπάρχουν ε, άλλε διαφορές με τα άλλα αθλήματα. Όχι, οι κανόνες είναι ίδιοι για όλους. Αυτό το οποίο κάνουμε είναι αυτό αυτό το οποίο λέγεται τα whereabouts, ο εντοπισμό τη ομάδα, όταν είπαμε ότι ένα άτομο πρέπει να μα δίνει το στίγμα, Φερρυπίν, που βρίσκεται η ομάδα. Και αυτό είδαμε ότι μπορεί να γίνει. Αυτή είναι η διαφορά, καμία αλλαγή όμω στου κανόνε. Επίση, αναφέρατε το profiling και τη WADA όπως γίνεται για να ε, δοθούν κάποια ειδικά χαρακτηριστικά όπως γίνεται στους ε, τρομοκράτες. Επίσης, είπαμε για το βιοδιαβατήριο. Εμείς έχουμε κάποια στοιχεία προσωπικά που αφορούν τους αθλητές. Το προφίλ λοιπόν, το περίγραμμα του κάθε αθλητή περιέχει κάποια στοιχεία και κυρίως από άποψη ηθικής είναι καθαρός. Κατά κάποιο τρόπο. Αυτή είναι η πρόθεσή μας, επαναλαμβάνω, να προστατεύσουμε τους καθαρούς αθλητές. Ίσως θα θυμάστε το 2006 χειμερινούς αγώνες του ε, Τωρινού ότι απο, ε, απαγορεύθηκε η συμμετοχή κάποιων αθλητών διότι υπήρχε κάποιο πρόβλημα στο αίματος, στην ανάλυση αίματος και πιστεύαμε ότι υπήρχε πρόβλημα ντόπιν. Ο μόνος τρόπος λοιπόν να είναι κανείς σύμφωνος είναι να έχει εκ των προτέρων κάποια στοιχεία που αφορούν προσωπικά τον αθλητή. Σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση την, ε, έχοντας κάνει προηγουμένως για ανάλυση αίματος να ξέρουμε αν πρόκειται για ντόπιν ή για μια φυσιολογική κατάσταση. Επίση, πρέπει να σα πω ότι εμεί δεν είμαστε η ιατρική περιοχή, περι, ε, επιτροπή. Αναφέρομαι στην τελευταία ερώτηση. Δεν μπορώ να σα δώσω τέτοιου είδου λεπτομέρεια. Τώρα, ένα άλλο θέμα πολύ σημαντικό είναι οι τραυματισμοί των αθλητών. Υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις. Όταν ένας αθλητής είναι άρρωστο ή έχει τραυματιστεί και χρειάζεται να του χορηγηθεί μία ουσία που είναι στην απαγορευμένη λίστα μπορεί να υποβάλει αίτηση να του χορηγηθεί για ιατρικούς λόγους. Και αυτό είναι κάτι το οποίο επιτρέπεται ή του χορηγείται μία παρεμφερής ουσία θεραπευτική η οποία δεν βρίσκεται στην απαγορευμένο κατάλογο. Και κάποιοι αθλητές ξέρουμε ότι προσπαθούν ε, μετά από τραυματισμό της ασθένειά τους να γυρίσουν ε, στο στάδιο του συντομάτερο δυνατό και ίσως πολλές φορές να υπερπρόβλημα. Τώρα, όσον αφορά την απάντηση στον ε, Ισπανό εκπρόσωπο. Πρέπει να σα πω ότι ο δικός εκπρόσωπος εκπρόσωπο είναι εξαιρετικός, Έχουμε την υποστήριξη της ομάδας, το ξέρουμε και ξέρουμε ότι έχει. Ε, ε, κατά τη διάρκεια της προεδρίας σας θα προχωρήσει και το πρόγραμμα. Το κόστος του εργαστηρίου είναι κάτι που το αφορά. Υπάρχουν ε, αναγνωρισμένα 35 εργαστήρια αντι-doping, τα οποία είναι διαπιστευμένα, αλλά εντελώς ανεξάρτητα από την Οάντα. Τη δουλειά τους όμως την κάνουν μόνοι τους ανεξάρτητα. Κάποια από αυτά είναι, ανήκουν στον ιδιωτικό τομέα, Κάποια χρηματοδοτούνται από κυβερνήσεις, κάποια άλλα από νοσοκομεία. Δεν συμμετέχουμε εμείς στις δαπάνες. Τα είπαμε ότι είναι ανεξάρτητα σχέση με εμά. Είναι δικό τους θέμα ο εξοπλισμός τους και η λειτουργία τους. Και πρέπει να πω ότι με την Ε, στην Αργεντινή και στο Μεξικό τα διαπιστευμένα εργαστήρια ξέρουμε ότι έχουν συνεργαστεί με εσά για να μπορέσουν να φτάσουν σε πολύ ψηλό επίπεδο. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Τώρα, τα δείγματα. Ε, συγγνώμη, οι κυρώσεις πρέπει να υπάρχει παγκόσμια και αμοιβαία αναγνώριση όλων των κυρώσεων που επιβάλλουν στους αθλητές σε εθνικό ή σε διεθνές επίπεδο για να μην υπάρχουν ε, ε, καταστάσεις όπως ε, αυτές στο παρελθόν όπου δεν υπήρχε ε, συμβατότητα ή αμοιβαία αναγνώριση μεταξύ των διαφόρων κυρώσεων όπως σε μία περίπτωση στο παρελθόν μεταξύ Δανίας και Βελγίου. οι περισσότερες ε, ε ομοσπονδίες ε, αναγνωρίζουν τις κυρώσεις σε εθνικό, σε διεθνές επίπεδο και βεβαίως υπάρχει σε ε, ίστατο βαθμό και η ε, διατησία της Λοζάνης, της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Σήμερα το πρωί βγήκε η απόφαση για μία ε, Γερμανίδα ανθλήτρια η οποία είχε κάποιο πρόβλημα με την απόφαση ενός δικαστηρίου ε, και μετά ομοσπονδιακού. Η Εθνική Ομοσπονδία Μπάσκετ ή Baseball, κυρίως τη ΣΥΠΑ είναι ε, ενώσεις ιδιωτικού δικαίου. Δεν έχουν καμία σχέση με την ε, Ολυμπιακή Επιτροπή, με την ε, κυβέρνηση της ε, Αμερικής. Δεν μπορούμε να τους ελέγξουμε επισήμως αν θέλετε. Ερχόμαστε σε συζητήσεις μαζί τους. Αλλά ε, όποιος συμμετέχει στα πλαίσια διεθνούς ομοσπονδίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες πρέπει να τηρεί τους κανόνες. Όσοι Φερρυπίν ε, πάνε στο Βανκούβαρ φέτος στα πλαίσια των Ολυμπιακών Αγώνων πρέπει να υπακούν στους ίδιους κανόνες. Και πρέπει να σας πω ότι προσπαθούμε με τον κατάλληλο τρόπο όλους όχουν έχουν σχέση με τα ε, σε διεθνείς αθλητικές οργανώσεις και τους Ολυμπιακούς Αγώνες να τους φέρουμε αν θέλετε στα δικά μας τα νερά για να μπορέσουν να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις πρέπει να συμμορφώνουν τους οργανώσεις. Ε, <coughs> ευχαριστώ σας ευχαριστώ κύριε Χοβάν που ήρθατε εδώ. Δεν πρόκειται να επαναλάβω όλες τις ερωτήσεις που έχουν υποβληθεί ήδη. Ιδίω όσον αφορά το στίγμα. Και εγώ θα αναφερώ στο άρθρο 165 της ειδήξης της Λισαβόνας. Μας είναι βέβαια πάρα πολύ αγαπητό. Θα μπορούσε κανένας να αντιδράσει και ε, ανάποδα. Δηλαδή, ίσως αυτό το θέμα του ντόπινγκ ε, έρχεται σε αντίθεση με κάποιες άλλες αξίες Αλλά εγώ για το στίγμα, να σας ρωτήσω για το θέμα που αναφέρατε της αυξημένης ευελιξίας του συστήματος των κυρώσεων. Αυτή η αυξημένη ευελιξία όμως ε, δεν είναι και τόσο ορατή ας το θέμα των ε, παικτών τέννις ε, που αναφέρθηκε προηγουμένως. Και εκτός αυτού, σε μια απάντηση κοινοβουλευτικής ερώτησης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απάντησε ότι θα πρέπει να διατηρηθεί η σωστή αναλογία και ότι η εφαρμογή θα πρέπει να γίνεται ατομικά. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι εξή. Ιδίω όταν εξετάζουμε τη δυνατότητα αθλητών που έχουν τη δυνατότητα προσφυγής ενώπιον των δικαστηρίων, όχι μόνο στη Λοζάνη, αλλά και σε εθνικό επίπεδο που αυτό δεν προβλέπεται αυτή τη στιγμή. Καταλαβαίνω ότι δεν μπορείτε να πείτε τίποτα εσείς για την περίπτωση του αθλητή τένις, αλλά ε, μπορείτε γενικά να μας πείτε κατά πόσο ένα τέτοιο νέο επίπεδο μέσα στα πλαίσια του συστήματος ε, θα μπορούσε να ληφθεί υπόψη. Ιδίως όσον αφορά το θέμα του στίγματος σε σχέση με το θέμα του δικαστηρίου σας ευχαριστώ κύριε Σφαίρ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Χόουμαν, θα ήθελα καταρχάς να υπογραμμίσω τον καθοριστικό ρόλο της Οάντα καθώς και τη δική σας προσωπική συμβολή στην καραποτέ λέμιση της φαρμακοδιέγερσης. Πιστεύετε ότι έχετε αρκετή υποστήριξη από πλευράς των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Γουάντα. Θα ήθελα να σας θυμίσω την σύγκρουση, κάποια παρανόηση, κάποια παρεξήγηση που έγινε το 2007-2008 κατά τη διάρκεια της Γερμανικής και της Σλοβενικής Προεδρίας. Και έγινε μια προσπάθεια να βρεθεί μια λύση στη συνάντηση Λουμπλιάνα το 2008. Ενδεχομένως θα το θυμάστε. Αυτή η σύγκρουση, αυτή η παρεξήγηση οφείλεται στην ε, διαφορά που υπάρχει μεταξύ της οικονομικής υποστήριξης των Ευρωπαίων μελών της ΓΟΑΝΤΑ από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά στην έλλειψη επιρροή στη Βάντα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της Βάντα στις ευρωπαϊκές χώρες. Πώς έχουν τα πράγματα σήμερα. Η επόμενη ερώτηση. Έχετε κάποια ιδέα για το πώς θα μπορούσατε να συμβάλλετε έτσι ώστε τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να διαδραματίσουν ένα πιο σημαντικό ρόλο στη Βόντα. Συνάδελφος Μάρτιν έχει το λόγο. Α. Ευχαριστώ. Είστε πάρα πολύ ξεκάθαρος και το εκτιμώ ιδιαίτερα. Κάνατε αναφορά στον κύριο Μπλάκτε και είπατε ότι είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό, ιδιαίτερα ικανό μέλος του Συμβουλίου. Τι εννοείται ακριβώς με αυτό. Η δεύτερη ερώτηση αφορά τη χώρα μου, την Αυστρία. Όπως ε, και πολλοί άλλοι της γενιάς μου, εγώ είμαι ε, ε, ιδιαίτερος λάτρης των σπορ και ιδιαίτερα των σημερινών σπορ. Και πραγματικά μετάραξαν οι εξελίξεις στον αθλητικό τομέα στην Αυστρία, όχι μόνο σε ό,τι αφορά τη Salt Lake και το Τωρίνο, αλλά για τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσονται τα πράγματα. Έχω την εντύπωση ότι σε ό,τι αφορά την Αυστρία υπάρχουν περισσότεροι κακοί και η συνεργασία με την οργάνωσή σας είναι χειρότερη από ό,τι είναι σε ό,τι αφορά άλλες χώρες. Μπορείτε να το επιβεβαιώσετε αυτό. Πραγματικά υπάρχει ένα πρόβλημα που αφορά την Αυστρία και μόνο είναι μια, ε, ένα μήνυμα που προωθείται από τα μέσα ε, ενημέρωσης και οφείλεται στο γεγονό ότι η Αυστρία είναι μια μικρή χώρα, έχει ε, πολύ λίγους αθλητές. Ότι υπάρχουν πολλά συμφέροντα θα, με ενδιαφέρει ιδιαίτερα να ακούσω τη δική σας άποψη σχετικά με αυτό το θέμα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να αναφερθώ για άλλη μια φορά στο θέμα της συνεργασίας των, της ΒΑΝΤΑ με τις εθνικές ε, ε, οργανώσεις ε, κατά πολέμησης φαρμακοδιέργεσης. Είχατε πει ότι ε, υπάρχει μια προσπάθεια να υπάρχει εναρμόνιση, σύγκληση αν θέλετε των αποφάσεων για κυρώσει στι διαφορέ ομοσπονδίε. Εγώ στο παρελθόν είχα μάλλον την εντύπωση ότι αυτό δεν γίνεται ακόμα και ότι υπάρχουν τεράστιε δυσκολίε και διαφορές μεταξύ της επόφασης μιας εθνικής ε, ομοσπονδίας ε, και οργάνωσης κατά της φαρμακοθεραπείας και της απόφασης ΒΑΝΤΑ. Κάτι να μου πείτε λοιπόν πάνω στο θέμα αυτό της συνεργασίας σε αυτό το τομέα. Και κατόπιν θα ήθελα να αναφερθώ ε, με δύο λόγια στο θέμα της δήλωσης στίγματος. Ε, είπατε ότι προσπαθείτε να επανεξετάσετε αυτό το σύστημα και να δείτε που υπάρχουν προβλήματα και που θα μπορούσε να βελτιωθεί. Θα πρέπει νομίζω ακριβώς και για την προστασία των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων των αθλητών να προσέξουμε να μην υπερβάλλουμε και θα πρέπει να υπάρχει πάντα μια αναλογικότητα των μέσων. Μέχρι στιγμής ξέρω ότι οι αθλητές έπρεπε από τρει μήνες από πριν να πούνε πού θα βρίσκονται. Δεν ξέρω πόσοι από εμά μπορούν να πούνε τρει μήνες προηγουμένω πού θα βρίσκονται μετά από τρει μήνες και τι θα κάνουν όλη την ημέρα. Και να το αποτούμε αυτού του αθλητέ και μετά να του. να τους επιβάλλουμε κυρώσεις εάν, όχι πατήσανε, απλώς ε, δεν το έκαναν μέσα στους, ε, στην περίοδο αυτών των τριών μηνών, αλλά μια-δύο μέρες καθυστέρηση. Θα ήθελα να μου εξηγήσετε λοιπόν εδώ κατά πόσον είναι κάτι το οποίο θα σας απασχολήσει και κατά πόσον θα μπορούν αυτές οι παράλογες κυρώσεις ε, για αυτό το θέμα, δηλαδή όταν η δήλωση στίγματος για τόσο μακριά στο μέλλον δεν γίνει την ακριβή στιγμή, εάν θα μπορούσατε κάτι να κάνετε, αν καταβάλλουν προσπάθειες να διατηρήσετε δηλαδή μια αναλογικότητα των κυρώσεων και να διασφαλίσετε και τα δικαιώματα των πολιτών αθλητών. Ευχαριστώ. Πρώτα, ευχαριστώ. Τέσσερις έχουν ακόμα ζητήσει το λόγο. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω κύριε Χάμαν να μας δώσετε σύνομες απαντήσεις, γιατί είπαμε έχουμε άλλες Τέσσερι ερωτήσει. Απαντήστε σύνομα λοιπόν σε αυτά που ερωτήθηκαν ήδη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Όσον αφορά την πρώτη ερώτηση για το στίγμα πάντα, να σας το εξηγήσω λίγο καλύτερα. Γιατί σωστά είστε καλά ενήμεροι. Μόνο οι λίγοι αθλητές σε ένα κατάλογο δεν δηλωμένο πρέπει να δίνουν το στίγμα τους. και τους λέει η χώρα τους ότι βρίσκονται σε αυτό το, ε, το κατάλογο και θα πρέπει τρεις μήνες από πριν να δηλώσουν και μέσα στους τρεις μήνες να μπορούν να αλλάξουν. Δηλαδή με ένα SMS μπορούν να αλλάξουν τη δήλωση αυτή. Πραγματικά και η ζωή μου δεν διαφέρει πολύ από αθλητή και δεν μπορώ να σας πω πουθενά καθόλου που θα είμαι μετά από τρεις μήνες. Και, σας το λέω, οι περισσότεροι αυτοί από τους αθλητές καθημερινά είναι στο facebook, στο twitter. Έχουν δηλαδή κάποια δυνατότητα ενημέρωσης συνεχώς. Και, μπορώ κι εγώ που δεν είναι και πολύ νέος να το κάνω. Αν μπορώ εγώ θα μπορούν και εκείνοι. Και αν ένας αθλητής δεν δηλώσει που βρίσκεται, τους στέλνουν ένα μήνυμα. Και έχει το δικαίωμα να απαντήσει στο μήνυμα αυτό ο αθλητής και να δώσει μια δικαιολογία. η δικαιολογία αυτή είναι λογική, δεν μετράει. Προτού περάσει δηλαδή στη διαδικασία κύρωσης θα πρέπει να υπάρχουν τρεις αποτυχίες. Σας λέω, αν μπορεί να δώσει μια δικαιολογία, μια φορά, εντάξει. Εάν το ξανακάνει, θα του πούνε, α, τώρα έχει άλλε δύο δυνατότητες. Και αν έχει τρεις αποτυχίες δήλωσης, τρεις ελλείψεις δήλωσης, μέσα σε ένα χρονικό διάστημα, τότε μπορεί να ε, επιβληθούν κυρώσεις. Όπως σας είπα, από την 1η Ιουνίου του 2009, τρεις αθλητές μονάχα δεν κατάφεραν να μας δηλώσουν. Δηλαδή άλλες 13.000 αθλητές που μας έδωσαν το στήμα του 1η Ιανουαρίου του 2009 δεν απέτυχαν, μας ενημέρωσαν πάντα. Αυτή είναι σήμερα η κατάσταση. Αν είμαστε ανοιχτοί για αλλαγέ, φυσικά. Αυτή τη στιγμή έχουμε πέντε δράσει. Πέντε περιπτώσει σε οποίες συμμετέχουμε και που ζητήσαμε το δικαίωμα να μπορούμε να παρέμβουμε. Ναι, είμαστε σίγουροι ότι τα διάφορα δικαστήρια έχουν όλες τις πληροφορίες που μπορούμε να τους δώσουμε. Γιατί πιστεύουμε ότι ο καλύτερος τρόπος να εμπλακούμε είναι να δίνουμε πλήρες πληροφορίες. Είμαστε δηλαδή, αν θέλετε, φίλοι του δικαστηρίου. Δίνουμε τις πληροφορίες αυτές. Ο φίλος από τη Σλοβενία ρώτησε τι γίνεται όσον αφορά την ε, ευρωπαϊκή ε, επίδραση. Η δομή του Συμβουλίου είναι η ίδια. Αλλά με κοιτάξουμε τις ομάδες εμπειρογνωμόνων, που έχουμε τέσσερις ομάδες εργασίας και πέντε ομάδες εμπειρογνωμόνων. Το 50% από τα μέλη στις ε, εννέα αυτές επιτροπές είναι Ευρωπαίοι. Και αυτό δείχνει ξεκάθαρα νομίζω πολύ επίδραση. Και εκτός αυτού την αναγνώριση της εμπειρογνωσίνης που έχουν οι Ευρωπαίοι. Ξεκολουθούμε λοιπόν να αναγνωρίζουμε πού υπάρχουν οι ικανότητες αυτή τη στιγμή και να την εκμεταλλευόμαστε. You ποιο είναι το αποτελεσματικό μέλος της Ουάντα. Εγώ ε, σας κάνω μια παρουσίαση ε, της Ουάντα. Όταν λέω εγώ ε, αποτελεσματικό είναι ο κύριος Μπλέντερ έρχεται στην συνεδριάσεις μας, συμμετάσχει στις συνεδριάσεις, έχει πολύ καλές σχέσεις εργασίας με τον πρόεδρο. Είχα μια πολύ ε, καρποφόρα συνέντευξη στη Ζυρίχη τον Οκτώβριο πάνω σε κάποια τα θέματα που θίγησαν και εδώ και το αποτέλεσμα ήταν ότι η FIFA αποδέχτηκε ότι αυτό που έκαναν έπρεπε να τροποποιηθεί. Και καταλήξαμε σε μετερική σχέση με τη FIFA και εξετάζουμε την έρευνα από κοινό. Και θα μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε ίσως ε, κάποια έρευνα σχετική. Κάθε χώρα στον κόσμο έχει ένα πρόβλημα με την φαρμακοδιέργηση. Καμιά χώρα δεν είναι ε, ικανή να πει ότι δεν έχει το πρόβλημα αυτό. Κανένας βέβαια θέλει η χώρα του να έχει περιπτώσεις τόπινγκ. Αλλά νομίζω ότι η χώρα δεν έχει κανένα πρόβλημα φαρμακοδιάργησης τόπινγκ σφάλεται. Εγώ είμαι κάποιος που βασίζομαι σε κανόνες και δίνω τα αποτέλεσμα με τους κανόνες. Εγώ θα έλεγα, η Αυστρία είχε πρόβλημα το 2002, είχε πρόβλημα το 2006 και ελπίζουμε να μην έχει πρόβλημα το 2010. I was asked in, uh, Madam Chair, about uh, the harmony between. Uh, Κοιτάξτε, είπατε ποια είναι η σχέση τώρα μεταξύ ΒΑΤΑ και εθνικών εργασμών. Είμαστε ένα γενικό σώμα. Στην κάθε χώρα, κάθε ομοσπονδία έχει τους δικούς κανόνες. Εμείς μπορούμε να δώσουμε τη δυνατότητα σε εκείνες χώρες που πιστεύουν ότι μέχρι στιγμής δεν είχαν εισακουστεί να εισακουστούν. είναι το ίδιο βέβαια όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν είναι κάθε μέλος που έχει γράψει τους κανόνες προς οποίους λειτουργεί. Όχι, αλλά προσπαθούμε να, και εμείς να έχουμε μία συνένεση πάνω στους κανόνες. Εμείς δεν παρεμβαίνουμε επί έξι μήνες για να έχουμε πλήρη διαβούλευση όταν υπάρχει ένα πρόβλημα. Λοιπόν, έχουμε παρέμβει, θα ξαναπαρέμβουμε αν χρειαστεί. Εάν κάποιος από τους κανόνες, κανένα από τα πρότυπά μας, χρειάζεται αλλαγή, θα το κάνουμε. Και αυτό μπορεί να γίνει μέσα σε κάποιους μήνες. Λοιπόν, τονίζω, πρέπει να διαβουλευόμαστε και πρέπει να διαβουλευόμαστε με τέτοιο τρόπο που να διαφανής και να ικανοποιεί τους πάντες. Δεν θέλουμε να υπεβάλλουμε. Μην πετάξουμε το μωρό μας με τον, με νερό του μπάνιου του μωρού. Υπάρχουν διαφοροποιημένες κυρώσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και μπορούν να εφαρμοστούν. Ο καθένας προσπαθεί βέβαια το δικαστήριο να το πείσει ότι δεν έσφαλε και αν το καταφέρει ίσως δεν ε, τιμωρηθεί καθόλου γιατί αρχίζουμε με μια προειδοποίηση και τελειώνουμε με, μια, με ένα αποκλεισμό δύο ετών. Και θα πρέπει ο καθένας βέβαια να έχει τα επιχειρηματά του, τα μπορεί να τα υποβάλει. Στο παρελθόν, ε, τότε που ήταν αυτόματη η επιβολή των δύο ετών αποκλεισμού, αυτό έχει περάσει. Υπάρχει λοιπόν σήμερα ευελιξία. Τώρα θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία ναι, εάν αυτό δειχθεί αναγκαίο. Εάν δειχθεί αναγκαίο, θα το σκεφτούμε, θα το μελετήσουμε. Αυτά μπορώ να σας πω, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Arvoisa rouva puheenjohtaja, kaksi kysymystä. Κοιτάξτε, από ό,τι φαίνεται, Πρόεδρε, Υπάρχει εδώ πρόβλημα ε, υγείας, δημόσιας υγείας και στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο. Ε, βεβαίως ε, υπάρχουν πολλά άλλα μεγαλύτερα προβλήματα από τον αθλητισμό. Τι μπορεί να κάνει η Γουάντα σε σχέση με αυτό το πρόβλημα. Ε, θίξατε το θέμα της ε, ε, χειραγώγησης των δόλων χειρισμών στα γονίδια. Αυτό όμως γίνεται με τη βοήθεια των γιατρών, γιατί για να γίνει κάτι τέτοιο χρειάζεται και η βοήθεια ειδικών. Δεν βοηθάει και πολύ ο όρκος του υποκράτη οι γιατροί βασικά θα έπρεπε να ε, σώζουν τους ανθρώπους, αλλά ε, ξεπουλούν την ηθική τους και καταστρέφουν ζωές. Η Γουάντα πώς ακριβώς βλέπει την ιατρική και το ρόλο των γιατρών. Και αν κάποιος γιατρός συλλαμβάνεται να παρανομεί, ε, και αυτό θα τιμωρηθεί όπως και οι αθλητές. Κύριε Παλιαδέλη. Δύο πολύ σύντομε ερωτήσει, κύριε Χόμαν. Ε, μιλάτε για έρευνα, στην οποία από το 2001 δόθηκαν 50 εκατομμύρια δολάρια θα μπορούσατε να μας εξηγήσετε τι είδου έρευνα, είναι επιστημονική, είναι στατιστικά. Και μια δεύτερη πολύ σύντομη επίσης, σε έναν χάρτη του κόσμου, της ε, παγκόσμιο, ε, έχουμε διάφορα χρώματα με χώρες που έχουν ε, με διάφορα, σε διάφορα επίπεδα αποδεχτεί τον κώδικα για το αντιντόπινγκ. υπάρχουν στατιστικά στοιχεία που να δείχνουν τα αποτελέσματα της εφαρμογής αυτού του κώδικα ε, σε σχέση με τα περιστατικά ε, ντόπινγκ στις συγκεκριμένες χώρες. Ευχαριστώ. Szanowna Pani Przewodnicząca, e, faktycznie wysłuchując i Ακούγοντας τα στατιστικά δεδομένα, νομίζω μπορούμε να ισχυριστούμε ότι τρελάθηκε ο κόσμος από ό,τι φαίνεται όλοι θέλουν να είναι επιτυχημένοι στο άθλημά τους. Ε, δεν είναι εύκολο όμως να εντοπίσει κανείς ε, τους ε, απαταιώνες γιατί η τεχνολογία εξελίσσεται συνεχώς. Εδώ μιλάμε για ηθική και, το, και διεντολογία και το ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσον έχει αναλυθεί σωστά το πρόβλημα της ε, φαρμακοδιέγερσης διότι ας μην ξεχνάμε ότι οι αθλητές βρίσκονται υπό την επιρροή των προπονητών και το, της ομάδας των γιατρών και πολύ συχνά οι ίδιοι αθλητές ε, δεν έχουν ειδικέ ε, ιατρικές γνώσεις. Ως ε, εκ τούτου, οποτεδήποτε πρόκειται για κατάχρηση ουσιών, πρέπει να δούμε ποια είναι, πόση, κατά πόσον φέρει ευθύνη ο προπονητής και ενδεχομένως και η ομάδα των γιατρών. Υπάρχει αυτό το τρίγωνο, ο αθλητής, ο προπονητής και ο, αθλητή, ο αθλητίατρος, ε, αυτοί όλοι εμπλέκονται στο παιχνίδι και για να περιορίσουμε την φαρμακοδιέγερση πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τις συνέπειες που υπάρχουν στην ΟΛΕ. Η Πρόεδρος, κοιτάξτε μια ερώτηση μου επιτρέψτε. Όσον αφορά τη μεταφορά ε, προσωπικών δεδομένων. Εδώ πραγματικά έχουμε να κάνουμε με θέμα δεοντολογίας, γιατί αυτό άπτεται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το Κοινοβούλιο ε, έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο επ' αυτού και θέλω να ρωτήσω. Τι γίνεται αν ένας αθλητής ε, στη ζωή του, στη σταδιοδρομία του έχει ε, αρρώστια ή έχει κάποια στιγμή ε, κάνει χρήση ήπιων ναρκωτικών, καταδικάζεται. Ε, αυτά τα δεδομένα πάνε στο Μονρεάλ και από το Μονρεάλ πού πάνε μετά. Δηλαδή, αν ε, θέλει ο αθλητής να εμφανιστεί κάπου, οποιοδήποτε έχει πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα και μπορεί να ισχυριστεί όχι, δεν τον ε, θέλω αυτόν τον αθλητή, διότι α πούμε όταν ήταν ε, πολύ νέος έκανε κάποια ήπια χρήση ναρκωτικών ή γιατί είναι ομοφυλόφιλο. Υπάρχουν πολλά πράγματα ε, που υπάρχουν στη ζωή των ανθρώπων και αυτά δεν είναι προς δημόσια χρήση, είναι καθαρά ατομικά δεδομένα, δεν είναι για τον καθένα. Εμείς λοιπόν ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ίσως εδώ μπορείτε να μας βοηθήσετε, ότι δυστυχώς ε, τέτοιου είδους δεδομένα δεν διαφυλάσσονται με ασφάλεια ε, και δεν βρίσκονται κάπου σε ένα υπόγειο στο Μορεάλ ε, ασφαλισμένα, αλλά κυκλοφορούν γενικώ ανά τον κόσμο. Αυτή ήταν η τελευταία ερώτηση που ήθελα να σας κάνω και αν δεν έχετε άλλες ερωτήσεις θα ήθελα να μου τρέψει να δώσω το λόγο για λίγα λεπτά στην Κομισιόν. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ στο θέμα της ε, δημόσιας υγείας. Κοιτάξτε, το θέμα αυτό μας απασχολεί πάρα πολύ και έχουμε απευθυνθεί στους, ε, στις κυβερνήσεις ε, για να μας βοηθήσουν διότι τα θέματα που έχουν σχέση με τα στεροειδή και άλλες απαγορευμένες ουσίες δεν είναι θέμα αθλητισμού και αθλητή. Ε, είναι γενικότερα δημόσια υγείας. Ε, τα γυμναστήρια, παραδείγματο χάρη. Εκεί, στα γυμναστήρια, υπάρχουν ε, πολλοί που μοιράζουν και πολλούν, διακινούν απαγορευμένες ουσίες. Η συνθήκη της UNESCO, στην οποία έχουν προσχωρήσει τα περισσότερα κράτη-μέλη που παρίστανται, αναφέρει ότι κάθε κράτος οφείλει να υπάρχει νομοθεσία που απαγορεύει την ε, διακίνηση αυτών των απαγορευμένων ουσιών. Άρα δηλαδή αυτή είναι η απάντηση. Πρέπει να πείσουμε την UNESCO να μεριμνήσει για την εφαρμογή αυτής της ε, συνθήκης, γιατί όπως σας είπα υπάρχει νομοθεσία περί απαγορευμένης διακίνησης. Ξέρω, ας πούμε, το δικό σας ε, το κράτος, η Γερμανία, έχει τέτοιες νομοθεσία και ξέρω και ένα πολύ καλό παράδειγμα όπου ίσχυσε αυτό. Αυτά που λέμε δεν είναι λοιπόν δική μας ευθύνη, αλλά αρμοδιότητα των κυβερνήσεων με τις οποίες συνεργαζόμαστε. Όσον αφορά το θέμα των γιατρών, νομίζω ότι το θέμα αυτό ετέθη επίσης σε κάποια ερώτηση. Εμείς πιστεύουμε οι γιατροί πρέπει να τιμωρούνται και οι ιατρικοί σύλλογοι που είναι αρμόδιοι για αυτούς θα πρέπει να τους αποσύρουν την άδειά τους. Ο γιατρός ε, όταν παραβιάζει έναν κανόνα χορηγώντας μία απαγορευμένη ουσία τότε θα πρέπει να ε, υφίσταται τις πειθαρχικές κυρώσεις. Δεν είναι ότι θα πρέπει μια ομάδα να τον απορρίπτει ως γιατρό, αλλά και οι ε, χώρες θα πρέπει να λένε, κοιτάξτε, ε, πρόκειται για πειθαρχικό παράπτωμα και αυτεπάγγελτα περνάτε μέσα από πειθαρχική δίωξη. Το ίδιο ισχύει και για τους ε, δικηγόρους και ενδεχομένως και για άλλα επαγγέλματα που εμπλέκονται σε τέτοιου είδους δραστηριότητες. Για να απαντήσω στην ερώτηση που τέθη σχετικά με την έρευνα. Κοιτάξτε, εμείς δαπανάμε περίπου το 25 μέχρι 30% του ετήσιου προπολογισμού μας για την έρευνα. Μιλάμε για 25 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, αυτό είναι ο προπολογισμό μα. Βλέπετε λοιπόν ότι τα κονδύλια που διοχετεύονται στην έρευνα είναι σημαντικά. Βέβαια, στον κόσμο της έρευνας μιλάμε για σταγόνα εν το ωκεανό. Ως εκ τούτου, ε, απευθυνόμεθα σε άλλους για να μας βοηθήσουν να αυξήσουμε τα κονδύλια αυτά για την έρευνα. Ε, επίσης, ρωτήσατε για τα στατιστικά δεδομένα και την συμβατότητα. Εμείς ε, έχουμε καταθέσει μια έκθεση περί συμβατότητας στατιστικών δεδομένων, που δεν έχω μαζί μου, αλλά μπορείτε να την βρείτε στην ιστοσελίδα μας. Και εκεί μπορείτε να δείτε ποιος ε, δεν εφαρμόζει τους ε, κείμενους κανόνες. Πρέπει να έχετε κατά νου ότι αυτή η έκθεση για τους κανόνες έχει σχέση με ε, την έκθεση που δημοσιεύτηκε στις 31 Δεκεμβρίου του 2008, άρα δηλαδή έχει πλέον θεωρείται παροχημένη έκθεση αυτή. Τώρα εμείς έχουμε προχωρήσει στην σύσταση σύνταξη μια νέα έκθεση που θα αφορά το 2009. Νομίζω ότι απάντησα ήδη στην ερώτηση σχετικά με την ομάδα των γιατρών και τις ε, κυρώσεις εις βάρος εκείνων που πείθουν τους ε, ε, αθλητές. Όμως, στον προπονητή και σε οποιονδήποτε άλλο συμμετέχει στην ομάδα θα πρέπει να εξηγηθεί επακριβώς περί τίνος πρόκειται. Το θέμα είναι ποιος έχει την αρμοδιότητα να επιβάλλει κυρώσει σε ένα και συγκεκριμένο άτομο. Μερικές φορές ε, είναι ο ίδιος ο αθλητισμός, άλλες πάλι φορές ο αθλητισμός λέει ή μπορεί να ισχυριστεί ότι ε, δεν μπορούμε εμείς ε, να επιβάλλουμε κυρώσεις ε, στου εθνικού προπονητέ. σω θα πρέπει να το κάνουν οι κυβερνήσει. Και γι' αυτό λέμε στι κυβερνήσει, ξέρετε να κάνετε, να αποσύρετε τη χρηματοδότηση, να αποσύρετε την έγκριση του προπονητή ή του γιατρού γιατί δεν το αξίζουν. Και ως εκ τούτου, όπως σας είπα, προσβλέπουμε στη συνεργασία με τις κυβερνήσεις για να μας βοηθήσουν. Ε, κυρία Πρόεδρε, αναφερθήκατε στη μεταφορά των δεδομένων. Εμείς συνεργαζόμαστε στενά τόσο με την Κομισιόν όσο και με το Συμβούλιο της Ευρώπης και φαντάζομαι ότι θα γνωρίσετε πολύ καλά ε, το άρθρο 29 της έκθεσης της ομάδας εργασίας. Είχαμε συναντήσεις με την Επιτροπή ε, και τον Νοέμβρη που μας πέρασε και υπάρχει ένα θέμα το οποίο εξακολουθεί να είναι ανοιχτό προς ε, συζήτηση το θέμα της διατήρησης των πληροφοριών και για ποιο χρονικό διάστημα. Οι πραγματικές πληροφορίες είναι ε, εκείνες οι οποίες αν παραβιωθούν οδηγούν σε κυρώσεις. Και αυτό πρέπει να δημοσιεύεται, να κοινοποιείται. Γιατί δεν μπορούμε, ας πούμε, ένας ε, ποδηλατής ε, να τιμωρηθεί για στην ποδηλασία και μετά να πάει στο τρίαθλο και να αγωνιστεί σε αυτό το άθλημα. Ε, δεν είναι δυνατόν να συμβεί κάτι τέτοιο. Άρα, δηλαδή, οι πληροφορίες σε κάποιο βαθμό πρέπει να διακινούνται για να αποδεικνύεται και ότι τα δικαιώματα του καθαρού αθλητή διαφυλάσσονται. Τίποτα άλλο, τίποτα παραπάνω. Δεν μπορεί, ας πούμε, ένας αθλητής που παραβιάσει του ε, στη Γερμανία, αυτό να πάει στην Αζηλανδία και να αποκρύψει ότι έχει τιμωρηθεί. Δεν γίνεται αυτό για να υπάρχει ε, αρμονική εφαρμογή σε όλο τον κόσμο, σε όλα τα αθλήματα. Πρέπει να υπάρχει κάποια διακίνηση πληροφοριών. Αυτό είναι το σκεπτικό που έχουμε ε, και που θα χρησιμοποιήσουμε και στις συζητήσεις με την Κομισιόν. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ναι, αλλά τίθεται το ερώτημα για πόσο χρόνο, για ποιο χρονικό διάστημα θα διατηρούνται τα δεδομένα. Η Κομισιόν έχει το λόγο για δύο λεπτά, εάν το επιθυμεί, και παρακαλώ να πει κάτι που με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Σε αυτόν τον τομέα της φαρμακοδιάγερσης, το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι ε, πραγματικά ο μεγάλος μας αδελφός. Ίσως αυτό να μην το γνωρίζουν πολύ και ίσως εσείς μπορείτε να προβάλλετε αυτή τη στενή σχέση που υπάρχει. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, πολύ σωστά ο κύριος Χάρμον αναφέρθηκε ε, στις νέα διατάξεις για τον αθλητισμό που περιλαμβάνονται στη συνθήκη της ε, Λισαβόνας. Ε, πρέπει να προστατεύεται η δεοντολογία και η ακαιρεότητα του αθλητή. Άρα δηλαδή καλούνται οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμβάλλουν στον αγώνα κατά της ε, φαρμακοδιάγερσης. Παράλληλα ε, πρέπει να σεβόμεθα τον ρόλο όλων των ε, παραγόντων που δραστηριοποιούνται, ο δικός μας ο ρόλος να είναι συμπληρωματικό σε αυτόν του Συμβουλίου της Ευρώπης, των κρατών μελών και των αθλητικών συλλόγων. Η Κομισιόν κατά τη διάρκεια του έτους ε, θα παρουσιάσει την ε, πολιτική της για τον αθλητισμό με βάση τις νέες διατάξεις της συνθήκης. Άρθρο 165 της συνθήκης. Επειδή υπάρχει αυτό, ε, θεωρώ ότι η απάντηση της Κομισιόν θα λάβει τη μορφή δύο εγγράφων. Αφενός έχουμε κατά νου έγγραφα χάραξης πολιτικής. Ο αγώνας κατά το ντόπινγκ είναι πολύ πιθανό να περιλαμβάνεται σε αυτά τα δύο έγγραφα. Και επίσης ε, προτιθέμεθα να καταθέσουμε μια πρόταση για τη χάραξη προγράμματος για τον αθλητισμό, όπως μας ζήτησε να το πράξουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εγκρίνονται μέσα από την πεπατημένη της νομοθεσίας, άρα το ερώτημα κατά πόσον ο αγώνας κατά του ντόπινγκ θα ε, στηριχθεί όχι, αυτό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Συμβούλιο της Ευρώπης. Η Κομισιόν έχει ε, δρομολογήσει ε, διαδικασίες διαπραγματεύσεων με τους άμεσα εμπλεκόμενους έτσι ώστε να υπάρχει ένα καλό πρόγραμμα για το μέλλον. Οι διαπραγματεύσεις αυτές μόλις έχουν ξεκινήσει αλλά ήδη υπάρχουν πολλές ενδιαφέρουσες απόψεις που μας τις έχουν εκφράσει πολλοί παράγοντες που δραστηριοποιούνται στον τομέα του ντόπινγκ. Και επιτρέψτε μου να σας δώσω κάποια τροφή για σκέψη. Σύντομα λοιπόν θα αναφέρω κάποιες από αυτές τις σκέψεις. Έχοντας κατά νου ότι η είναι και οι άλλοι παρεμφερείς ε, φορείς ε, εστιάζουν την προσοχή τους στον πρώτο αθλητισμό, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδέχεται να ασχοληθεί περισσότερο με τον εραστεχνικό αθλητισμό ε, και τον αθλητισμό για τη φυσική κατάσταση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στον προϋπολογισμό του 2010 έχει συμπεριλάβει κάποια κονδύλια για να γίνει πειραματική χρήση προγραμμάτων. Γνωρίζουμε ότι οι αποφάσεις που επηρεάζουν το σύστημα του αντιντόπινγκ doping εκφράζονται κυρίω σε βήματα όπου δεν συμμετέχει όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό μας προτάθηκε ε, λόγω της συνθήκης της Λισαβόνας η Ευρωπαϊκή Ένωση να σκεφτεί, να προσχωρήσει σε σημαντικές συνθήκες αντιντόπινγκ όπως είναι αυτή του Συμβουλίου της Ευρώπης και της UNESCO. Και τέλο, θα ήθελα να αναφέρω ότι η Κομισιόν ε, συμμετέχει ενεργά σε συζητήσει που έχουν άμεση σχέση με την προστασία των ε, προσωπικών δεδομένων, ε, τη φαρμακοδιέγερση, τη συνεργασία ανάμεσα σε διαπιστευμένα εργαστήρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλα θέματα, τα οποία ανέφερε ο κ. Χάρμον. Ε, έτσι λοιπόν αυτά ε, θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν και στο ε, προγραμματισμένο έγγραφο που σας είπα και στο πρόγραμμά μας. Πολύ ωραία λέει η Πρόεδρος, πολύ επικοδομητικά όλα αυτά και ευχαριστώ που ήσασταν και σύντομος. Νομίζω ότι είπατε και ορισμένα πράγματα τα οποία θα τα εξετάσουμε στο μέλλον και θεωρώ ότι το Κοινοβούλιο θα στηρίξει την Κομισιόν, όταν θα καλέσουμε εμείς την Κομισιόν να υπογράψει ε, τη συνθήκη. Αυτό το δικαίωμα πλέον το έχουμε. Υπάρχει νομική βάση και πρέπει να προχωρήσουμε. Γιατί αυτό θα είναι και ένα καλό δείγμα για τη στράτευσή μας στον αθλητισμό. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και τον κύριο Χάρμον. Νομίζω ότι ήταν πολύ σημαντικό για όλους μας να μας πείτε πώς λειτουργούν όλα αυτά και μπορείτε να είστε σίγουρος ότι εμείς στον αγώνα κατά της φαρμακοδιάγευσης, είμαστε στο πλευρό σας, αλλά και υπέρ της διαφύλαξης της διοντολογίας. Ε, για αυτό το θέμα είμαστε πολύ προσεκτικοί, ε, δικαίως βέβαια, ε, γιατί γι' αυτό μας εξέλεξαν και μεριμνούμε έτσι ώστε να υπάρχουν ε, προσαρμογές. Ε, και η Κομισιόν θα σας βοηθήσει. Η Κομισιόν πάντα βοηθάει. Και έτσι λοιπόν ε, μπορούμε και μέσω Κομισιόν να είμαστε πάντα σε επαφή. Ευχαριστούμε πολύ και τους συναδέλφους. Έχουμε τώρα την Ισπανίδα Υπουργό Πολιτισμού κοντά μας.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 I speak in German. Sehr gut. Ja, verstehen Sie Deutsch? Das ist ja wunderbar. So, vielen Dank, Frau Minister. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Υπουργέ, που ήρθατε. Κυρία Υπουργέ Άγγελες Κονσάλη Σίντε, δεν ξέρω αν ε, πρόφερα καλά το όνομά σας. Άγγελες σας λένε. Ας τα αφήσουμε καλύτερα. Γκονσάλης, ε, αρκεί. Εχθές λοιπόν είχαμε ε, τον συνάδελφό σας από το Υπουργείο Παιδείας και χαιρόμαστε πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα κοντά μας. Από ό,τι καταλάβαμε, η Ισπανική Προεδρία έχει κάποιες προτεραιότητες ε, οι οποίες συμπίπτουν με τις δικές μας. Εσείς ε, ακούσαμε επιθυμείτε να προάγετε τον πολιτιστικό τουρισμό, δηλαδή προτίθεστε να ε, στηρίξετε και αυτά που προτείνει η Κομισιόν, ε, την Ευρωπαϊκή Κληρονομιά. Αυτό τα θέλουμε κι εμείς. Και η Κομισιόν τις επόμενες εβδομάδες θα καταθέσει σχετική πρόταση. Επιθυμείτε επίσης να στηρίξετε την ε, επικοδομητική, τον επικοδομητικό κλάδο, ενδιαφέρεστε ιδιαίτερα για το ψηφιακό κινηματογράφο και αυτό μας ενδιαφέρει και εμάς πάρα πολύ. Είδαμε επίσης στο πρόγραμμά σας ότι ε, προβλέπετε να διοργανώσετε και κάποιες ε, σημαντικές συνεδριάσεις και συνέδρια ε, σε σχέση με τον πολιτισμό. Αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Νομίζω λοιπόν ότι έχετε και πολύ ενδιαφέρουσα σταδιοδρομία. Εσείς κύριε Υπουργέ έχετε μεγάλη πειρά από ό,τι μου είπαν σεναριογράφου. Άρα δηλαδή ε, θεωρώ ότι έχουμε εδώ το σωστό άνθρωπο ο οποίος ε, θα μπορέσει να μας ε, ενημερώσει για τους επόμενους πέντε μήνες. Επιτρέψτε μου λοιπόν να σας δώσω το λόγο και προσβλέπω στο να μας πείτε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για, τις, για την ισπανική πολιτική. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, με μεγάλη τιμή σας απευθύνω το λόγο, όχι μόνο ως υπουργό Πολιτισμού της Ισπανικής Κυβέρνησης, αλλά απλώς και μόνο ως πολίτης μιας χώρας που είναι μια νέα δημοκρατία με μεγάλη πολιτιστική παράδειση και είναι και προευρωπαϊκή. Και αυτός είναι ο κύριος στόχος μου. Σας παρουσιάσω τις γενικές γραμμές δράσης της Ισπανικής Προεδρίας ε, σε θέματα πολιτιστικά. Με μεγάλο ενθουσιασμό και με φιλόδοξα σχέδια και με θέληση συνεργασίας μαζί σας αντιμετωπίζουμε την Προεδρία. Μετά από πολύ σοβαρή ανάλυση σχεδιάσαμε την πολιτική μας βάσει κάποιων πολιτικών και πολιτιστικών αρχών. Θέλουμε ο πολιτισμός να βρίσκεται στην καρδιά των προγραμμάτων της Ευρώπης για το μέλλον λαμβάνοντας υπόψη και την οικονομική παγκόσμια κρίση, αλλά και τονίζοντας χρόνο τις δημοκρατικές μας αρχές. Διότι να θεωρήσουμε ότι είναι ο πολιτισμός θέμα προτεραιότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα συνεισφέρει μόνο στην οικονομική ανάπτυξη, δημιουργία θέσεων απασχόλησης, αλλά θα ενισχύσει και τους πολίτες και θα κάνει ακόμη πιο ισχυρό το κοινό ευρωπαϊκό σχέδιο που μας ενώνει. Αυτό είναι το πνεύμα με το οποίο οι τρεις προεδρίες, το Βέλγιο, η Ουγγαρία και εμείς προσπαθούμε να αναπτύξουμε τα σχέδιά μας στα πλαίσια της περίοδου που ζούμε μετά την υπογραφή της συνθήκης της Λισαβόνας. Και βεβαίως αυτό το οποίο μας ενώνει είναι η δημοκρατία, η ειρήνη, ο πολιτισμός και η ευημερία στον ευρωπαϊκό χώρο. Τα επόμενα δέκα χρόνια θα γίνουμε περισσότεροι και θα είμαστε μία ήπειρος της ψηφιακής οικονομίας, της, κοινωνικής ε, ε, συνοχής και της καινοτομίας. Το κλειδί θα είναι η στρατηγική 2020 και η στρατηγική μετά τη Λισαβόνα για να μπορέσουμε να ζήσουμε όλοι καλύτερα από κοινού. Απ' την άλλη είναι πάρα πολύ σημαντικό να εναρμονίσουμε δύο δικαιώματα. Το δικαίωμα που έχουν όλοι οι εργαζόμενοι οι οποίοι αναπτύσσουν δραστηριότητα στον τομέα πολιτισμού να γίνονται σοβαστές οι προσπάθειές τους με το δικαίωμα που έχουν όλοι οι πολίτες να έχουν πρόσβαση σε θέματα πολιτιστικά. Απ' την άλλη, το να συνεισφέρουμε στην ενίσχυση της ε, βιομηχανίας των πολιτιστικών αγαθών που δημιουργεί θέσεις απασχόλησης και οικονομική και κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη είναι επίσης ένα θέμα που αφορά όλους τους πολίτες. Κυρίες και κύριοι, σας είπα ποιες είναι οι αξίες και που μας διέπουν στα πλαίσια της Προεδρίας μας. Σας ανέφερα τις προκλήσεις και τη στρατηγική μας και ενώ τώρα θα σας πω ποιες είναι οι τρεις προτεραιότητες μας στα πλαίσια του πολιτισμού. Πρώτα απ' όλα, να μπορέσουμε να προωθήσουμε τις δυνατότητες που έχει η κουλτούρα στα πλαίσια της ε, περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης. Δεύτερον, να παγιώσουμε τον πολιτισμό σε αν ε, συνιστόσα οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής. Και τρίτον, να αναπτύξουμε και να διαδώσουμε τα πολιτιστικά ψηφιακά περιεχόμενα. Στα πλαίσια των δράσεων αυτών φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η καινοτομία τους ε, ευρωπαϊκής πολιτιστικής ε, σφραγίδας, η ετικέτας αν θέλετε. Αυτό είναι κάτι το οποίο ως πρωτοβουλία άρχισε να ε, προωθείται τον Απρίλιο του 2006 από τους Υπουργούς Πολιτισμού της Γαλλίας και της Ισπανίας. Τι προσπαθούμε να κάνουμε? Να προωθήσουμε μεταξύ των πολιτών της Ευρώπης και κυρίως μεταξύ των νεότερων την κοινή μας ιστορία και τον κοινό μας ε, πολιτισμό. Προσπαθούμε να προωθήσουμε την ευρωπαϊκή ταυτότητα και την συμμετοχή των πολιτών στην οικοδόμηση της Ευρώπης. Και επίσης προσπαθούμε να βελτιώσουμε τις περιοχές μας, να τις κάνουμε πιο ελκυστικές για να προωθήσουμε την αηφόρο ανάπτυξη. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, η Επιτροπή πάρα πολύ σύντομα θα παρουσιάσει την νομοθετική της πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο και πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε επιτυχώς μαζί σας για να προωθηθεί αυτό το θέμα που μας φαίνεται τόσο σημαντικό. Άρα το θέμα αυτό μπορώ να πω ότι θα συζητηθεί στο Συμβούλιο Υπουργών 11 και 12 Μαΐου. Και μπορώ να σας εγγυηθώ ότι η Ισπανική Προεδρία θα κάνει ό,τι μπορεί και το εγγυάται αυτό για να προχωρήσει το πρόγραμμα αυτό. Από... Συγχρόνως με αυτό το θέμα πρέπει να σας πω ότι θα κάνουμε και μία ε, συνάντηση επιρρογνωμόνων στο Κάθερες από 19 έως 21 Απριλίου. Απ' την άλλη, έχουμε θέσει ως στόχο να αναλύσουμε τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για θέματα συνεισφοράς του πολιτισμού σε σχέση με την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη. Θα πρέπει λοιπόν να αναλύσουμε τον ρόλο που διαδραματίζει στις διάφορες ευρωπαϊκές διαθροτικές πολιτικές η κουλτούρα και ιδιαιτέρως στα πλαίσια του ΕΤΠΑ. Δεύτερος άξονας προτεραιότητας στα πλαίσια του πολιτισμού για την Προεδρία μας είναι η παγίωση του πολιτισμού ως συντελεστού οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής. Σιγά σιγά βλέπουμε ότι όλο και περισσότερο αυξάνεται η συνεισφορά των δημιουργικών πολιτιστικών επιχειρήσεων στην οικονομική ανάπτυξη. Πρόκειται για τις περιφερήμες ε, βιομηχανίες ταλέντων που μπορούν με πολύ έξυπνο τρόπο να απορροφήσουν τις ε, αρνητικές επιπτώσεις ε, της οικονομικής κρίσης και να δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης. Γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να προωθηθεί το θέμα αυτό περαιτέρω. Γι' αυτό είναι το θέμα του δεύτερου Ευρωπαϊκού Φόρουμ Οικονομίας και Πολιτισμού που θα οργανωθεί στη Βαρκελόνη 29 με 31 Μαρτίου. Θα ήθελα να σας καλέσουμε να συμμετάσχετε σε αυτό το φόρουμ και με μεγάλη ευχαρίστηση θα σας υπερεχθούμε στη Βαρκελόνη. Η συνάντηση αυτή θα ακολουθηθεί από την άτυπη συνάντηση των Υπουργών Πολιτισμού στην Βαρκελόνη της 31 Μαρτίου για να συζητηθούν αυτές οι βιομηχανίες, οι πολιτιστικές και να συζητηθεί η πράσινη βίβλος σε σχέση με το θέμα αυτό την οποία έχει συντάξει η Κομισιό. Και όλα αυτά τα θέματα θα παρουσιαστούν στις 10 ε, και 11 Μαΐου στην συνάντηση του Συμβουλίου. Εμείς έχουμε αναλάβει επίσης ε, την μελέτη των θεμάτων που αφορούν το πρόγραμμα εργασίας 2008-2010 σε θέματα πολιτιστικά. Στις 25 με επίσης στη Μαδρίτη θα γίνει μία συνάντηση μεταξύ των εκπροσώπων των ε, καλών τεχνών και του κινηματογράφου, όπου θα συζητηθούν ε, θέματα κινητικότητας των καλλιτεχνών. Επίσης, ε, πρέπει να σας πω ότι εκείνο που μας ενδιαφέρει επίσης είναι να ασχοληθούμε στα πλαίσια του τρίτου άξονα με την διάδοση των ε, ψηφιακών πολιτιστικών περιεχομένων. Αυτό είναι κάτι το οποίο αφορά επίσης και την ψηφιακή βιβλιοθήκη Ευρωπαίνα. Πρέπει να σας πω ότι όλα όσα κάνουμε στα πλαίσια αυτών των προγραμμάτων έχει στρατηγική σημασία, διότι ε, θέλουμε να προωθήσουμε την ψηφιοποίηση της πολιτικής μας κληρονομιάς να βοηθηθούμε από την εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών σε όλη την Ευρώπη, όχι μόνο για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις τεχνολογικές αλλαγές, αλλά να μπορέσουμε να έχουμε και ε, ηγετικό ρόλο. Και αυτό είναι το ε, πλαίσιο ενός σεμιταρίου, το οποίο τον Απρίλιο θα γίνει στη Μαδρίτα. Πέρασαν δύο χρόνια από τότε που ε, η Επιτροπή δημοσίευσε την ανακοίνωσή της για θέματα ε, πολιτιστικών και δημιουργηθών περιεχομένων online. Δεν θα πρέπει να σταματήσουμε, δεδομένου ότι τα πράγματα εξελίσσονται πάρα πολύ γρήγορα. Γι' αυτό αυτά τα θέματα θα τα συζητήσουμε στο Συμβούλιο Υπουργών που θα λάβει χώρα, επαναλαμβάνω και πάλι, το Μάιο. Σε σχέση με το μέλλον της Ευρωπαϊκής, της ψηφιακής Ευρωπαϊκής Βιβλιοθήκης, πολύ πιθανώς θα προσπαθήσουμε να υιοθετήσουμε στα πλαίσια του Συμβουλίου κάποια συμπεράσματα, ώστε να μπορέσει η Ευρωπαϊκή να γίνει μια κοινοτική πρωτοβουλία ώστε να μπορέσουν να, γίνουν, να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες ψηφιοποίησης, να έχουμε μεγαλύτερη ε, δημοσιονομική σταθερότητα και να μπορέσουμε να κάνουμε πιο προσβάσιμη την ε, ε, ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε επίσης πολλές προκλήσεις στο θέμα του κινηματογράφου το ψηφιακό, ο ψηφιακός κινηματογράφος είναι μία αλλαγή με τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται τα έργα τα οπτικοακουστικά, με τον τρόπο με τον οποίο παράγονται, διανέμονται και προβάλλονται. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να δούμε με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε να ε, συνοδεύσουμε αυτή τη μεταβατική περίοδο προς την ψηφιοποίηση. Το θέμα λοιπόν είναι να κάνουμε τα πράγματα με τρόπο που δεν θα προκαλέσει αρνητικές επιπτώσεις ε, στον ε, τομέα αυτό, λαμβάνοντας κυρίως υπόψη ότι θα πρέπει να διατηρήσουμε τους μικρούς τους κινηματογράφους που υπάρχουν στις μικρότερες πόλεις. Η Προεδρία μας το θέμα αυτό επίσης θα το συμπεριλάβει στο ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου Υπουργών του Μαΐου. Στον Βαρκελόνη θα κάνουμε στις 5 και 6 Μαρτίου ένα σεμινάριο για τις ψηφιακές ταινίες, ώστε να μπορέσουν οι υπεύθυνοι του τομέα και οι σκηνοθέτες να μας δώσουν τις ιδέες τους για την ψηφιοποίηση του κινηματογράφου στην Ευρώπη. Κυρίες και κύριοι, αυτές, αυτοί είναι οι τρεις γενικοί άξοδες της δράσης μας. Τελειώνοντας, θα ήθελα να τονίσω δύο άλλα θέματα τα οποία δημιουργήθηκαν με την ε, γέννηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δύο θέματα τα οποία θα πρέπει να ασχοληθούμε από κοινού. Πρώτα απ' όλα, να καταπολεμήσουμε την διάκριση. Οι γυναίκες, οι μειονότητες και κάποιες οργανώσεις της χώρας μας θα πρέπει να τύχουν τις υποστήριξής μας ώστε να μπορέσουν όλοι οι πολίτες να έχουν πρόσβαση στην κουλτούρα, στον πολιτισμό. Και δεν εννοώ μόνο να μπορούν να, ε, να υποφελούνται των πολιτιστικών αγαθών μας, αλλά να μπορούν ε, να δημιουργούν επίσης. Γι' αυτό θα πρέπει να μην φυστούμε προσπαθειών και οι προσπάθειες που θα καταβληθούν θα πρέπει να τύχουν τη υποστήριξη όλων των δημοσίων οργών. Επίσης θα ήθελα να, πόσο, να υπογραμμίσω πόσο σημαντική είναι η πολιτιστική μας ε, ε, ποικιλομορφία. Θα πρέπει να προχωρήσουμε ο καθένα τον πολιτισμό του και τη γλώσσα του, ώστε να μπορεί ο κάθε Ευρωπαίος πολίτης να μπορεί να απευθύνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση τη μητρική του γλώσσα. Διότι έτσι υπογραμμίζοντας την πολυπολιτισμικότητά μας, ενισχύουμε τις ρίζες μας, εμπλουτίζουμε ε, την Ευρώπη για τον κοινό δρόμο που την περιμένει στο μέλλον. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε αυτό που μας προτείνεται είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικά μεγάλο έργο. Το θέμα της ψηφίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βλέπω ότι όλοι ζητούν τον λόγο. Ελπίζω να προσέξατε, δεν προφτάνει κανείς να τα γράψει όλα αυτά. Για ε, δω που είναι ο κατάλογος. So. Okay, So, Frau Badia. Η κυρία Μπαδία. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω την Υπουργό για την παρουσίασή της, την εμπεριστατωμένη της συγκεκριμένη και με πολύ ευρωπαϊκά και φιλόδοξα στοιχήματα και προκλήσεις για την ε, Ισπανική Προεδρία όλα τα θέματα που μας αφορούν είναι θέματα τα οποία θίξατε εσείς στα πλαίσια των προτεραιοτήτων της Ισπανικής Προεδρίας. Αλλά θα ήθελα να αναφερθώ στην δεύτερη προτεραιότητα που παρουσιάσατε σε σχέση με τις δημιουργικές ε, βιομηχανίες του κλάδου για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την οικονομική κρίση και να δημιουργήσουμε νέες θέσεις απασχόλησης. Υπό τις παρούσες συνθήκες της οικονομικής κρίσης, το γεγονός ότι θέλουμε να ενισχύσουμε τέτοιου είδους δημιουργικές και πολιτιστικές δραστηριότητες είναι από τα πιο έξυπνα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε σκεφτόμενοι την απασχόληση στην οικονομία και τον πολιτισμό. Έχω κάποια στοιχεία τα οποία δεν είναι ενημερωμένα, διότι δεν βρήκα πιο τελευταία, πρόκειται για στοιχεία του 2006, αλλά ξέρω ούτω ή άλλω ότι τα παρόντα στοιχεία συνηγούν περισσότερο υπέρ αυτών που λέω. Ξέρω ότι το 2006 η πολιτιστική ε, βιομηχανία ήταν ε, αντιπροσώπευε μόνο το 2% του ΑΕΠ και εάν το συγκρίνουμε με την χημεία που ήταν 2,3 και τον ε, τομέα των ειδών διατροφής που είναι το 1,9 μιλούμε για ένα τομέα που έχει πάρα πολύ μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης και οι οικονομικές δυνατότητες και οικονομικές δημιουργίας απασχόλησης πάρα πολύ μεγάλες. Αν ήταν δυνατό λοιπόν θα ήθελα υπουργό να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες για το πώς θα ενισχύσουμε τον τομέα αυτό που είναι τόσο σημαντικός για το μέλλον της Ισπανίας, χώρας μας, αλλά και όλης της Ευρώπης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κυρία. Δεν ανήκουμε στο ίδιο πολιτικό κόμμα, αλλά ξέρετε πόσο εκτιμώ και εσάς και αυτά τα οποία κάνετε για τον πολιτισμό. Όπως ε, είπε η Πρόεδρος, είναι αυτή η πολιτιστική ετικέτα που θέλουμε να βάλουμε, πολύ σημαντική για την πολιτιστική ε, κληρονομιά της αγαπημένης μας γυρεάς Ευρώπης. Κυρίως σε σχέση με τον τουρισμό. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά η Υπουργός ότι στην Ισπανία η περιοχή η οποία αντιστάθηκε περισσότερο στην οικονομική κρίση είναι η Μαδρίτη, που δεν έχει ούτε παραλίες, ούτε άλλα πράγματα που έχουν οι τυπικά τουριστικές περιοχές, αλλά σε θέματα πολιτισμού είναι το νούμερο ένα. Και βεβαίως ξέρουμε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο απαιτεί και μεγάλες οικονομικές θυσίες ε, από τα ε, υπουργεία που ασχολούνται με την αποκατάσταση μνημείων και με την πρόθεση των πολιτιστικών ε, ε, στοιχείων της Μαδρίτης και της περιοχής που είναι τόσο πλούσια. Θα πρέπει λοιπόν να μας πείτε αυτή η πολιτιστική ετικέτα, αυτή η πολιτιστική σφραγίδα αν θέλετε, πώς δίνεται στις διάφορες περιοχές. Καταρχήν πρέπει να δημιουργηθεί αυτό το πρόβλημα. Κύριε Κώστα. Saluto naturalmente la ministra θα ήθελα να καλωσορίσω βέβαια και την Υπουργό Πολιτισμού της Ισπανίας και την ευχαριστώ πάρα πολύ για το ότι μας παρουσίασε αυτό το στρατηγικό σχέδιο με απόλυτη σαφήνεια και με στόχους τους οποίους εκτιμώ ιδιαίτερα. Από ό,τι άκουσα, εσείς ε, επικεντρώσατε τη και επικεντρώνετε τη στρατηγική σας σε τρεις άξονες. Ε, νομίζω αυτοί οι άξονες ε, και πολλά σημεία αυτών υπάρχουν και στη δική μας την ημερήσια διάταξη και τα θεωρούμε και εμείς όλα αυτά σημαντικά. Πρώτη ερώτηση. Όσον αφορά την ε, προώθηση του τουρισμού, του πολιτιστικού τουρισμού και της ε, πολιτιστικής ε, κληρονομιάς. Υπάρχει ως Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε μεγαλύτερη αρμοδιότητα για θέματα τουρισμού. Ε, τη συμμεριζόμαστε βέβαια αυτή την αρμοδιότητα και ε, με την Επιτροπή έχουμε επιτρόπους ε, οι οποίοι είναι, έχουν και επικάλυψη αρμοδιοτήτων όσον αφορά τον τουρισμό. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξή. Όσον αφορά το θέμα της, του να μπορούμε να υιοθετήσουμε ένα πρόγραμμα, το οποίο συζητήθηκε στο Συμβούλιο της ε, Ευρώπης, ε, πέρα από το Σαντιάγκο. Έχουμε και άλλες ε, πολιτιστικές διαδρομές, οι οποίες κατά την άποψή μου θα μπορούσαν να αποτελούν μια πραγματική ευρωπαϊκή στρατηγική, όπου θα διασταυρώνονται η ανάπτυξη του τουρισμού, η ευρωπαϊκή, το ευρωπαϊκό σήμα και θα διασταυρώνονται και τα κονδύλια γιατί ξέρετε, νομίζω ότι και το Κοινωνικό Ταμείο της Ευρώπης, τουλάχιστον αυτή την εμπειρία έχω κάνει εγώ σε δική μου την περιοχή, ε, μέσα από το Ταμείο αυτό προωθούνται όλες ε, οι δραστηριότητες ε, και ο πολιτισμός και οι βιομηχανικές δραστηριότητες. Άρα δηλαδή πρέπει να συνεργαστούμε σε μεγάλο βαθμό με το Κοινωνικό Ταμείο και αυτό θεωρώ ότι είναι ένας πολύ καινοτόμος άξονας. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω από την Ισπανική Προεδρία να αρχίσει να σκέπτεται το κατά πόσον πράγματι τα πολιτιστικά αγαθά μπορούν να ενταχθούν σε ένα πρόγραμμα που να το εγκρίνει και το Συμβούλιο της Ευρώπης. Δεύτερο σημείο, όσον αφορά το θέμα της ε, ψηφιοποίησης. Μιλήσατε για την ε, ε, ψηφιοποίηση σε σχέση με τα πολιτιστικά αγαθά και τον πολιτιστικό κλάδα γενικότερα. Εγώ αναφέρομαι στις κινηματογραφικές αίθουσες. Θα ήθελα να πω λοιπόν ότι σε ορισμένε χώρες όπως και στην Ιταλία υπάρχει κάποια εξαίρεση μόνο για ένα χρόνο βέβαια για να μπορούν οι κυβερνήσεις ε, να προχωρήσουν στην ψηφιοποίηση των κινηματογραφικών αιθουσών. Αυτό που αναφέρετε κι εσείς. Αυτή τη στιγμή υπάρχει βέβαια μια εξαίρεση που όπως σας είπα όμως έχει χρονικό περιορισμό. Και ε, κατ' ουσίαν κατά την άποψή μου πρόκειται για ένα στρατηγικό στόχο για να μπορεί κανείς να εκμεταλλευτεί καλύτερα την πολιτιστική κληρονομιά, να είναι πιο ανταγωνιστικό το ευρωπαϊκό σύστημα και όσον αφορά την ε, διανομή αλλά και τον πραγματικό κινηματογράφο. Άρα δηλαδή θεωρώ ότι και αυτό είναι ένα θέμα ε, που θα μπορούσε να αποτελεί στόχο σας και σωστά ε, το αναφέρατε και το συσχετίσατε με, τις, τα πολιτιστικά αγαθά. Ο κύριος Παπα-Νικολάου παρακαλώ. Καλή επιτυχία κυρία Υπουργέ. Ευχαριστούμε πράγματι για την παρουσίαση. Το πρόγραμμα είναι φιλόδοξο και ελπίζουμε τα αποτελέσματα να είναι και ανάλογα. Θέλω να σας κάνω ένα συγκεκριμένο ερώτημα για ένα ζήτημα που ενδεχομένως δεν γνωρίζετε και το αντιλαμβάνομαι. Θα ήθελα όμως να το θέσω υπόψη σας. Στην ε, στον τελευταίο προϋπολογισμό, όπως ψηφίστηκε από το Κοινοβούλιο μας, ε, υπήρξε, ε, προβλεφ, υπήρξε πρόβλεψη για διάταξη η οποία ξεκίνησε από την Επιτροπή μας σε σχέση με τη δημιουργία ενός πιλωτικού προγράμματος ε, για την δημιουργία ενός δικτύου για την ανέβρεση κλεμμένων έργων τέχνης, την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και βεβαίως την δημιουργία και την ανάπτυξη δράσεων για την καταπολέμηση Τη αρχαιοκαπηλεία και όχι μόνο. Και βεβαίως αυτό στοχεύει και στην προστασία της πολιτισμικής κληρονομιάς και την αντιμετώπιση ενός σύγχρονου φαινομένου που πραγματικά μαστίζει τις κοινωνίες μας σε σχέση με το εμπόριο των κλεμμένων έργων τέχνης. Ε, αφενός θέλω να, το θέσω σε γνώση σας, αφετέρου θα ήθελα την άποψή σα αν συμφωνείτε με αυτό και αν σκοπεύετε να προωθήσετε αυτή την προσπάθεια. Vielen Dank. Frau Minister, die ersten vier Fragen bitte. Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, μπορείτε να απαντήσετε αυτές τις ερωτήσεις. Bien, eh, muchas gracias, eh, señorías, muchas gracias, eh, señora Badía. Σας ευχαριστώ κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ την κυρία Μπαδία, την κυρία Κώστα, τον κύριο Φίσες και τον κύριο Παπα-Νικολάου. Όντως, η πολιτιστική βιομηχανία είναι σημαντικές. Είναι ανα... Είναι αδιάψευτα τα στοιχεία που έχουμε και βλέπουμε ότι μπορεί η Ευρώπη να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο, όχι μόνο παρουσιάζοντας ιδέες, αλλά και να δημιουργήσει με σταθερό τρόπο πλούτο, θέσεις απασχόλησης. Η σημασία του πολιτισμού σε σχέση με το ε, και τα ποσοστά που ανέφερε η κυρία Μπαντία, όντως αποδεικνύουν ότι υπάρχουν πολλές δυνατότητες ανάπτυξης. Και βεβαίως αυτό το οποίο θέλουμε είναι να διασφαλίσουμε την ανάπτυξη του πολιτισμού, την διαφοροποίηση και τη στιγμή που αλλάζει το οικονομικό πρότυπο στις κοινωνίες μας, αυτό το θέμα θα πρέπει να το εξετάσουμε με μεγάλη προσοχή. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό στα πλαίσια της ε, Προεδρίας μας να προτείνουμε και να μελετήσουμε διεξοδικά και, διεξοδικά, και αυτό είναι κάτι που θα το, θα το συζητήσουμε την επόμενη εβδομάδα στη Σαραγώσα, πώς η τοπική και η περιφερειακή οικονομία και η ανάπτυξή τους μπορεί να βοηθήσουν για την ανάπτυξη αυτών των πολιτιστικών διαδρομών που ανέφερε η κυρία Κώστα και πώς μπορούμε να κάνουμε μία, ένα συσχετισμό μεταξύ οικονομίας, πολιτισμού και άλλων. Ακριβώς όπως είπε και ο κύριος Φίσας, εμείς στην Ισπανία γνωρίζουμε πάρα πολύ πόσο καλά μπορεί να λειτουργήσει το σύστημα αυτό σεβόμενοι και τις διάφορες ε, γλωσσικές και πολιτιστικές ε, διαφορές και διαφοροποιήσεις που έχουμε στην Ισπανία. Τώρα, σε θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς. Είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στην Ισπανία. Ξέρουμε και σεβόμεθα απόλυτα την παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά την οποία έχει θεσπίσει η UNESCO και πάντα κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να προωθήσουμε πρωτοβουλίες που πάνε προς αυτή την κατεύθυνση. Προστασία της πολιτιστικής μας ε, κληρονομιάς και συγχρόνως καινοτομία όσον αφορά τις ε, τεχνικές ε, διατήρησης και αποκατάστασης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα συζητηθεί στην συνάντηση εμπειρογνωμόνων που θα γίνει στο Κάθερες, καθώς και στα πλαίσια των άλλων πολιτιστικών προτεραιοτήτων που αναλαμβάνουμε. Και αυτό εξάλλου είναι κάτι το οποίο απασχολεί το Υπουργείο Πολιτισμού, όχι τώρα μόνο στα έξι μήνες της Ισπανικής Προεδρίας, αλλά γενικότερα. Τώρα, όσον αφορά την ψηφιοποίηση των κινηματογραφικών αίθουσων, συμφωνώ με την κυρία Κώστα ότι το θέμα αυτό έχει μεγάλη σχέση με τις δυνατότητες διάδοσης του ευρωπαϊκού κινηματογράφου, που στις ε, χώρες μας έχει σχέση με την διανομή κάποιων κινηματογραφικών έργων. Αυτό λοιπόν ψηφιοποιημένων. Ξέρουμε λοιπόν ότι κάποιες χώρες ήδη το θέμα αυτό το αντιμετωπίζουν με διαφορετικό τρόπο, αλλά εμείς πιστεύουμε ότι θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί με το θέμα αυτό, να το συζητήσουμε πολύ προσεκτικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να υιοθετήσουμε τα μέτρα που θα μας επιτρέψουν να προχωρήσουμε και να μην δημιουργήσουμε αυτό το δίκτυο ψηφιοποιημένων αιθουσών. Χωρίς συγχρόνως να αποκλείσουμε και τους μικρούς κινηματογράφους των μικρών πόλεων που έχουν ε, λιγότερους θεατές αν θέλετε, αλλά θα πρέπει και αυτόν τα συμφέροντα να σεβαστούμε. Τώρα, όσον αφορά την... Ε, αυτά τα οποία ανέφερε για την αρχαιοκαπηλεία ο κύριος ε, Παπανικολάου, τα έργα τα οποία έχουν κλαπεί Εδώ είναι και θέμα εθνικής νομοθεσίας τη κάθε χώρας και είμαστε περισσότερο σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργών Εσωτερικών κάθε χώρας. Είναι όμως σημαντικό το θέμα και οποιαδήποτε ε, συνεργασία μπορούμε να προσφέρουμε στις αρχές, της δικαστικές ή στις αστυνομικές για την εξέβρεση ε, αρχαιοτήτων που έχουν κλαπεί είναι σημαντική οποιαδήποτε συνεργασία, επαναλαμβάνω. Πιστεύω ότι έχω απαντήσει σε ερωτήσεις σας. Ο Αντιπρόεδρος κύριος Μπίσκι έχει το λόγο. Κύριε Υπουργέ, ε, το βρίσκω πάρα πολύ ευχάριστο το ότι τον πολιτιστικό τομέα ε, τον θεωρείται προτεραιότητα. Και χαίρομαι πάρα πολύ που ο κινηματογράφος είναι σημαντικός για σας. Ο κινηματογράφος σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες βρίσκεται σε ιδιαίτερα ανησυχητική κατάσταση, τουλάχιστον στη δική μου τη χώρα. Κινηματογράφος είναι όμως κομμάτι του πολιτισμού. Ο κινηματογράφος ε, έχει σχέση με τις ε, μικρές ε, πόλεις, όπου δυστυχώς πολλές φορές δεν υπάρχει καν εκεί, έχει εξαφανιστεί από εκεί, από τις μικρές πόλεις. Τώρα, το να περάσουμε στην ε, ψηφιοποίηση του κινηματογράφου, αυτό θα μπορούσε ίσως να μας επιτρέψει να ασχοληθούμε περισσότερο με τον κινηματογράφο. Εγώ θέλω να προβάλλουμε περισσότερο τον ευρωπαϊκό, αλλά δεν σημαίνει ότι πρέπει να παραμελήσουμε άλλες μορφές κινηματογράφου. Κάναμε πολύ καλή εμπειρία ο ευρωπαϊκός ε, κινηματογράφος ε, σε διάφορα φεστιβάλ στην Ανατολική Γερμανία, στο Κότμπους, παραδείγματος χάρη, υπάρχει φεστιβάλ ε, ανατολικοευρωπαϊκών ταινιών. Πολύ καλό αυτό. Ε, ίσως, ε, λοιπόν, το, τις ευρωπαϊκές ε, ταινίες και τις μεγάλες ισπανικές ταινίες μπορείτε να τις προβάλετε περισσότερο, έτσι ώστε να έχουν και περισσότερους θεατές. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι τα ταλέντα που υπάρχουν σε αυτόν τον τομέα στην Ευρώπη πρέπει να τα στηρίξουμε περισσότερο. Δεν καταλαβαίνω γιατί μέχρι σήμερα δεν υπάρχει κανένας χώρος εκπαίδευσης κινηματογραφιστών, όπου ταλέντα από διάφορες χώρες να συναντιόνται και από κοινού να μαθαίνουν κινηματογράφο. Αν αυτό μάλιστα ήταν υπό την αιγίδα των μεγάλων σκηνοθετών, αυτό θα ήταν καταπληκτικό. Ε, εντάξει, ανταλλαγή, καλή ανταλλαγή, αλλά ίσως πιο έντονη ανταλλαγή και ίσως και το θάρρος να συστήσουμε μια μονάδα κινηματογραφιστών υψηλού επίπεδου. Αυτό ε, θα έπαιζε σημαντικό ρόλο στις, στα οπτικοακουστικά μέσα στην Ευρώπη. Η κυρία Τρούπελ έχει το λόγο, η αντιπρόεδρος. Χαίρομαι πάρα πολύ που αυτό το θέμα του ψηφιακού κινηματογράφου το θεωρείτε προτεραιότητά σας. Και εδώ θέλω να επισημάνω με αυτή την ευκαιρία ότι την Πέμπτη εδώ στο Κοινοβούλιο ε, θα έχουμε συνέδριο με Ευρωπαίους κινηματογραφιστές. Ίσως αυτό να ενδιαφέρει ε, τους συναδέλφους. Πέμπτη, 9 ώρα το πρωί θα ξεκινήσει. Και αν είμαι καλά, στην υγεία μου θα μιλήσω και εγώ και ο κύριος ε, Σάμπο, ο Ούγγρος ε, σκηνοθέτης. Εγώ έκανα μια έκθεση για το θέμα αυτό και χαίρομαι πάρα πολύ που κι εσείς ε, αναγνωρίζετε ότι το πρόγραμμα «Ο Ευρωπαϊκά είναι σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, ε, είπατε ότι πρέπει να υπάρχει ε, μεγαλύτερη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Και γι' αυτό θεωρώ ότι όταν θα συνταχθεί ε, η συνταχθούν οι επόμενε δημοσιονομικέ πρακτικέ και θα γίνει και κουβέντα για τι συνθήκε Λισαβόνα. Θα ήταν καλό αν στο Συμβούλιο γίνει κατανοητό ότι ένα τμήμα των κονδυλίων τη στρατηγική Λισαβόνα θα πρέπει να διοχετευθούν στην Ευρωπαϊκή και στην ψηφιοποίηση γιατί ε, θεωρώ ότι αν θέλει να προχωρήσει η Ευρώπη, αυτό είναι καθοριστικό τμήμα η ψηφιοποίηση. Επίσης, επειδή πολλοί από εμάς ε, ψάχνουν να βρουν ε, ποια είναι η σωστή σχέση ανάμεσα στην εύκολη πρόσβαση στο διαδίκτυο, και εσείς το είπατε ότι αυτό είναι στόχος σας, και αφετέρου τη σωστή προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων. Μάλιστα, ανακοινώσατε ότι θα γίνουν και συνέδρια για αυτό το θέμα. Μήπως μπορείτε ήδη σήμερα να μας πείτε τι θα γίνει τελικά με αυτά τα θέματα ο κύριος Μπορίς. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ, όπως και οι άλλοι συνάδελφοι, καταρχήν να σας συγχαρώ και να σας ευχαριστήσω για την παρουσίασή σας και για την σημασία που δίδεται στον κινηματογράφο και στην ψυχιοποίησή του. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η δυνατότητα διάθεση κινηματογραφικών ταινιών σε όλη την Ευρώπη, γιατί έτσι μπορούμε να κατανοήσουν οι πολίτες καλύτερα την Ευρώπη, όταν γνωρίζουν ότι υπάρχει ευρωπαϊκός κινηματογράφο Εγώ θα ήθελα να σας πω, ρωτήσω, όταν είσαστε εσείς πρόεδρος τώρα του Συμβουλίου Υπουργών Πολιτισμού, θα προβλέψετε ίσως ένα χρονοδιάγραμμα για τη μεσηφιοποίηση. Γιατί σε άλλες χώρες, στις διάφορες χώρες, συγγνώμη, υπάρχει διαφοροποίηση του ποσοστού ε, βελτίωση προς την κατεύθυνση αυτή. Εσείς λοιπόν θα έχετε ένα χρονοδιάγραμμα για να διευκρίνετε την δυνατότητα πρόσβασιμότητας στις ψηφιακές αυτές ταινίες. Και επίσης, ε, τι έχετε να πείτε για την χρηματοδότηση του κινηματογράφου. Αυτό συχνά συμπίπτει με τη χρηματοδότηση ευρωπαϊκών ταινιών. Ξέρω στη Γαλλία, στην Ισπανία υποστηρίζετε τους νέους ε, σκηνοθέτες. Προβλέπετε κάτι σε ευρωπαϊκό επίπεδο προς την αυτή κατεύθυνση, την υποστήριξη δηλαδή νέων σκηνοθετών, νεαρών σκηνοθετών. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ. Άκουσα με μεγάλο ενδιαφέρον την παρουσίαση των προτεραιοτήτων σας. Κυρίως όταν τονίσετε ότι είναι απαραίτητο να μπορέσει η γλωσσική και πολιτισμική διαφορετικότητα να υποστηριχθεί και η τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη. Επίσης, τα θέματα ε, δικαιωμάτων που αναφέρατε είπατε ότι είμαστε σε ένα ειδικό τομέα σε θέματα ε, πολιτιστικά και μιλήσατε για το δικαίωμα της προσβασιμότητας και της δημιουργικότητας. Πρόκειται για ένα βασικό δικαίωμα, για ένα θέμα θεμελιώδες, το οποίο βρίσκεται και στο ε, κέντρο του προγράμματος Ευρωπαίνα. Ποια είναι η άποψή σας για αυτό το θέμα, κάτι άλλο που θα ήθελα να αναφέρω. Είναι ότι ο τομέας ο πολιτιστικός είναι ένας τομέας ο οποίος είναι πάρα πολύ ελκυστικός για θέματα που αφορούν τη δημιουργία επιχειρήσεων, ενώσεων και ξέρω ότι γίνονται πάρα πολλά πράγματα σε αυτό το τομέα στην Ισπανία. Και σε θέματα κοινωνικής οικονομίας πάρα πολλά θέματα, πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν ε, έχοντας ως βάση τον πολιτισμό. Τι μπορείτε να μας πείτε για την ανάπτυξη των διαφόρων ε, περιφερειών και τοπικών κοινωνιών σε σχέση με αυτό το θέμα που αναφέρατε. Σας ευχαριστώ. Κυρία Υπουργέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ για τις παρατηρήσεις σας, κυρίες και κύριοι, βουλευτές. Για μας όλα τα θέματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή καθώς και η ψηφιοποίηση και τα δικαιώματα είναι πάρα πολύ σημαντικά και άπτονται όλα των θεμάτων των πολιτιστικών. Θα ήθελα να υπενθυμίσω κάτι το οποίο τόνισε ο Πρωθυπουργό στο Πατέρο. Δηλαδή, ότι ο πολιτισμός συνεισφέρει πάρα πολύ στην ανάπτυξη των κοινωνιών μας, όπως και οι νέες τεχνολογίες. Και βεβαίως θα πρέπει, εφόσον όλο και περισσότερο προχωρούμε προς τη δημιουργία μιας ε, ψηφιοποιημένης ε, κοινωνίας, να δώσουμε και περιεχόμενα σε όλα αυτά τα θέματα στον τομέα των του πολιτισμού. Πιστεύω λοιπόν ότι ως Ευρωπαίοι και σε σχέση με τις ε, γιγαντιές ε, επιχειρήσεις τύπου Google θα πρέπει κάτι να κάνουμε. Και εδώ θα αναφερθώ ιδιαίτερα στην Ευρωπαϊκή. Ξέρουμε βεβαίως ότι τα πολιτιστικά θέματα είναι θέματα τα οποία είναι πολύπλοκα και άπτονται των αρμοδιοτήτων ε, κάθε κράτους σε διαφορετικά επίπεδα. Όπως είπε και η κυρία Βερζά πρόκειται για νέες δυνατότητες, για νέες μορφές δημιουργίας και για νέες μορφές πρόσβασης. Θα πρέπει λοιπόν το θέμα αυτό να το μελετήσουμε διεξοδικά. Και πρέπει να πω ότι όσε φορέ αντάλλαξα απόψε με του συναδέλφου υπουργού για τέτοιου θέματα, το θέμα αυτό μα απασχολεί και προσπαθούμε να βρούμε τον πιο κατάλληλο τρόπο για να αντιμετωπίσουμε τις αλλαγές αυτές, οι οποίες έχουν πάρα πολλές θετικές προκλήσεις, αλλά συγχρόνως μας οδηγεί πολλές φορές σε πρωτόγνωρους δρόμους τους οποίους πρέπει να ακολουθήσουμε και αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν και διάφορα ερωτηματικά στα οποία πρέπει να απαντήσουμε. Θα πρέπει λοιπόν κατά κάποιο τρόπο να υιοθετήσουμε μία κοινή βάση εργασίας, κάποια κοινά κριτήρια που θα ακολουθήσουμε από κοινού για να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό. Είμαστε σε συνεργασία με την Κομισιό, με τα κράτη-μέλη επίσης για να βρούμε την πραγματική φόρμουλα που θα μας οδηγήσει σε συμβατότητα των δικαιωμάτων όλων. Συγχρόνως θέλουμε το ψηφιακό περιεχόμενο, τα περιεχόμενα online των πολιτιστικών ε, δραστηριοτήτων να τα αναπτύξουμε ακόμη περισσότερα. Ίσως θα έπρεπε να δημιουργήσουμε μία επιτροπή σοφών ad hoc που θα μας βοηθήσουν και θα μας επιτρέψουν να προχωρήσουμε στην επίλυση προβλημάτων που είναι πολύπλοκα και απασχολούν σε κάθε χώρα διαφορετικούς υπεύθυνους οργανισμούς. Αυτό για να έχουμε μία συνεκτική θεώρηση όσον αφορά την ε, προστασία τη πολιτιστικής μας κληρονομιάς και την ε, διασφάλισή της. Σε θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ευρώπη έχουμε ηγετικό ρόλο. Και θα πρέπει σε τέτοιου είδους θέματα πολιτιστικά να μπορέσουμε ως Ευρωπαίοι να προχωρήσουμε και ενωμένοι. Διότι αυτό είναι ένα στοιχείο της ευρωπαϊκής μας ταυτότητας. Θα πρέπει να προστατεύσουμε την διαφορετικότητά μας, αλλά να προχωρούμε και προσεκτικά και με συνέχεια. Λαμβάνοντας υπόψη ότι βρισκόμαστε σε κοινωνίες που αλλάζουν με ταχύτητα και οι τεχνολογίες αλλάζουν με μεγάλη ταχύτητα. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα μπορέσουμε να νομοθετούμε, πώς, θα πρέπει, πώς μπορούμε να νομοθετούμε και σωστά, ώστε να διασφαλίσουμε αυτή την πολιτιστική κληρονομιά. Θα πρέπει λοιπόν να αναλύσουμε τα θέματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε ώστε να μπορέσουμε να συνεργαστούμε για να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα προβλήματα συνεργαζόμενοι και με πιο συντονισμένο τρόπο. Διότι μέχρι τώρα ο καθένας προσπαθεί τον πολιτισμό, την κουλτούρα του να τον ε, διαδώσει και να τον διασφαλίσει κατά κάποιο τρόπο με διαφορετικό τρόπο. Θα πρέπει λοιπόν κάτι να κάνουμε από κοινού για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε με συνεκτικό τρόπο. Σα ε, <laughs> euh, σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ κύριε Υπουργέ για την παρουσίασή σας που ήταν τόσο ενδιαφέρουσα. Θα ήθελα να αναφερθώ στην ψηφιοποίηση των ταινών κειμενογράφου. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποιες μικρές αίθουσες που συμβάλλουν πάρα πολύ στην ενδυνάμωση της ε, ευρωπαϊκής πολιτιστικής ταυτότητας. Ο κίνδυνος της ψηφοποίησης των ταινιών ε, που δείχνουν τις θέσεις αυτές, όπως το είδαμε και στη Βαρσοβία, τελευταία στην εκδήλωση αυτή, υπάρχει, έχει δύο προβλήματα. Καταρχήν, το πάρα πολύ σημαντικό κόστος για την ψηφιακή ε, προβολή στις αίθουσες αυτές. Και αναρωτιέμαι πως υπάρχουν κάποιοι πόροι που θα μπορούσαν να χορηγηθούν. Συμφωνείτε εσείς ότι θα μπορούσαμε να συμβάλλουμε στην ε, χρηματοδότηση αυτή της ψηφής των μικρών αυτών αιθουσών κινηματογράφου. Δεύτερον, το πρόβλημα είναι η επιλογή του στάνταρ που θα επιλογεί, του προτύπου που θα ε, χρηθεί. Δεν ξέρουμε ακόμα ποιο θα είναι το πρότυπο που θα ακολουθεί, γιατί υπάρχουν διαφόρων τύπων στάνταρ και θα κάνετε εσείς κάτι για να επιταχύνετε τον ορισμό του προτύπου που θα επιλεχθεί για να μην γίνουν σοβαρές επενδύσεις που θα καταστούν χωρίς αντικείμενο εάν τελικά δεν είναι αυτό το σύστημα που θα γενικοποιηθεί. Θα σας ευχαριστώ κύριε Χανίμπαλ. Thank you, And uh, welcome. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και θα ήθελα να χαιρετήσω την παρουσία της Υπουργού εδώ μεταξύ μας θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια από τα σχόλια που έλεγχαν για την ε, πολιτιστική βιομηχανία, όπως είπε η κυρία Μπαντία στην αρχή της συζήτησης. Εγώ προέρχομαι από το Λονδίνο, που έχουμε ένα τεράστιο τομέα στο, το, της ε, πολιτιστικής βιομηχανίας, ένας από τους κύριους τομείς ε, της οικονομίας της πόλης. Και αυτό χαίρομαι που είπατε ότι θα υπάρχει μια επιτροπή ad hoc για να δει εξετάσει τα διάφορα θέματα που, θέματα που θίγουμε σήμερα. Αλλά εγώ θα ήθελα να μου πείτε κάτι όσον αφορά τα δικαιώματα των εργαζομένων στον τομέα του πολιτισμού και κατά πόσο θέλετε ίσως να το εναρμονίσετε αυτό με τα δικαιώματα της ε, πρόσβασης στο πολιτισμό των ε, πολιτών γενικά. Γιατί ξέρετε ότι υπάρχει πολύ έντονος κατακαιρματισμός στον τομέα και γι' αυτό οι εργαζόμενοι έχουν πολλά προβλήματα. Έχετε δίκιο να θίγετε το θέμα. Θα ήθελα όμως να μου δώσετε κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς διαβλέπετε η Ισπανική Προεδρία να προωθήσει το θέμα αυτό και πώς θα συνεργαστείτε και στα πλαίσια των προσδοκιών σας, ότι όλοι δηλαδή οι πολίτες θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα πρόσβαση στον πολιτισμό. Η κυρία Παλαδέλη. Ευχαριστώ και πάλι κυρία Πρόεδρε. Ε, χαίρομαι ιδιαίτερα αγαπητή κυρία Υπουργέ ότι η Ισπανική Προεδρία έθεσε σε τόσο υψηλό επίπεδο, σε τόσο μεγάλη σπουδαιότητα δύο πολύ σημαντικά αντικείμενα με τα οποία ασχολείται η Επιτροπή μας και με την παιδεία και με τον πολιτισμό. Βέβαια η έννοια πολιτισμός είναι ένας τεράστιος, ε, έχει ένα τεράστιο εύρος, είναι μια πολύ μεγάλη έννοια Φαντάζομαι ότι περισσότερο σας ενδιαφέρει ο σύγχρονος πολιτισμός και το σέβομαι παρόλο που προέρχομαι από μια χώρα με μάλλον περισσότερο αρχαίο ε, πολιτισμό. Ε, η ερώτηση πρώτη είναι αν σκοπεύετε να υποστηρίξετε την ε, διατήρηση, the preservation των αρχαίων μνημείων της Ευρώπης, ένα, αν έχετε κάποια άποψη για αυτό τον τομέα και ε, να, να, να επενέσω πραγματικά το ενδιαφέρον σας για την ε, Ευρωπαϊκή που είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία αυτής της Επιτροπής και μια ερώτηση που ε, πώς θα μπορούσαμε ενδεχόμενα ως, ε, που αφορά στα films πώς εκτιμάτε ότι θα μπορούσαν τα ηλεκτρονικά μέσα και κυρίως η τηλεόραση η οποία κατακλείζεται η ευρωπαϊκή τηλεόραση η οποία κατακλείζεται από πάρα πολύ φτηνής ποιότητας ε, αμερικανικά ε, προγράμματα να αντισταθεί μέσα από αυτήν την ψηφιοποίηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Θα υποβάλω και εγώ μια ερώτηση, κύριε Υπουργέ. Προηγουμένως απαντώντας ε, σε κάποια ερώτηση αναφερθήκατε στις εξωτερικές σχέσεις. Κατά διάρκεια της δικής σας ε, προεδρίας θα ιδρυθεί, θα εγκαθιδρυθεί μάλλον η εξωτερική, το σύστημα εξωτερικών υπηρεσίας ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελπίζω αυτό το όλο σύστημα να μην είναι μόνο διπλωματικό, ή υπέρ των οικονομικών σχέσεων, αλλά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την υπηρεσία εξωτερικών σχέσεων για την προώθηση του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Θα μπορούσατε να συμφωνήσετε ότι ακριβώς η Ισπανία μαζί με τις άλλες κυβερνήσεις βέβαια, θα μπορούσε να βοηθήσει ούτε ώστε να υπάρξει κατανόηση στην Κομισιόν και στη νέα υπεύθυνη την κυρία Άστον για τα θέματα αυτά γιατί νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Μας ενδιαφέρει όλους. Αυτός είναι ο μεγάλος θησαυρό που έχουμε και θα πρέπει να προωθήσουμε αυτή την την ευρωπαϊκή εικόνα σε όλο τον κόσμο. Οι Αμερικανοί μα έστειλαν τις του του εικόνες. Εμείς δεν έχουμε κάνει κάτι παρόμοιο. Θα ήταν πάρα πολύ γνώμη μπορούσατε να μα βοηθούσατε λοιπόν κατά τη διάρκεια τη Προεδρία σα. Και ακριβώ αυτή είναι η χρονική στιγμή κατά την οποία θα υπάρχουν οι πρωτοβουλίε. Υποβλήθηκαν όλε οι ερωτήσει, Κύριε Υπουργέ, μία λίγες απαντήσεις ακόμα και μετά θα μπορέσουμε να τελειώσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, ήταν εξαιρετική η τελευταία σας ερώτηση. Όντως, είναι η πολιτιστική μας κληρονομιά ο θησαυρό μας. Και νομίζω ότι η φωτογραφία αυτή όλων είναι, από κοινού είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να εξάγουμε προς τον, ε, και να δείξουμε προς τον υπόλοιπο κόσμο. Συμφωνώ ότι στο πλαίσιο του δυνατού θα πρέπει να συνεργαστούμε με την κυρία Άστον ότι στα πλαίσια της εξωτερικής ευρωπαϊκής πολιτικής να υπάρχει και λίγος χώρος για τον πολιτισμό, πράγμα που είναι και εξαιρετικό σύμμαχος της διπλωματίας ο πολιτισμός. Και Νομίζω ότι οι φίλοι μας οι Αμερικανοί πάντα ήξεραν πάρα πολύ καλά και να προάγουν και να εξάγουν πολύ καλά την ε, ε, κουλτούρα τους και τον πολιτισμό τους. Όντως, όπως είπε και κάποια συναδελφό σας, οι Ευρωπαίοι βλέπουμε ότι στην μεγάλη και στη μικρή μας οθόνη πολύ συχνά προβάλλονται οπτικοακουστικά προϊόντα που δεν προέρχονται από τις χώρες μας. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε από κοινού να καταβάλουμε προσπάθεια όχι μόνο στον κινηματογράφο ε, που θέλουμε να προωθήσουμε τον ευρωπαϊκό, αλλά και την κινηματογραφική παραγωγή άλλων ε, υπήρων και χωρών όπως ε, τον κινηματογράφο από την Ασία ή από άλλα μέρη του κόσμου που έχουν να προβάλλουν ε, πολύ καλές ταινίες και αυτό είναι όντως ένας από τους θησαυρούς μας. Στην Ισπανία, για να καθισκάσω την κυρία Παλιαδέλη, θα πω ότι εγώ έχω σπουδάσει κλασική φιλολογία. Η αρχαιότητα λοιπόν είναι κάτι το οποίο το έχω μελετήσει πάρα πολύ καλά. Και το αγαπώ το θέμα. Αυτό μου είναι ιδιαίτερα προσφυλές, όχι μόνο γιατί το έχω σπουδάσει. Η αρχαιολογία είναι κάτι που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και στην ε, Ισπανία. και στην Καρθαγένη κατά τη διάρκεια της Προεδρίας θα κάνουμε ένα ε, σεμινάριο για την υποθαλάσσια αρχαιολογία και νομίζω ότι το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα πρέπει να το σκεφτούν όλοι οι Ευρωπαίοι, διότι όλοι οι Ευρωπαίοι έχουμε ένα παρελθόν. Και μεγάλοι θησαυροί βρίσκονται στις θάλασσές μας και με τη βοήθεια της τεχνολογίας σήμερα μπορούμε να κάνουμε στον τομέα αυτό έρευνες και να μπορέσουμε να σταματήσουμε τις ε, λαιλασίες. Πρόκειται λοιπόν για ένα πολύ σημαντικό θέμα. Το θέμα της Ευρωπαϊκής πρέπει να πω ότι είναι ένα θέμα σημαντικό το οποίο απασχολεί τους υπουργούς ήταν το κεντρικό θέμα της συνάντησης της τελευταίας που είχαμε στις Βρυξέλλες και όσον αφορά τα δικαιώματα των εργαζομένων που ανέφερε η κυρία Χόνιμπολ, όντως ο κατακαιρματισμός ή τα διαφορετικά δίκαια ή ο συγκερασμός, η συμβατότητα μεταξύ όλων αυτών των ε, δικαίων είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει. Ξέρουμε ότι τα θέματα της ε, πνευματικής ε, ιδιοκτησίας αυτή τη στιγμή είναι ένα θέμα το οποίο συζητείται και το όλο καθεστώς αναθεωρείται σχέση με το θέμα αυτό σε κάποιες χώρες. Καταλαβαίνω ότι για το Ηνωμένο Βασίλειο το θέμα είναι πρωταρχική σημασία. Εγώ μπόρεσα να συναντηθώ και να συζητήσω διεξοδικότητα με τον ε, Υπουργό Πολιτισμού της Μεγάλης Βρετανίας και να το συζητήσουμε αυτό το θέμα. Είναι λοιπόν σημαντικό αυτό το οποίο αναφέρθηκε για την κατάρτιση των καλλιτεχνών, για την κινητικότητα των καλλιτεχνών και θα ήθελα να σας πω το εξής. Δεν θα πρέπει η ψηφιοποίηση να μας κάνει να ε, σταματήσουμε να βλέπουμε τις άλλες τέχνες τη μουσική, το τσίρκο, όλες τις άλλες, τις καλές τέχνες με τις οποίες πρέπει να ασχοληθούμε. Επαναλαμβάνω λοιπόν τα περιεχόμενα online και η ψηφιοποίηση είναι σημαντικά θέματα, αλλά θα πρέπει να συνεχίσουμε να μελετάμε και όλα τα άλλα θέματα που άφηναν των υπολείπων τεχνών και καλών τεχνών. Δεδομένου ότι είμαστε στην Ευρώπη πάρα πολύ πλούσιοι. Έχουμε αυτούς τους θησαυρού τους πολιτιστικούς, όπως είπε και η Πρόεδρος. Πριν να ολοκληρώσω την παρέμβασή μου, επιτρέψτε μου να κοιτάξω τις σημειώσει μου εντάχει, να δω πως δεν έχω απαντήσει σε κάποιο θέμα. Ένα σημαντικό θέμα, το οποίο ξέρω ότι επίσης απασχολεί, σας απασχολεί όλους σας, είναι τα δύο διαφορετικά δικαιώματα που υπάρχουν και πώς θα μπορέσουμε να τα συγκεράσουμε. Δηλαδή, πρόσβαση σε θέματα πολιτιστικά, πρόσβαση μέσω ίντερνετ, χωρίς να υπάρχουν όλες οι αρνητικές πλευρές. Αυτή τη στιγμή στην Ισπανία η κυβέρνηση μελετά ένα σύνολο κανόνων, ένα πρότυπο, ώστε να υπάρχει συμβατότητα μεταξύ όλων των δικαιωμάτων, σεβασμό των δικαιωμάτων όλων, αλλά χωρίς να χάσουμε τις ε, θετικές δυνατότητες που μας προσφέρει το ίντερνετ, πράγμα που έχει γίνει καθημερινότητα για όλους, να μην οδηγήσουμε και σε ε, παραμερισμό των δικαιωμάτων κάποιων άλλων. Το ίντερνετ, όπως ξέρουμε, είναι για όλους κάτι το οποίο μας Πασχολεί καθημερινά. Σχεδόν όλος ο κόσμος είναι χρήστης πλέον. Και είναι και πολύ σημαντική η παρουσία του για τα θέματα τα πολιτιστικά. Αλλά θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί πάντα. Και βεβαίως θα ήθελα να πω ότι είμαι ανοιχτή σε συνεργαστία κάθε φορά που θέλετε να με συναντήσετε. Είμαι στη διάθεσή σας για να εμβαθύνουμε στα θέματα που μας ενδιαφέρουν από κοινού και είμαι πάντα στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ. Minister. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστώ για τις πολλές απαντήσεις που μας δώσατε. Καμιά φορά είναι δύσκολα τα πράγματα γιατί υπάρχουν επικαλύψεις στους ερωτήσεις. Ίσως θα μπορούσαμε να εδραιώσουμε, να οργανώσουμε καλύτερα την επόμενη φορά, να πούμε σήμερα θα συζητήσουμε αυτό, μετά θα συζητήσουμε και το άλλο. Γιατί καμιά φορά οι ερωτήσει επικαλύπτονται, είναι δύσκολο να λέτε όλα τα ίδια πράγματα. Τι να κάνουμε, έτσι έχουν τα πράγματα, δεν πρόκειται να αλλάξουμε του συναδέλφου. σω και η κυρία Υπουργό ήταν βουλευτή, ξέρει λοιπόν τι γίνεται. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Καλή τύχη, καλή επιτυχία κυρία Υπουργέ. Γιατί χρειάζεται επιτυχία ο πολιτισμός, χρειάζεται δυναμικούς και δεσμευμένους πολιτικούς σε όλα τα επίπεδα. Wir fahren in unserer Tagesordnung fort. Alle, die nicht Συνεχίζουμε την λυσία μα διάταξη. Όποτε δεν θέλουν να συμμετάσχουν, παρακαλώ να βγουν από την αίθουσα. Περνάμε στο σημείο 11 τη ημερησία διάταξη. Speak outside. Huh? I like you all, but uh, please. Wir kommen zum Λέγα ότι περνάμε στο σημείο 11 τη ημερησία διάταξη. Μια στρατηγική Ευρωπαϊκή Ένωση για την Ιωλία. επένδυση και ενδυνάμωση. Ο εισηγητή μας είναι ο συνάδελφος Παπα-Νικολάου και θα του δώσω το λόγο και να παρακαλέσω όσο πιο σύντομα, όσο πιο καλά μπορεί να μας κάνει την εισαγωγή του. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Για να συνδέσω την προηγούμενη συζήτηση που είχαμε και για να εξηγήσω πού ακριβώς βρισκόμαστε σήμερα, εντάχει θα πω τα εξής. Οι πρώτες αναφορές στις συνθήκες μας για τα ζητήματα νεολαίας ξεκινάνε από τη συνθήκη του Μάστριχτ και το πρώτο κείμενο συνολικά που περιγράφει όρους και τρόπους συμμετοχής των νέων και ενδυνάμωση των νέων το έχουμε το 2001 με την Λευκή Βίβλο τότε ε, που ήταν ένα σημαντικό κείμενο ε, της εποχής εκείνης που ακόμη και σήμερα ε, έχουμε αναφορές. Στη συνέχεια ε, δημιουργήθηκε το 2002 ένα πλαίσιο για την συνεργασία στα θέματα νεολαίας, το οποίο ανανεώθηκε το 2005 με το ε, Σύμφωνο για την Νεολαία και ε, φτάνοντας στο τέλος της προηγούμενης περίοδου, για το Σύμφωνο για την Νεολαία είχε έναν ορίζοντα ε, τετραετίας. Σήμερα ερχόμαστε με ένα νέο τίτλο και μια νέα ανακοίνωση της Επιτροπής να συζητήσουμε για τις πολιτικές για την νεολαία για την επόμενη δεκαετία. Εξέδωσε λοιπόν μια ανακοίνωση η Επιτροπή, ακολούθησε με μια νέα ανακοίνωση το Συμβούλιο, ε, πολύ αναλυτικά περιγράφονται μέσα κάποια πεδία ε, στα οποία πρέπει να δραστηριοποιηθούμε προκειμένου να ενισχύσουμε τις πολιτικές μας για τους νέους, προκειμένου να δώσουμε τη δύναμη και την ε, ενδυνάμωση στους νέους ανθρώπους προκειμένου να μπορέσουν οι ίδιοι να σταθούν στα πόδια τους και να προοδεύσουν. Και βεβαίως η Επιτροπή αλλά και το Συμβούλιο προσπαθούν να δώσουν κατευθύνσει πώς μπορούμε να προωθήσουμε ακριβώς αυτές τις επιδιώξει. Ερχόμαστε λοιπόν εμείς σήμερα εδώ και έχετε ένα σχέδιο, ένα draft report ενώπιόν σας προκειμένου να δούμε πώς μπορούμε να συνδράμουμε και να συνεισφέρουμε σε αυτή την προσπάθεια. Ξεκινάω λέγοντας το εξής. Δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι εκείνη που έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει καθοριστικές αποφάσεις για τα θέματα των νέων. Όπως όλοι γνωρίζετε ισχύει η αρχή της επικουρικότητας, ως εκ τούτου η πρωτοβουλία ανήκει στα κράτη-μέλη. Και αυτό ακριβώ καθιστά πιο δύσκολο το ρόλο μα σε σχέση με αυτά που επιδιώκουμε να κάνουμε, σε σχέση με αυτά που θέλουμε και καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να γίνουν. Γιατί στα πλαίσια τη επικουρικότητας αυτό που πρωτίστω πρέπει να κάνουμε είναι να προσπαθούμε να συντονίζουμε δράσει, να λαμβάνουμε πρωτοβουλίες ούτω ώστε τελικά να πείθουμε τα κράτη-μέλη προκειμένου το υλικό που προκύπτει και τα συμπεράσματα που έχουμε από όλη αυτή τη διεργασία να μπορέσουμε εν τέλει να το ε, αξιοποιήσουμε σε εθνικό επίπεδο. Σε όλη την διαδικασία που έχει προηγηθεί και στις συναντήσεις που είχα και σε όλες τις συζητήσεις και με συναδέλφους και με την Κομισιόν και με το Συμβούλιο προσπάθησα ακριβώς να καταλάβω πώς μπορούμε να συνδράμουμε περισσότερο και να καταλήξουμε σε αυτούς τους στόχους. Και σε αυτή τη βάση ε, κατέληξα σε αυτό το σχέδιο που έχετε μπροστά σας και νομίζω ότι τα πιο βασικά σημεία αυτού του σχεδίου είναι ακριβώς τα key Μάρξ, οι βασικές παρατηρήσεις που αφορούν την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής για την νεολαία. Πρέπει να ε, πω σε όλους ότι νομίζω ότι στο επίπεδο της Κομισιόν γίνεται σημαντική δουλειά. Ε, ξεκίνησαν και πλέον ε, πραγματοποιούν και έρευνες σε συγκεκριμένα ε, στοιχεία που αφορούν τους νέους ανθρώπους, στα θέματα ανεργίας, στα θέματα εκπαίδευσης, σε θέματα που αφορούν τη ζωή των νέων ανθρώπων, για αυτούς που φεύγουν από το σχολείο, για, τις, για εθισμούς, για πάρα πολλά πράγματα. Τα είχαμε πει αν θυμάστε και την προηγούμενη φορά. Και το ζητούμενο είναι πώς όλα αυτά μπορούν να είναι χρήσιμα στα κράτη-μέλη και να καταλήξουμε στο να ε, έχουμε πραγματικά αποτελέσματα και να, να προχωρήσουμε κάποια βήματα από τη θεωρητική συζήτηση. Γιατί πράγματι σε επίπεδο θεωρητικό Είμαστε πάρα πολύ καλά και έχουμε πολύ σημαντικά εργαλεία στα χέρια μας, τα οποία όμως πρέπει να αφομοιωθούν από τα κράτη-μέλη. Ακριβώς λοιπόν γι' αυτό καλωσορίζουμε τι πρωτοβουλίε που λαμβάνονται και από την Επιτροπή και από το Συμβούλιο και επαναλαμβάνω επειδή έχουμε επικουρικότητα κάθε τέτοια συζήτηση είναι σημαντική και πολύτιμη για να υπενθυμίζει πάντοτε την αγωνία μα και το ενδιαφέρον του Κοινοβουλίου μα για τους νέους ανθρώπους. Οι νέοι άνθρωποι είναι το μέλλον της Ευρώπης, οι νέοι άνθρωποι σήμερα και μέσα στην παγκόσμια οικονομική κρίση έχουν τα μεγαλύτερα προβλήματα και ω εκ τούτου πρέπει να δίνουμε έμφαση στα προβλήματα αυτά. Επειδή ακριβώς έχουμε την επικουρικότητα, το, η μέθοδος η οποία υιοθετείται προκειμένου να συντονίζονται οι δράσεις και να λαμβάνονται πρωτοβουλίες είναι η ανοιχτή μέθοδος συνεργασίας. Μέσα από την ανάλυση που και εγώ πραγματοποίησα και νομίζω και σε πολλές, σε πολλές άλλες ε, πολιτικές αντίστοιχες έχουμε το ίδιο ε, εργαλείο, διαπίστωσα και εγώ πολλές αδυναμίες σημαντικέ αδυναμίες, οι βασικότερε είναι το έλλειμμα νομιμοποίησης που υπάρχει στη συμμετοχή στην ανοιχτή μέθοδο συντονισμού. Ε, πολλές, δεν συμμετέχουν κοινοβούλια, δεν συμμετέχουν κοινωνικοί φορεί. Συνήθω η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών πραγματοποιείται σε ένα επίπεδο κυρίω δημοσίων λειτουργών και ε, για να γίνω όσο περισσότερο αντιληπτός καταλήγω στο ότι η ανοιχτή μέθοδος συνεργασίας είναι μια ευρεία έννοια συνεργασίας με το συντονισμό κατά κανόνα της Κομισιόν όπου τα κράτη-μέλη προσέρχονται, αναλύουν όσο μπορούν τα δεδομένα που έχουν και με βάση την ανταλλαγή των απόψεων και τα παραδείγματα που υπάρχουν καταλήγουν σε κάποια συμπεράσματα στα οποία ε, βασίζονται για να, για να προάγουμε τις πολιτικές μας. Δυστυχώς όμως στην ανοιχτή μέθοδο συνεργασίας επίσης σε εθνικό επίπεδο δεν έχουμε κάποιους δείκτες κάποια δεδομένα σταθερά, τα οποία θα μπορούσε να αναζητήσει ο καθένα από εμά, προκειμένου να δούμε το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται το κάθε κράτο μέλο. Θα ήθελα πολύ εγώ που βρίσκομαι στην Ελλάδα να ξέρω τι κάνει η Ιταλία ή η Γερμανία για συγκεκριμένα θέματα που αφορούν τους νέους, τι δράσεις υιοθετούν προκειμένου με βάση τους καλούς δείκτες ή τους κακούς να κρίνω και να μπορώ να βγάλω συμπεράσματα. Αυτά δεν υπάρχουν. Όπως επίσης μέσα και αυτά όλα τα γράφουμε, ε, ε, γράφονται στο σχέδιο που έχετε. Όπως επίσης δεν μπορούμε ε, εύκολα να βρούμε δημοσιοποιημένα κάποια πορίσματα από τις συζητήσεις που γίνονται στην ανοιχτή μέθοδο συντονισμού. Πραγματοποιείται δηλαδή ένας διάλογος, ανταλλάσσονται κάποιες απόψεις, τελικά δεν μπορούμε να μάθουμε που, ποια είναι τα συμπεράσματα και ως εκ τούτου και εμείς ως Κοινοβούλιο δεν μπορούμε να βοηθήσουμε περισσότερο και νομίζω πραγματικά ότι ειδικά στα θέματα αυτά, στον καθορισμό κάποιων θεμάτων, στο, στους κύκλους εργασιών που προβλέπει η ανακοίνωση και της Επιτροπής και του Συμβουλίου θα μπορούσε να έχει άποψη το Κοινοβούλιο προκειμένου να μπορούμε και εμεί να συνεισφέρουμε στα, στα μα, μας, σε επίπεδο κοινοβουλίου και όχι μόνο, στα ε, ζητήματα αυτά και να δίνουμε έμφαση στα ζητήματα αυτά. Κάτι το οποίο δυστυχώ δεν σημαίνει όσο θα θέλαμε. Και βεβαίως έχουμε σημαντική αδυναμία, και αυτό το γράφουμε στο σημείο 8, ότι ε, δεν αξιολογούμε τις πολιτικές τις οποίες εφαρμόζουμε. Έχουμε κάποιες εκθέσεις πρόοδου των κρατών μελών, οι οποίες όμως και πάλι δεν δημοσιοποιούνται. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι σε κάποια σημεία τα κράτη-μέλη δεν θέλουν να πούν περισσότερα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει όμως οφείλουμε να προσπαθήσουμε να τους πείσουμε να καταλήγουμε σε κάποιους κοινού όρους ε, σε σχέση με τη δημοσιοποίηση προκειμένου να καταλαβαίνουμε και σε τι επίπεδο βρισκόμαστε. Και βεβαίως φτάνω σε ένα πολύ κέριο ζήτημα που ε, νομίζω ότι το σκέπτεστε όλοι και αφορά τα προγράμματα που ήδη υπάρχουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε σχέση με τους νέους ανθρώπους και όχι μόνο. Γνωρίζετε πολύ καλά όλοι το πρόγραμμα Εράσμους, το Νταβίντσι, το Κομένιους και πολλά άλλα. Όλα αυτά τα, τα προγράμματα δεν αναφέρονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής και του Συμβουλίου. Όπως ενημερώθηκα μάλιστα στην Επιτροπή υπάρχει διαφορετική μονάδα για τα προγράμματα και είναι διαφορετική η μονάδα σε σχέση με τις ε, πολιτικές και τις στρατηγικές που έχουμε για την νεολαία και ενώ τελικά τα μόνα χειροπιαστά εργαλεία, στα οποία δηλαδή συνεισφέρουμε και με όρους οικονομικούς, για να βοηθήσουμε τους νέους ανθρώπους είναι τα προγράμματα και εκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση κάθε χρόνο πληρώνει εκατομμύρια ευρώ, τελικά τα προγράμματα αυτά δεν πηγαίνουν χέρι με χέρι, και αυτό γράφουμε ακριβώς στο σημείο 9, με τις ε, πολιτικές που χαράσουμε προκειμένου να δούμε πώς σε κάθε πεδίο δράσης μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα προγράμματα και πώς αντιστοίχως μπορούμε τα προγράμματα να τα προσαρμόζουμε στις ανάγκες και στις στρατηγικές που έχουμε προκειμένου να καταλήγουμε στα καλύτερα δυνατά χειροπιαστά συμπεράσματα. Κλείνοντας ε, με την ανοιχτή μέθοδο συνεργασίας, βεβαίως ε, είναι επίσης πολύ σημαντικό το γεγονός ότι για τις πολιτικές για την νεολαία πρέπει κάθε φορά να έχουμε διατομεακή προσέγγιση. Αυτό σημαίνει ότι κάθε φορά που συζητάμε για μείζοντα ζητήματα, για το ασφαλιστικό, συζητάγαμε τις προάλλες με την κυρία Κώστα και στο σημείο αυτό θέλω να ευχαριστήσω όλους τους κοιόδης συζητητές, τους συζητητές των άλλων ομάδων ε, για την εξαιρετική συνεργασία που έχουμε μέχρι σήμερα. Ε, συζητάμε για το περιβάλλον, συζητάμε για, για τόσα κρίσιμα ζητήματα. Σε αυτά ακριβώς τα δεδομένα πρέπει να προσαρμόζουμε και τι ανάγκες των νέων που αυτό καλό ή κακό πολλέ φορέ το αφήνουμε σε δεύτερη μοίρα. Και είναι στο χέρι μα ω πολιτικό όργανο κορυφαίο, ε, συλλογικό όργανο, να, επιδιώκουμε να δίνεται έμφαση στα θέματα των νέων. Και, σε... και σε αυτό ακριβώ πρέπει στην ανοιχτή μέθοδο συνεργασία εμεί ω Κοινοβούλιο να έχουμε μεγαλύτερη παρέμβαση. Στη συνέχεια βεβαίω, επειδή στη συνέχεια του σχεδίου που έχετε μπροστά σα, και κλείνω κυρία Πρόεδρε καταρχήν, και αφού επαναλάβω ότι κατά τη γνώμη μου στην παρούσα φάση αυτό που εμείς έχουμε περισσότερο να συνεισφέρουμε ως Κοινοβούλιο είναι ακριβώς να επιδιώξουμε την, ε, την εφαρμογή και την ενσωμάτωση των πολιτικών που προτείνουμε για την νεολαία, το συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών, τη δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων και αφομοίωση των συμπερασμάτων από τα κράτη-μέλη, σας λέγω ότι δεν είναι ε, δεν, δεν, δεν είναι δυνατό και δεν επιτρέπεται και εμεί ως Κοινοβούλιο να μην έχουμε μια ε, τοποθέτηση σύντομη βεβαίω σε ένα πολύ περιορισμένο πλαίσιο αυτού του πρώτου σχεδίου. Υπενθυμίζω ότι μόνο 6.000 χαρακτήρε έχουμε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε. Ε, να μην γίνει μια σύντομη αναφορά στου τομεί δράση. Προσπάθησα λοιπόν με ε, ε, απλέ αναφορέ σε συγκεκριμένα σημεία όμω τα οποία θεωρώ ευαίσθητα να ε, κάνω μια σύντομη ε, τοποθέτηση σε ό,τι αφορά το κοινοβούλιο μας ε, για την εκπαίδευση και την κατάρτιση, για την απασχόληση και το επιχειρηματικό πνεύμα, για την υγεία, την ευζοία και το περιβάλλον. Το περιβάλλον το αναφέρουμε εμείς ως ε, πεδίο δράση δεν αναφέρεται στο, στις, στην ανακοίνωση Επιτροπής και του Συμβουλίου. Θέλω να πω δηλαδή αυτούς τους τίτλους εμείς τους αλλάζουμε προκειμένου ε, κατά τη γνώμη μου να τους προσαρμόσουμε περισσότερο ε, σε αυτά που αντιλαμβανόμαστε ως, ως προτεραιότητες. Καθοριστικό είναι το ζήτημα της συμμετοχής. Στο σημείο αυτό, να σας πω μόνο στο, στην παράγραφο 27, ε, δηλώνουμε ότι λυπούμαστε για το γεγονός ότι πέραν των άλλων δεν έχει προταθεί ε, μια συγκεκριμένη δράση για τη βελτίωση της παρουσίας των προγραμμάτων στους νέους. Έχουμε μια αξιολόγηση των προγραμμάτων στα χέρια μα, η οποία όμω προέρχεται από εκείνου που συμμετέχουν στα προγράμματα. Εγώ θα ήθελα να έχω αξιολόγηση από όλου του νέου σε κάθε κοινωνία, να μάθω αν γνωρίζουν τα προγράμματα οι νέοι άνθρωποι και αν έχουν πρόσβαση σε αυτά, ειδικά σε απομακρυσμένε περιοχέ, στην επαρχία, εκεί που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη τα νέα παιδιά. Δεν το βλέπουμε αυτό. Ε, και βεβαίω, ό,τι αφορά τι εθελοντικέ δραστηριότητε, οφείλουμε να χαιρετήσουμε την απόφαση και είχαμε και έκθεση τις προάλλες για, την, για το Ευρωπαϊκό Έτος του Εθελοντισμού. Στην κοινωνική ένταξη οφείλουμε να κάνουμε αναφορά και βεβαίως στα ζητήματα της νεολαίας και του κόσμου. Κλείνοντα την πρώτη μου εισαγωγή, θέλω να πω ότι η συζήτηση σε σχέση με τα ζητήματα νεολαία είναι μια συζήτηση η οποία θα συνεχίζεται πάντοτε, δεν τελειώνει ποτέ. Οι ανάγκε των νέων ε, πάντα θα είναι υπαρκτές και αυξανόμενες. Είναι καθήκον μας σε κάθε επίπεδο να συνεισφέρουμε όσο το δυνατόν περισσότερα μπορούμε, γιατί ακριβώς το μέλλον της Ευρώπης είναι οι νέοι. Αναφέρω στα, ε, στην εισαγωγή της νεολαίας ότι μέσα από αυτές τις πολιτικές μπορούμε καθοριστικά να συμβάλλουμε και στην ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής συνείδησης για τους νέους ανθρώπους, για τη νέα γενιά της Ευρώπης και ε, ε, κλείνω ακριβώς με αυτό υπάρχουν σημαντικά δεδομένα, έχουμε τη δυνατότητα ως κράτη-μέλη, ως ε, Ευρωπαϊκή Ένωση με την Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο να δρομολογήσουμε δράσεις και να ιεραρχήσουμε τις προτεραιότητες, να μπορέσουμε να, με, με όλες τις δομές που έχουμε να εξηγήσουμε στα κράτη-μέλη πώς θα μπορούσαμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Χρειάζεται όμως προσήλωση και των κρατών μελών, χρειάζεται προσπάθεια όλων μας προκειμένου να δοθεί έμφαση σε αυτή την προσπάθεια και μόνο έτσι θα μπορέσουμε κάποια στιγμή στα πλαίσια της επικουρικότητας να έχουμε την περηφάνεια να ανακοινώνουμε χειροπιαστά αποτελέσματα. Αυτά καταρχήν ελπίζω να μην σας κούρασα κυρία Πρόεδρε. πολύ έντονα και πολύ γλίγορα όλα αυτά Γιώργο. μίλαγε τόσο γλίγορα που μα έβγαλε νοκάουτ λίγο πολύ. Ευχαριστώ πάντω φαίνεται ότι μελέτησε το θέμα εις βάθος. Αρχίσουμε τη συζήτηση τώρα. Ποιο θα ήθελε το λόγο, η κυρία Χίρσου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή και τους κοιόδους εισηγητές για τη συνεργασία είναι ένα θέμα στο οποίο μπορούμε πραγματικά από κοινού να κινηθούμε προς την διακατεύθυνση. Γιατί η πολιτική για την ενολία δυστυχώ και στα κράτη-μέλη δεν έχει την κύρια προτεραιότητα. Το βλέπουμε αυτό συνεχώς. Είναι δύσκολο το θέμα λοιπόν. Αυτό που χαιρετίζω είναι που συμπεριλαμβάνεται για μια φορά το θέμα των δικτών. Θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα αποτελέσματα στα μέτρα που εφαρμόζουμε. Έχω την εντύπωση ότι σε πολλές πόλεις, σε πολλές το, τοπικές αυτοδικείς, σε πολλές χώρες ακολουθείται τώρα πια αυτή η προσέγγιση και νομίζω ότι είναι η σωστή προσέγγιση να έχουμε αυτούς τους δείχτες για να μπορέσουμε να κάνουμε καλύτερη αξιολόγηση και να μπορέσουμε να έχουμε προγράμματα για νεολαία που ταιριάζουν πολύ καλύτερα γιατί δεν υπάρχει η νεολαία δεν υπάρχει ο νέος ή νέα, θα πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα ε, προσαρμογής των προγραμμάτων μας σε κάστοτε ανάγκες. Επίσης, ο τομέας της άτυπης εκπαίδευσης θα πρέπει να τονιστεί περισσότερο, πράγματι. Στον τομέα της ε, πολιτικής για την νεολαία θα μπορέσουμε να έχουμε την καλύτερη επίδραση εάν ασχοληθούμε κυρίως με τη δε δυνατότητα εκπαίδευσης, κατάρτισης των νέων της, του να δώσουμε στους νέους δυνατότητες, να τους κάνουμε να καταλάβουν ότι μπορούν να δράσουν. Αυτό είναι κάτι που θα τους ακολουθήσει σε όλη τους τη ζωή και έτσι θα μπορούμε να έχουμε μια κοινωνία ατόμων που θα προωθεί ακόμα και τη δημοκρατία. Θα ήθελα να αναφέρω ότι στο σημείο 19 στην απασχόληση ίσως τα πράγματα δεν είναι τόσο εις βάθος, αυξανόμενο ρυθμό των νέων που πήθαν από την ενεργεία. Εγώ θεωρώ ότι η ανεργία είναι ένα πιο επίγοντα θέματα που πρέπει να αντιμετωπίσει η Ευρώπη και θα πρέπει να είμαστε πιο έντονοι στη διατύπωσή μας. θα ε, μπορούμε να είμαστε πιο ακριβείς και πιο συγκεκριμένοι στη διατύπωση του θέματος της ανεργίας. Επίσης, στο θέμα της συμμετοχή στα κοινοβούλια νέων είναι κάτι που πραγματικά έχει αποδειχθεί πάρα πολύ καλό σε διάφορα κράτη-μέλη και θα πρέπει να δούμε κατά πόσον εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούμε να προωθήσουμε κάποια σχέδια, κάποια προγράμματα, ούτε ακριβώς να προωθήσουμε κάτι τέτοιο όπως τα κοινοβούλια νέων. Αυτό που μου έλειψε είναι το θέμα της αρκανότητας για τα ΜΜΕ. Ακριβώς παιδιά και νέοι θα πρέπει να γνωρίσουν καλύτερα τους κινδύνους που υπάρχουν. Και πώς μπορούν να προχωρήσουν και αργότερα όταν είναι ενήλικες παραδείγματος κάνει διαβίου, εκμάθηση κλπ. Αυτά έχω να πω. Ε, κατά τα άλλα θα ήθελα πραγματικά να ευχαριστήσω ιδιαίτερα και ξέρω ότι δεν υπήρχε δυνατότητα να υπάρχει μεγαλύτερη ανάπτυξη του θέματος, όπως όλοι να συμπεριληφθούν και θα δω τι θα γίνει με τις τροπολογίες. Ευχαριστώ. Πρώτα, ευχαριστώ κύριε Χίρσα. Νεφιταλόβα. Ďakujem Ja by som sa v prvom rade chcela poďakovať pánovi spravodajcovi, lebo myslela som si, že taký entuziastický človek θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισήγητη. Είχα την εντύπωση ότι εγώ είμαι η μόνη εδώ που εμφορείται από ενθουσιασμό, αλλά από ό,τι φαίνεται υπάρχουν και άλλοι, όπως η κυρία Χίρς. Ε, ίσως ε, δεν θα πρέπει μάλλον να το εκλάβετε αυτό ως κριτική στη δική μας την Επιτροπή και εγώ θα το πω, ε, πρέπει το Κοινοβούλιο γενικότερα να ασχοληθεί περισσότερο με την νεολαία. Όταν ήρθε, ας πούμε, η κυρία Βασιλείου, μόνο μία ερώτηση της έγινε για την νεολαία και αυτή μάλιστα παρέμεινε αναπάντητη. Γι' αυτό λοιπόν όταν θα αναλάβει το, το αξίωμά τη θα πρέπει να τη ασκήσουμε μεγαλύτερη πίεση να ασχοληθεί περισσότερο με το θέμα τη νεολαία η κυρία Βασιλείου. Τώρα, όσον αφορά τον ορισμό τη πολιτική νέων, ποικίλουν οι ορισμοί στα ε, διάφορα κράτη-μέλη, κυρίως αφορά το θέμα του ορίου ηλικία. Υπάρχει λοιπόν το εξής θέμα. Η νεολαία οι νέοι γενικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, έχουν την αίσθηση ότι δεν τους αφορά η πολιτική, δεν βλέπουν να υπάρχει καμία αντίδραση στις δικές τους τις επιθυμίες, κανένας ε, συσχετισμός με μέτρα που λαμβάνονται για αυτούς. Και θέλω να σας πω ότι πρέπει να συνεργαστούμε περισσότερο και με εκπροσώπους νεολαίων, γιατί αυτά είναι θέματα που θέλω να συζητήσω μαζί τους. Όταν, ας πούμε, μιλάμε για την απασχόληση, τότε τι γίνεται. Βλέπουμε εκπροσώπους των οργανισμών απασχόλησης, γίνονται συζητήσεις, αλλά δεν βλέπουμε εκπροσώπους νεολαίας. Εγώ θέλω να το κουβεντιάσω αυτό με νέους. Γι' αυτό λοιπόν, κύριε Σιγητά, σας ερωτώ. Εσείς συζητήσατε με το Φόρουμ Νέων Ευρώπης και με άλλες ε, νεολαίες, άλλους οργανισμούς. Ελπίζω στο μέλλον να συνεργαστούμε σωστά. Τώρα, η επόμενη νεολαία, η κυρία Παλιαδέλη. Ε, μόνο ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δεν έχω καμία σχέση με τους νέους βιολογικοί βεβαίως αλλά τους ξέρω και ως μητέρα και ως ε, διδάσκουσα. Ε, εκτιμώ ότι αυτή η έκθεση, όχι η άποψη του, του πολύ καλού συναδέλφου και συντοπίτη μου, του κυριου Παπα-Νικολάου, ε, αντιμετωπίζει το ζήτημα από έξω, από μια ε, απόσταση μιλώντας λίγο γεροντίστικα θα έλεγα και συμφωνώ απόλυτα με την γειτόνισά μου εδώ ε, για τους νέους χωρίς τους νέους. Ε, νομίζω το μεγάλο πρόβλημα και τη μεγάλη πρόκληση για προκειμένου να λυθούν ζητήματα που αφορούν στους νέους είναι η, ο τρόπος με τον οποίο θα αντιμετωπίσουμε τη συμμετοχή. Οι νέοι αδιαφορούν για τη συμμετοχή, αδιαφορούν για την Ευρώπη, αδιαφορούν για τους θεσμούς της, ε, ίσως γιατί είναι πολύ απογοητευμένοι από τους πολιτικούς και την πολιτική όπως εκφράζεται και στην πράξη αλλά και όπως διαγκώνεται μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εκτιμώ λοιπόν ότι η μεγάλη πρόκληση και δε, ίσως δεν θα έπρεπε να τονιστεί λίγο περισσότερο είναι η ενεργοποίησή τους, η, ε, πώς θα τους πείσουμε, πώς θα τους ανθαρρύνουμε να συμμετέχουν πολιτισμικά ε, σε ομαδικές δράσεις και πώς θα ξανακάνουμε την πολιτική πιο ελκυστική. Να ανατρέψουμε δηλαδή την εικόνα των πολιτικών στα εθνικά κράτη και των πολιτικών ε, the politicians I mean, έτσι, στην Ευρώπη ως ε, ομάδων διαχείρισης οικονομικών άντε και κοινωνικών προβλημάτων χωρίς όμως να πηγαίνουν στην ουσία. Αυτό δεν ξέρω αν μπορεί να περιληφθεί σε μια τέτοια ε, εισήγηση για την ε, αναφορά που ε, για την έκθεση του, της Ευρωπαϊκής, ε, ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά ως ψήφισμα μπορεί τουλάχιστον να αποτελέσει μια αρχή για μια ουσιαστικότερη προσέγγιση των ζητημάτων που αφορούν στη Λεόλαια. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κοιτάξτε, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά το συνάδελφο κύριο Παπανικολάου γιατί πραγματικά, ε, πρέπει να το πω, συμπεριέλαβε όλους μας στην επιθυμία που προκάλεσε σε όλους να έχουμε ένα κείμενο το οποίο όλοι να συμμερίζονται. Όλοι αυτό θέλουμε. Υπάρχει βέβαια ένα θέμα αρχής που δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε και προφανώς ε, αφορά την ανακοίνωση της Κομισιόν. Είμαστε σε ένα φρικτό έτος θα έλεγα, ανορύμπιλης για τους ε, νέους, με την έννοια ότι αυτό αφορά κυρίως όσους ζουν στην Ευρώπη. Έχουμε τα τελευταία στοιχεία που αναφέρουν ότι οι πολιτικές για τους νέους δεν μπορούν πλέον να είναι όπως ήταν παλαιότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή οι πολιτικές συμπληρωματικές, περιθωριακές και ε, με πιο απλά λόγια πολύ περιορισμένες. Πρέπει να ανατρέψουμε τις προοπτικές για το μέλλον. Σήμερα η θέση των νέων στην Ευρώπη σε όλα τα επίπεδα, οριζόντια. Η θέση λοιπόν των νέων είναι μια θέση που οδηγεί στο να πιστεύουμε ότι οι νέοι είναι κατά κύριο λόγο εκείνοι που πληρώνουν την οικονομική κρίση. Φέτος λοιπόν αυτή η χρονιά σε ολόκληρη την Ευρώπη είχαμε μεγάλη ζημιά που προκλήθηκε κυρίως για τους νέους. Εγώ θέλω να σας πω ότι υπάρχει εδώ ένα σημείο ε, και ευχαριστώ που το αναφέρετε, σωστά το αναφέρετε, αλλά θα πρέπει να το τονίσετε περισσότερο. Δηλαδή ότι σε επίπεδο ευρωβαρόμετρου και επίση και όσον αφορά τι εκθέσει που αφορούν αφορούν τους νέους στην Ευρώπη θα πρέπει να αναφέρονται περισσότερο δείκτες σε ευρωπαϊκό επίπεδο να προβάλλουν στοιχεία που σήμερα δεν είναι σαφή. Δηλαδή, το όριο ηλικία. Α πούμε, δεν μπορεί κανεί να συγκρίνει την ε, ανεργία των 15 ετών με των 25 ετών. Κατόπιν το θέμα του φύλου. Ε, επίσης και αυτό να προβληθεί περισσότερο τι δυσκολίες έχουν τα κορίτσια σε σχέση με τα αγόρια, κυρίως όσον αφορά την ένταξή τους στην αγορά Τρίτον, ε, το κατά πόσον ζει κανεί σε αστικό πλαίσιο ή στην επαρχία. Υπάρχουν δηλαδή θέματα, δείκτες που είπα προηγουμένω, που βοηθούν στο να μπορούμε να κάνουμε καλύτερη σύγκριση. Ε, εγώ λοιπόν θα ήθελα να καλέσουμε και τους εθνικούς φορείς για τους νέους, οι εθνικοί οργανισμοί να ασχοληθούν περισσότερο με το θέμα αυτό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο να οργανώσουν συζητήσεις ε, που να αφορούν όμως τα επίκαιρα θέματα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά που είναι απαρχαιωμένα και εξακολουθούν να αναφέρονται σε αυτά. Σήμερα πρέπει να ασχοληθούν με την κοινωνική πρόνοια, την αγορά εργασίας, με τέτοιου είδους θέματα. Είμαι σίγουρη ότι ελέγχθη, αλλά παρόλα αυτά επιτρέψτε μου να πω ότι στο, ε, στο αιτιολογικό, εκεί στην αρχή, θα ήθελα να προβληθεί περισσότερο αυτό που επιθυμεί η Επιτροπή μας, αλλά ακόμα δεν υπάρχει ως πραγματικότητα στην Ευρώπη. Δηλαδή, το ότι οι πολιτικές για τους νέους δεν θα πρέπει να είναι μόνο προγράμματα που να καταρτίζονται και μάλιστα με λιγότερους πόρους από ό,τι στο παρελθόν θα πρέπει να ζητήσουμε 3 δις ευρώ περισσότερα, ε, περισσότερο για προγράμματα όπως είναι το Erasmus Mundus και άλλο. Και πέρα από αυτό να μην ξεχνάμε ότι η πολιτική για τους νέους στην Ευρώπη, αυτό αναφέρεται στο ψήφισμα, αλλά ξέρετε εγώ θέλω να το προβάλλω ακόμα περισσότερα, Η πολιτική λοιπόν για τους νέους στην Ευρώπη θα πρέπει να είναι ένας τρόπος, το εργαλείο που θα μας επιτρέψει να αναθεωρήσουμε τη συνθήκη της Λισαβόνας και τη στρατηγική του 2020. Όπως ακριβώς κάνει η ε, Κομισιόν για την κρίση και για τη στρατηγική της Λισαβόνης. Σας υπενθυμίζω ότι όταν κάναμε μία ακρόαση, ακούσαμε σχετική με το θέμα, ακούστηκε ότι θα πρέπει να αναθεωρηθεί η πολιτική για τους νέους, όχι μόνο όσον αφορά τα προγράμματα, αλλά και όλες οι πολιτικές, όπως είπε και ο κ. Πανικολάου, όλες οι πολιτικές να υιοθετήσουν μία διάσταση που να αφορά τους νέους και να προβλέπουν περισσότερο το θέμα της χρηματοδότησης. Χρηματοδότησης λοιπόν Λοιπόν για τους νέους χρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά προγράμματα και από ε, κονδύλια από τον προπολισμό, γιατί φοβάμαι ότι σε αυτό το θέμα δεν έχει δοθεί ιδέουσα σημασία. Να καταλήξω και να πω, συμφωνώ με πολλά από αυτά που λέει ο κ. παπα πάρα πολλά ε, τα υιοθετώ και εγώ. Είναι σημαντικό να πούμε ότι υπάρχει και ένα νέο στοιχείο σε συνταγματικό επίπεδο. Δηλαδή, το ότι οι νέοι πρέπει να συμμετέχουν στο δημοκρατική ζωή της Ευρώπη. Και αυτό σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει υπάρχει πλέον αδιαφορία στον τρόπο με τον οποίο διαρθρώνεται ο διάλογος. Γιατί αν συγκρίνει κανείς τους πραγματικούς νέους με τις ενώσεις νέων, θα διαπιστώσει ότι δεν υπάρχει δέουσα προσοχή ε, στα κράτη-μέλη, γιατί ο τρόπος με τον οποίο προσπαθούν να προσελκύσουν τους νέους ε, δεν είναι σωστός. Υπάρχει κάποια κριτική που ασκήθηκε και εγώ τη συμμερίζομαι, δηλαδή ότι θα πρέπει στην έκθεση να ε, προβάλλονται περισσότερο ορισμένα στοιχεία. Γιατί βλέπω, ας πούμε, ότι και η Ισπανική Προεδρία ξαναμπαίνει στον διαρθρωτικό διάλογο. Αναθεώρηση, λοιπόν και ευχαριστώ πάρα πολύ που αναφερθήκατε και στο θέμα των νέων τεχνολογιών. Να υπάρξουν νέες μέθοδοι. Ε, peer communication, αν θέλετε, επικοινωνία μέσα από την τεχνολογία, να υπάρχουν φόρουμ online και αυτό για να μπορούν οι νέοι να εκμεταλλευτούν τις ευρωπαϊκές ευκαιρίες. Γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι η Ευρώπη δεν ενδιαφέρει τους νέους. Οι νέοι απλά δεν έχουν την αίσθηση ότι καλούνται να είναι ενεργοί συνομιλητές στην πολιτική. Όχι μόνο στα προγράμματα που καταρτίζονται και είναι σημαντικά για αυτούς. Ένα άλλο που κατά την άποψή μου είναι πολύ σημαντικό είναι να ενισχύσουμε το ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων πέρα από το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις πολιτικές ε, των νέων. Αυτό ε, είναι μια πολιτική που κατά το παρελθόν ε, αφέθηκε στην Επιτροπή, σε κυβερνήσεις, σε κυβερνητικούς φορείς, όμως τα κοινοβούλια, κυρίως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν συμμετείχαν επαρκώς. Και τώρα πλέον με τις συνθήκες της Λισαβόνας προβλέπεται μεγαλύτερο έλεγχος, ε, διαπραγματεύσεις και ούτω καθεξής. Και αυτή η έκθεση για την νεολαία που γίνεται σε κοινοτικό επίπεδο, η τελευταία έγινε το 2009, αυτή η έκθεση είναι πολύ περιγραφική και δεν περιλαμβάνει αναλύσεις, δεν περιλαμβάνει κατευθυντικές για τι πολιτικέ που πρέπει να χαραχθούν. Το λέει βέβαια και ο εισηγητή, αλλά ίσω αυτό θα πρέπει να το προβάλλει περισσότερο. Κάτι άλλο τώρα. Εγώ το θέμα της επικουρικότητας το κατανοώ βεβαίως, ε, δεν υπάρχει διάσταση απόψεων από αυτού, σαφές, ε, και συμφωνώ απόλυτα σε αυτό το θέμα με τον εισηγητή. Όμως στο ψήφισμα ε, θα πρέπει να είμαστε πιο γενικοί στην έκφρασή μας, ε, γιατί μιλάμε γενικά για την επικουρικότητα. Όμως παρόλα αυτά θα μπορούμε να είμαστε λίγο πιο θαραλέοι. Δηλαδή, να ε, πούμε στην Κομισιόν ότι παρότι ορίζονται διάφοροι τομείς, να αρχίσει η Κομισιόν να σκέπτεται κάπως πιο συγκεκριμένα, θα μπορούσε κανείς να κάνει και πειραματισμούς με συνδυασμένες δράσεις. Α Ας πούμε, να φέρω ένα παράδειγμα. Σήμερα έγινε μια ανακοίνωση από τον Επίτροπο, τον Αρμόδιο, για την ασπρή βίβλο σχετικά με την αναθεώρηση της ε, κοινωνικής ασφάλισης και της πρόνοιας. Μέχρι σήμερα η νέα ήταν εκτός. Να πούμε λοιπόν στην Κομισιόν ότι στο πλαίσιο αυτής της λευκής βίβλου των ασφαλιστικών συστημάτων να βάλει και το θέμα της νέας πρόληψης και πρόνοιας και κοινωνικών επιδοδημάτων για τους ε, νέους. Κατόπιν το θέμα ε, της ε, εργασίας και της εκπαίδευσης. Ε, εντάξει, αναφέρεται κάποια ευχή. Όχι, να γίνει πιο συγκεκριμένα πειραματισμός, πιο, πιο έντονος πειραματισμός ε, για απόψεις που είναι ας πούμε το basic income, το βασικό εισόδημα. δηλαδή να παρεμβαίνει κανείς στα εισοδήματα και να δώσει κίνητρα που να αφορούν καθαρά και μόνο τους νέους. Να είμαστε λίγο περισσότερο θαραλέα, αν βέβαια συμφωνείτε κι εσείς. Αλλά εγώ νομίζω ότι είναι σωστό να το κάνουμε αυτό. Ε, βρισκόμαστε, διανύουμε μια κρίση και δεν φτάνει να εκφράζει κανείς μια ευχή. Αποτύχαμε πλήρως αναφορά αφορά τις ευχές. Και ως εκ τούτου το θέμα είναι να δίνουμε πιο ουσιαστικές κατευθυντήριες γραμμές, ε, προγράμματα και πειραματισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα καλεί τα κράτη-μέλη να προχωρήσουν πέρα από την πεπατημένη. Ευχαριστώ πολύ τον κυριο Πανικολάου γιατί πάρα πολλά από αυτά που λέει τα ε, δέχομαι και εγώ, αλλά βεβαίως θα μου επιτρέψετε να επανέλθω αργότερα με πιο συγκεκριμένες προτάσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν είναι μόνο η νεολαία που είναι υπέρ της νεολαίας εδώ λοιπόν από ό,τι βλέπω και κάποιοι συνάδελφοι που είναι κάποιος, κάπως μεγαλύτεροι δεσμεύονται επίσης. Μια Σκουρία. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή μας για το περιεχόμενο της έκθεσής του και για τη δόνηση, το τράνταγμα που προκάλεσε στη συζήτηση. Εγώ θεωρώ ότι ε, όσον αφορά αυτά που λέει θα πρέπει να είναι το σημείο κίνησης για τους νέους. Πρέπει να βάλουμε κάποια τάξη. Τόσο όσον αφορά τις ευρωπαϊκές ε, πολιτικές όπου ο κύριος ε, Παπα-Νικολάου μας παραθέτει προγράμματα τα οποία πολλές φορές επικαλύπτονται και μόνο αυτό αλλά μερικές φορές δεν επικοινωνούν καν μεταξύ τους. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο ε, να ε, επικοινωνήσουμε με τα κράτη-μέλη, να τους ανακοινώσουμε το τι είναι σωστό να γίνει γενικότερα σε επίπεδο πολιτικών για τους νέους. Θέλω λοιπόν να πω ότι όταν έλαβε χώρα η ακρόαση της Επιτρόπου που είναι αρμόδια ε, για μας, τον έφερε αυτό και η προαλήσα, αυτή για τις πολιτικές, για τους νέους, δεν μας έδωσε ιδιαίτερα ακριβείς ε, απαντήσεις ε, πέρα από αυτό το πρόγραμμα για τη νεολαία και σε κάποια άλλα θέματα εντάξει απάντησε. Όμως εγώ πιστεύω ότι βρισκόμαστε μπροστά σε προβλήματα που αφορούν στους νέους και που πραγματικά είναι έκτακτης ανάγκης. Πρέπει λοιπόν να δούμε πώς ακριβώς μπορούμε να ασχοληθούμε με αυτό το παρετηρητήριο όπως αποκαλείται, να ανταλλάσσουμε απόψεις με ανθρώπους που έρχονται από διαφορετικά κράτη-μέλη έτσι ώστε να δοκιμάσουμε, να βοηθήσουμε τα κράτη για, τους, για τις πολιτικές των νέων. Εδώ ε, αναφέρονται κάποιες αναγκαιότητες και κάποια ειδικά προβλήματα. Θέλω όμως να προσθέσω ότι δεν αρκεί αυτό ε, γιατί είναι σαν μια ε, επιδημία που που πλήττει την Ήπειρό μας ε, μια επιδημία που ε, θίγει κυρίως ε, τα νέα κορίτσια. Και ακόμα δεν έχουν βρεθεί οι σωστές απαντήσεις τόσο όσον αφορά την πρόληψη όσο και όσον αφορά την δυνατότητα επίλυσης. Έχω κατά νου την ένταξη των νέων, ας πούμε των εγκλήστων σε φυλακές, των φυλακισμένων. Δεν ξέρω αν υπάρχουν προγράμματα επανένταξής τους. Το 60% των ε, εγκλήστων ε, σε φυλακές ε, θα πρέπει να υπάρχει ένας τρόπος ένταξής τους στο κοινωνικό σύστημα. Δεν πρέπει να το παραμελούμε αυτό. Ε, πολλές φορές έχει κανείς κατά νου ότι υπάρχει μια νεολαία που αποτελείται μόνο από κούκλες και από ε, τα βέλτιστα πρότυπα. Όχι, δεν είναι έτσι ακριβώς. Βεβαίως, μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν κάποιοι που είπε ότι οι νέοι δεν έχουν ε, ανάγκη κριτικής, αλλά έχουν ανάγκη παραδείγματος, προτύπου. Αυτό λοιπόν μπορούμε να το κάνουμε ως κοινοβούλιο και ως άτομα που έχουμε ευθύνη σε πολιτικό-κοινωνικό επίπεδο. Εγώ λοιπόν θεωρώ καταλήγοντας ότι αυτή η έκθεση, την οποία επιμελώς ε, ε, Παρουσίαση ο κ. θα πρέπει να είναι μόνο το σημείο εκκίνησης. Πρέπει να δουλέψουμε πάνω σε αυτό. Η Επιτροπή μας να επανέλθει με τα εργαλεία που εμείς κρίνουμε απαραίτητα. Εχθές, ε, δυστυχώς, δεν είχαμε τον αρμόδιο Ισπανό Υπουργό που ασχολείται με τα θέματα, γιατί αν ήταν εδώ θα μπορούσαμε να έχουμε έτσι μια άμεση συζήτηση με το θέμα αυτό. Εγώ πιστεύω ότι το μέλλον της Ευρώπης περνάει μέσα από τις νέες γενές. Κατόπιν τούτου, πέρα από αυτήν την έκθεση που παρουσίασε ο κύριος θα πρέπει να επανέλθουμε στο όλο θέμα, να προσπαθήσουμε να βάλουμε τάξη στον τομέα που είναι καθοριστική σημασία για το μέλλον. Kolega Boris. Ja również chciałem podziękować koledze za bardzo ambitny i odważny raport. On wskazuje na de facto brak do tej pory jednolitej i skutecznej polityki do spraw młodzieży. ευχαριστήσω τον συνάδελφο. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει συνεκτική πολιτική στην Ευρώπη για την νεολαία. Θα ήθελα να κάνω τα εξή σχόλια. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον εισηγητή και να πω ότι στα πλαίσια της στρατηγικής της Λισαβόνας θα πρέπει να μπορούμε να υπολογίζουμε στην δημιουργικότητα των νέων. Και συγχρόνως θα πρέπει να μπορέσουμε και να τονίσουμε και να προωθήσουμε το πνεύμα επιχειρηματικότητας των νέων. Επίσης, να προωθήσουμε διάφορες πρωτοβουλίες. Θα ήθελα επίσης να αναφέρω τον ρόλο του αθλητισμού για την εκπαίδευση των νέων, καθώς και την συμμετοχή των νέων στα θέματα πολιτιακά, σε θέματα συμμετοχής τους στις εκλογές. Η κυρία Βασιλείου, Επίτροπος, σε συνεργασία με το Συμβούλιο και τα κράτη-μέλη, θα πρέπει κάτι να κάνει. Είπαμε ότι έχουμε επίσης ελλειπή στοιχεία για τους νέους και τα κράτη-μέλη δεν νομίζω ότι έχουν αναλάβει σοβαρές δεσμεύσεις για να βοηθήσουν τους νέους. Πιστεύω ότι η κυρία Βασιλείου θα διαραματίσει σημαντικό ρόλο. Αυτό τουλάχιστον αναμένουμε από την νέα Επίτροπο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι για θέματα παιδείας και κατάρτισης σφαιρικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι η πολιτική για τους νέους, ε, συμφωνώ με τους προελίσσαντες, δεν είναι και πάρα πολύ καλή. Όσον αφορά το θέμα της κατάρτισης και της εκπαίδευσης των νέων για την επαγγελματική και τεχνική κατάρτιση θα πρέπει να εισαγάγουμε και θέματα πολιτιστικά και πολιτιακά, δεδομένου ότι πρέπει να αισθανθούν οι νέοι ότι είναι Ευρωπαίοι πολίτες. Είπαμε ότι η συμπενοχή τους στα πολιτιακά θέματα είναι πολύ περιορισμένη. Τώρα, και πάλι σε θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, όπως λέγεται στο σημείο 17, και αυτό είναι αληθές, θα πρέπει να υπάρξει η πολιτική της δεύτερης ευκαιρίας, και να γίνει κάτι για να καταπολεμήσουμε την εγκατάλειψη τους, ε, της ε, εκπαίδευσης εκ μέρους κάποιων νέων. Το θέμα της εκμάθησης των γλωσσών επίσης είναι σημαντικό. Θα πρέπει να μπορούν οι νέοι να αξιολογούν σωστά και να γνωρίζουν την ε, κουλτούρα των γονιών τους επίσης. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι θετικό για την δική τους ένταξη στις κοινωνίες στις οποίες ζουν. Η κοινωνική ένταξη επίσης είναι σημαντική. Στο σημείο του 93 αναφέρεται ότι είναι αναγκαίο να δημιουργηθούν προβλήματα για κάποιους νέους που είναι περιθωποιημένοι και δεν νομίζω ότι θα πρέπει τέτοιου είδους προγράμματα να αφορούν μόνο τους νόμιμους μετανάστες, διότι η ένδυα είναι κάτι το οποίο χτυπά και τους ε, παράνομους μετανάστες σε μια χώρα και θα πρέπει να τους προωθήσουμε με κάποιες λύσεις ε, για να γίνουν κάποια στιγμή νόμιμοι πολίτες κοινωνίας στην οποία βρίσκονται και να συμπεριλάβουμε και αυτούς τους μετανάστες σε οποιαδήποτε δράση προβλέψουμε. Όσον αφορά το θέμα, λέει στον κόσμο, νομίζω ότι πρέπει να τονιστεί περισσότερο ένα θέμα το οποίο αναφέρεται στο ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση στην Ευρώπη. Υπάρχει μεγάλο υψηλό ποσοστό, ε, υπάρχει υψηλό ποσοστό ανεργίας και θα πρέπει να προωθηθούν ανταλλαγές και αδελφοποιήσεις με χώρες του Νότου, με κοινότητες ε, χωρών του Νότου, ώστε να μπορέσουν οι νέοι αυτοί κατά κάποιο τρόπο να εμπνευστούν από ένα κοινό σχέδιο που θα τους ενώσει. Ευχαριστώ. Λοιπόν, έχουμε μόνο 10 λεπτά στη διασύνη μας. Ο κύριος Φίσας, μετά η Κομισιόν και μετά ο αγαπητέο Γιώργος και μετά λιώνουμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το θέμα της νεολαίας είναι ένα εγκάρσιο θέμα, κοινό σε όλους. Δηλαδή, επηρεάζει όλα τις ε, απόψεις ζωής και όλες τις πολιτικές που μπορούμε να κάνουμε. Πιστεύω ότι αντί να έχουμε, όπως συνήθως, σε γενικές γραμματείες, γενικές ε, ε, τμήματα, αν θέλετε, που να ασχολούνται με τους νέους, σε κάθε τμήμα Υπουργείου, σε κάθε Υπουργείο να έχουμε σε όλα τα τμήματα ένα νέο, ώστε να εξετάζει τι γίνεται για τους νέους κάθε Υπουργείο και κάθε υπεύθυνο για τους υπόλοιπους νέους. Το λέω αυτό από τη δική μου εμπειρία, διότι τελικά μια γενική διεύθυνση ή μια γενική γραμματεία που ασχολείται με τέτοιου είδους θέματα έχει δευτερεύουσες αρμοδιότητες και δεν μπορεί να επηρεάσει τις πολιτικές για τους νέους. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι πρωταρχική σημασία νέοι να μπορέσουν να ενσωματωθούν σε όλα τα υπεύθυνα υπουργεία και στις σχετικές τους επιτροπές που ασχολούνται με τα προβλήματα της γενιάς, της νέας. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λέγομαι Σερογκέτ Κόπρατ. Είμαι από την ε, μονάδα για την ε, Εθνόλια στην Γενική Δευτέρα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τον εισηγητή για την πολύ καλή και οικοδομητική του έκταση. να αναφερθώ στην ανακοίνωση τη ε, Κομισιόν. Στην τελευταία σελίδα λέγεται ότι η Κομισιόν καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αντιδράσει στην ανακοίνωση αυτή και σκοπεύει να κρατήσει ενήμερο το Κοινοβούλιο για την εφαρμογή του. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτό τώρα το πραγματοποιούμε. Δεν υπερβάλλω νομίζω να πω ότι η πολιτική για την νεολαία πέρασε σε μια νέα εποχή. Έχουμε την θέση ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας που αναφέρεται και στην συμμετοχή της νεολαίας. Έχουμε μια νέα κλειστική επιτροπή, ε, νέα θέματα που θα να απασχολήσουν, που θα τονίσουν και το θέμα της νεολαίας και επίσης έχουμε μια νέα κοινοτική στρατηγική και ήταν καλό να σας υπενθυμίσω ότι πέρσι τον Απρίλιο δημοσιεύσαμε μία ανακοίνωση στην οποία βασιστεί η έκθεση αυτή, αλλά τον Νοέμβριο προετοιμάσαμε ένα ψήφισμα του Συμβουλίου όπου τα κράτη-μέλη ε, επικύρωσαν τη χρηματοδότηση της ανακοίνωσή μας. Και η ανακοίνωση αυτή βασίζεται σε 1,5 χρόνο διαβουλεύσεων με ομάδες νεολαίων, με νέους, με εμπειρογνώμονες κλπ. Ήταν πάρα πολύ βάσιμο κείμενο λοιπόν. Το 2010 είναι το έτος εφαρμογής. Και θα ήθελα να σας υπενθυμίσω σε όλους ότι έχουμε ε, μία τρόικα, Ισπανία, Βέλγιο και Ουγγαρία. Η Ισπανία θα διαφερθεί για την ε, ε, κοινωνική ένταξη Οι άλλε χώρε θα ασχοληθούν με διαφορετικού τομεί ε, του ιδίου θέματο όμω και έτσι θα μπορέσει να προχωρήσουμε. Κάθε Προεδρία έχει το δικό τη ειδικό κέντρο βάρου. Αυτό που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα είναι η απασχόληση των νέων. Διάφοροι αναφερθήκαν στο θέμα της ανεργίας των νέων. Σε ορισμένε χώρε είναι 20%, σε ένα μέσο όρο μάλιστα τη Ευρώπη είναι 20% για τους νέους. Αυτό είναι ένα θέμα που θα μας ε, προσφέρει. Η έκθεση Παπα-Νικολάου το μηνίζει την ανάγκη να υπάρχουν σχετικέ πολιτικέ και σα δείχνω ότι εδώ πέρα τελευταία προετοιμάσαμε διάφορε δίκε. Μία νέα έκθεση για του νέου. Η πρώτη πλήρη εικόνα που δημοσιάζει η Κομισιόν για την Ολέα. Εδώ ένα άλλο βιβλίο που σα δείχνει που σας δείχνω και επίσης και η Eurosat προετοίμασε κάποια στατιστικά στοιχεία γι' αυτό. Βλέπετε λοιπόν, έχουμε διάφορα στοιχεία στα χέρια μα και ευχαρίστω να σα τα δώσουμε δείκτες. Αύριο μάλιστα συνεδριάζει μια ομάδα προγραμμών για τους ε, δείκτες αυτούς. Και ε, έχουμε συμφωνήσει ήδη ότι θα πρέπει να υπάρχουν δείκτες και θα εξετάσουμε τους διάφορους δείκτες που υπάρχουν και να δούμε πώς μπορούμε να τους συμπληρώσουμε με νέους ενδεχομένως. Κάποιος αναφέρθηκε στο ευρωβαρόμετρο και στα στοιχεία. Ναι, σκοπεύουμε να έχουμε ένα ευρωβαρόμετρο για την ολέα και το μέλλον της. Έχουμε και άλλα θέματα. Ε, προ, προσεχώς θα για την κοινωνικότητα των νέων εθελοντών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση για τους νέους επιχειρηματίες, μια ομάδα εμπειρογνωμόνων για την παιδεία των νέων και ούτω καθεξής. Και θέλω να αναφέρω ότι χθε μάλιστα είχαμε μια πρώτη συνεδρίαση του ανανεωμένου διορθωμένου διαλόγου με την νεολαία. Είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι. Στο ψήφισμα είχαμε πει ότι θα συγκληθεί από την Επιτροπή. Ναι, έτσι έγινε, αλλά αυτό είναι κάτι στο οποίο συμμετέχουν ενεργά το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας, παραδείγματος χάρη. Και βλέπουμε εδώ ότι οι νέοι είναι εκείνοι που έχουν το τιμόνι στα χέρια τους, αν θέλετε. Μια γενική εικόνα λοιπόν είναι αυτή του τι γίνεται αυτή τη στιγμή για να είσαστε ενήμεροι. Και σαν τελευταίο σχόλιο θα ήθελα να πω ότι εκτιμώ ιδιαίτερα το ότι ο κύριος Παπα-Νικολάου ε, τονίζει το θέμα ότι θα πρέπει να γίνει πιο γνωστό το θέμα αυτό, να υπάρχει μεγαλύτερη κατανόηση και από τους ευρωβουλευτές. Είσαστε εκλεγμένοι από τους ε, ε, εκλογές στις διάφορες χώρες, στις διάφορες περιοχές και αν γίνει πιο κατανοητό το πρόβλημα αυτό της νεολαίας είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας γιατί η πολιτική για τους νέους ξεπερνάει τον παλιό τομέα στον οποίο ασκείτο και βέβαια οι ευρωβουλευτές ε, ε, είναι πάντα καλόδεκτοι να βοηθήσουν στην προώθηση της ε, κοινωνικής διάστασης σε κάθε θέμα μας Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, Γιώργο, πολύ σύντομα, γιατί θα έχουμε τη δυνατότητα να ξανασυζητήσουμε όταν θα κατατεθούν οι τροπολογίες των συναδέλφων. Ο Γιώργος, παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για, τις, ε, για το σχολιασμό και τις παρατηρήσεις τους. Θα πω όσο μπορώ πιο σύντομα ε, ως απάντηση αλλά και ως δεύτερη τοποθέτηση δική μου τα εξή. Εγώ είμαι βέβαιος ότι όλα όσα κουβεντιάσαμε σήμερα εδώ, τα οποία είναι πολύτιμα και χρήσιμα. Ε, αντίστοιχη συζήτηση γίνεται στη διαδικασία της ανοιχτής μεθόδου συντονισμού, όπως περιγράφεται, και αντίστοιχη συζήτηση γίνεται και σε εθνικά κοινοβούλια και σε εθνικούς φορείς, σε υπουργεία, σε γραμματείες για τους νέους. Το πρόβλημα είναι ότι όλα αυτά τα συμπεράσματα δεν φτάνουν σε ένα τελικό στόχο κάθε φορά, σε πράξη, σε λύσεις, και τελικά όλες αυτές οι συζητήσεις παραμένουν θεωρία. Και γι' αυτό επαναλαμβάνω ότι το βασικό αναφέρεται στο πώς θα μπορέσουμε όλα αυτά και πράγματι η Επιτροπή έχει πολλά στοιχεία να μας παράσχει, εγώ πολλά δεν τα γνώριζα και τα είδα, ε, πώς θα μπορέσουμε όλα αυτά να τα αφομοιώσουμε στα κράτη-μέλη και να μπορέσουν να αξιοποιηθούν και να οδηγήσουν σε αποτελέσματα. Σε σχέση με όλα όσα υπόθηκαν, πολύ σύντομα να απαντήσω ότι Πράγματι, κάποια ζητήματα πρέπει να τα προβάλλουμε και πιο έντονα. Σα λέω ξανά όμω ότι ο χώρο είναι περιορισμένο και εγώ προσπάθησα όσο μπορούσα να γράψω τίτλου και ζητήματα τα οποία ούτω ή άλλω αγγίζουν και πρέπει να αναφερθούν σε μια έκθεση με τρόπο αξιόπιστο του Κοινοβουλίου. Και βεβαίω και εγώ είμαι έτοιμο να κάνω πολλέ τροπολογίε για να ήταν ο μόνο τρόπο να, να, να συνεισφέρω περισσότερο σε αυτή την έκθεση γιατί δεν είχα άλλο χώρο. Ε, σε σχέση με εκείνο που αναφέρθηκε από συναδέλφους για επιφανειακή προσέγγιση ή για ε, προσέγγιση που δεν, ανα, που δεν ε, προέρχεται από νέους κλπ. Εγώ θα σας πω ότι βεβαίως και συνάντησα όλες τις νεολαίες, το, το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας, τις νεολαίες όλων των πολιτικών ομάδων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στην χώρα μου συνομίλησα με όλες τις νεολαίες. Να σας πω ότι προέρχομαι και εγώ, υπήρξα επικεφαλής της νεολαίας του κόμματός μου στην Ελλάδα για πολύ καιρό και νομίζω ότι είχα την ε, άριστη και αγαστή συνεργασία τους και μπορέσαμε και ε, ανταλλάξαμε πολύ σημαντικές απόψεις. Ε, Βεβαίω για το θέμα του ορισμού της νεολαία, στο σημείο 3, αν θα δείτε, γράφουμε ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένος ορισμός και πράγματι υπάρχουν διαφοροποιήσει μεταξύ των κροτών μελών και τις σεβόμαστε. Φυσικά έχουμε οικονομική κρίση. Φυσικά η ανεργία είναι το κυρίαρχο θέμα. Φυσικά την εκπαίδευση πρέπει να τονίσουμε. Επαναλαμβάνω όμως ότι αυτά, αν αρχίσουμε να τα καταγράφουμε, θέλουμε τόμου δεν αρκεί ούτε ένα βιβλίο. Έχουμε ήδη πολύ υλικό και από την Επιτροπή και πολλοί άλλοι έχουν συγγράψει και με στοιχεία θέσεις για τους νέους. Το ζήτημα είναι πώς θα μπορέσουμε, επαναλαμβάνω, να καταλήγουμε σε πρακτικά συμπεράσματα. Και κλείνοντας, επειδή η κυρία Πρόεδρος θα με μαλώσει, ε, θέλω να πω το εξή. Είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε πολύ σημαντικές τροπολογίες και είναι ε, μεγάλη χαρά να βλέπω ότι έχουμε αυτό το ενδιαφέρον. Ε, εγώ ήδη έχω παρακαλέσει, κυρία Πρόεδρε, και τον κύριο, στον κύριο Σκουρία το έχω πει στο συντονιστή μας, αν μπορούμε να το ε, θέσουμε αυτό και ως θέμα στην Ολομέλεια, όταν θα ψηφιστεί για να υπάρξει μια νέα συζήτηση και να δώσουμε έμφαση στην αγωνία μας για τους νέους ανθρώπους. Επαναλαμβάνω όμως κάτι δεν μπορούμε να εξαντλήσουμε περιπτωσιολογικά όλα τα θέματα που αφορούν τους νέους σε μια τέτοια έκθεση. Η μεγαλύτερη συνεισφορά αυτού του Κοινοβουλίου και αυτής της απόφασης αυτή τη χρονική στιγμή θα είναι να κατορθώσουμε όσο μπορούμε να προωθήσουμε το συντονισμό και την ενσωμάτωση αυτών των πολιτικών με τους τρόπους που περιγράψαμε και στην αρχή. Σας ευχαριστώ πολύ προς το παρόν. Μην με χτυπήσετε με το σφύρι κυρία Πρόεδρε. Κοιτάξτε, οι διερμηνείς εργάζονται μέχρι τις 6.30. Δύο λεπτά, λέει η πρόεδρο, θα του εκμεταλλευτούμε παραπάνω. Θα υπογραμμίσω κάτι που είπε ο Γιώργο. Η έκθεση αυτή είναι απάντηση σε μια ανακοίνωση τη Κομισιόν. Βασικά, δεν, θα, δεν δικαιούμεθα να πούμε τίποτα. Μπορούμε να λάβουμε γνώση, να γκρινιάξουμε, να πούμε ό,τι θέλουμε, αλλά αυτό το θέμα υπάγεται στην ε, επικουρικότητα. Αυτό λοιπόν που πρέπει να κάνουμε είναι να καλέσουμε τα εθνικά μα κοινοβούλια να δραστηριοποιηθούν. Αυτό είναι ε, καθήκον που πρέπει να το αλάβει γίνεται στις χώρες σας. Και μετά, από το 2011, ε, θα υπάρχει συζήτηση για το πρόγραμμα νεολαίας. Εκεί λοιπόν μπορούμε να εκφράσουμε τις δικές μας τις ε, ιδέες, τις οποίες ε, θα έχουμε αποκομίσει μέσα από έρευνες τα επόμενα τρία χρόνια. Έχουμε άπλετο χρόνο για να υλοποιήσουμε αυτά που θέλετε. Τροπολογίες μέχρι τις 8 Φεβρουαρίου, Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου, 12 η ώρα και αυτές θα συζητηθούν στις 23 Φεβρουαρίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον εισηγητή, τους συναδέλφους που συμμετείχαν. Ήταν μια πολύ ζωντανή, νεολαίστικη συζήτηση, σημείο 12 της ημερήσιας διάταξης, εχθές το βράδυ ή σήμερα το πρωί. Είχατε όλοι σας την ευχαρίστηση να δείτε και να διαβάσετε τα αποτελέσματα των συντονιστών. Φαντάζομαι συμφωνείτε. Συμφωνείτε πολύ ωραία. Το γράφουμε στα πρακτικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τη Γερμανία, Γεια.